Good morning, ladies and gentlemen. Καλημέρα κυρίες και κύριοι, παρακαλώ καθίστε. Και ας ξεκινήσουμε τη συνεδρία της Επιτροπής Ρέτζη. Έχουμε κάποια μέλη της Επιτροπής μας, αρκετά μέλη για να ξεκινήσουμε τις εργασίες μας. Λοιπόν, ξεκινάμε τη συνεδρίαση. Έγκριση της ημερήσιας διατάξης. Εγκρίνεται η σημερινή διάταξη. Κύριε Βανίστελροι, έχω τρία σχόλια. Πρώτα απ' όλα, σημείο 5 ασαφές για την ομάδα μου μάλλον. Κάποιος που είναι από την περιφέρεια, τελάσια περιφέρεια, τι, τι είναι αυτό, ποιος έρχεται μάλλον, ποιος θα έρθει, κάποιες πληροφορίες, μας δίνετε κάποιες πληροφορίες. Δεύτερον, έχουμε τον Επίτροπο σήμερα, ε, Είχαμε κάποια μέλη που έχουν ερωτήσεις, ε, έχουν προτεραιότητα αν είναι παρόντα. Για το σημείο 13 μετά, είναι το τρίτο σημείο μου. Μπορούμε να το συνδυάσουμε με κάποιες, κάποια σημεία περισυνοχής. τα σημεία για, την ε, συμμετοχή, για το θέμα του, ε, του Συμβουλίου, της απόψης του Συμβουλίου, κυρίως για αυτό το σημείο το 13. Πρώτα απ' όλα απάντηση για το σημείο 5 της ημερήσιας ε, διάταξης. Συζητήσαμε με τη διάσκεψη των περιφερειών των θασίων περιοχών της Ευρώπης εδώ και μήνες. Προσπαθήσαμε να συμπεριλάβουμε την συμμετοχή τους στην ημερήσια διάταξη, να παρουσιάσουν τις δραστηριότητές τους, αλλά ήταν αδύνατον Είχαν ανηλυμένε υποχρεώσει, είχαμε εμεί προβλήματα με την ημερήσια διάταξη, οπότε εμφανίζεται το σημείο αυτό στη σημερινή ημερήσια διάταξη. Ήταν επιθυμία μου αυτή, εν μέρη, να καλέσω κάποιους οργανισμούς όπως αυτόν τον φορέα να παρουσιάσουν την ε, άποψή του, άποψή τους μάλλον, συγγνώμη, και είναι προσπάθεια που καταβάλουμε όλοι μαζί να γίνει, να δώσουμε χρώμα στις εργασίες της Επιτροπής και γι' αυτό εμφανίζονται εδώ στην ημερήσια διάταξη σήμερα. Θα έρθουν αργότερα. Εντάξει, εγώ θετικό. είμαι. Φτάνει να ξέρουμε ποιο θα είναι το θέμα θα καλύψουν για να μπορέσουν να ετοιμαστούμε θεματική προσέγγιση, τον οργανισμό του, θα δούμε, θα δούμε, λέει και η θα δούμε, θα δούμε και έχουμε τη δυνατότητα να το συναντήσουμε ξανά οποιαδήποτε χρονική στιγμή, αν έχουμε και άλλες ερωτήσεις. Μπορούμε να τους ξανακαλέσουμε. Τώρα, όσον αφορά την ερώτησή σας που αφορά το σημείο 13, Επίτροπος. Λοιπόν, Επίτροπος Κρέτσο θα έρθει στις 3 το απόγευμα και θα ξεκινήσει η συνεδρίασή μας το απόγευμα με ανταλλαγή με την κυρία Επίτροπο. Αυτό που αναφέρεται στην ημερήσια διάταξη είναι ανταλλαγή απόψεων, αλλά όσοι ήθιστε θα τις δώσουμε το λόγο για 10-15 λεπτά να παρουσιάσει τη θέση της, να δώσει πληροφορίες για, την άτυπη, για το άτυπο Συμβούλιο Υπουργών, να μας ενημερώσει ποια είναι η κατάσταση στην DG Regio, ότι γίνεται με τα επιχειρησιακά προγράμματα, σε ποια φάση βρίσκονται και μετά από αυτό θα έχουμε τη δυνατότητα να θέσουμε τις ερωτήσεις μας και να λάβουμε απαντήσεις. Αυτό περιμένουμε. Την περασμένη φορά πρέπει να αποχωρήσουμε πολύ γρήγορα. Μάλλον έφυγε πιο γρήγορα η Επίτροπο και ήταν μέλη παρόντα και δεν έφεσαν ερωτήσει. Αν είναι παρόντα τα μέλη, μπορεί να τι ερωτήσει πρώτα. Απάντηση. Α ακούσουμε την Επίτροπο. σω να έχετε και άλλε ερωτήσει μετά από αυτά που θα πει. Ελπίζω τα μέλη που είχαν τι ερωτήσει Ελπίζω αυτοί που ήθελαν να, τα μέλη που ήθελαν να υποβάλουν ότι στην περασμένη φορά να μην απογοητευτούν εκ νέου, λέει ο κ. Βανίστελρο. Εντάξει, λέει πρόεδρο. Λοιπόν, θα ζητήσω να πάρουν το λόγο εκείνοι που έχουν υποβάλουν ε, τι ερωτήσει εδώ και μήνε. Αν έχουν και άλλε νέε ερωτήσει όμω τα μέλη, και αυτό είναι εντάξει. Τώρα για το σημείο 13, σωστά τα λέτε το δεύτερο τμήμα, το δεύτερο έγγραφο μάλλον. Είναι αυτό που παρουσιάστηκε στην άτυπη διπουργική διάσκεψη περί αποτελεσματικότητας και προστιθέμενης αξίας της πολιτικής συνοχής. Αυτό το έγγραφο, από ό,τι θυμάμαι, το αναφέρατε εσείς, ε? ζητήσατε να συμπεριληφθούν τα σχόλια εδώ στην Επιτροπή μας, την Επιτροπή Ρέτζη. Το έγγραφο έχει διανεμηθεί σε όλα τα μέλη νομίζω ήδη. Έχουμε ενημερωθεί δεόντως και θα ακούσουμε την παρουσίαση της Επιτροπής που θα είναι πάρα πολύ σύντομη και θα έχουμε τη δυνατότητα να ανταλλάξουμε κάποιες απόψεις. Γι' αυτό εμφανίζεται το θέμα και συνδυάζονται τα δύο έγγραφα εργασίας σε ένα σημείο. Αυτά λοιπόν για την ημερήσια διάταξη. Υπάρχουν άλλες ερωτήσεις, ε, προτάσεις. Άρα εγκρίνεται η ημερήσια διάταξη. Επόμενο σημείο. Έγκριση των πρακτικών. Από τις 4 και 5 Μαΐου του 2015 το σχέδιο των πρακτικών είναι στα έγγραφά σας. Όσοι ήθιστε, αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις που θα προβληθούν, κατά τη διάρκεια της παρούσης συνεδριάσεως θεωρούνται ως συγκεκριμένα τα πρακτικά. Δεν υπάρχουν προτάσεις, δεν υπάρχουν σχόλια. Τρίτο παραδοσιακό σημείο. Ανακοινώσεις Προέδρου. Έχω δύο. Μία τεχνικής φύσεως, πρώτα απ' όλα. Θυμηθείτε τις κάρτες ψηφοφορίας για το απόγευμα παρακαλώ. Τις κάρτες σας. Έχουμε τρεις ψηφοφορίες. Και θα χρειαστούμε κάρτες για ηλεκτρονική ψηφοφορία σε κάποιες περιπτώσεις. Στην ψηφοφορία. Αυτή ήταν η πρώτη μου ανακοίνωση, τεχνικής φύσεως. Δεύτερη ανακοίνωση. Άτυπη Διπουργική Σύνοδος στη Ρήγα. 9 και 10 Ιουνίου. δύο συναντήσεις. Παρέστην σε δύο συνεδριάσεις. Στη δεύτερη ήμουν με τον κύριο Γκοτσολίνο και τον κύριο Βανίστελ Ρόι. Η πρώτη συνεδρίαση εστιάστηκε επί της νέας πολιτικής ε, συνοχής. Έγινε ανταλλαγή απόψεων μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Προεδρίας και κρατών μελών. Περί των νέων σημείων της πολιτικής συνοχής και πώς γίνονται αποδεκτά από τα κράτη-μέλη, πώς εφαρμόζονται και αν θεωρούν ότι η αιρεσιμότητα εκ των προτέρων, τα δημοσιονομικά, τα χρηματοστικά εργαλεία και η απλούστευση, αυτά τα σημεία, πώς εφαρμόζονται σε κάθε κράτος μέλος συμβάλαμε και εμείς στις συζητήσεις. Δώσαμε μια επισκόπηση για τα νέα στοιχεία της πολιτικής συνοχής. Έγινε αποδεκτή θέση μας στα κράτη-μέλη. Βασικό σημείο ενδιαφέροντος για όλα τα κράτη-μέλη είναι η απλούστευση. Έχουμε πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα δημιουργηθεί μια ομάδα εργασίας υψηλού επίπεδου που θα ασχοληθεί με την απλούστευση της πολιτικής συνοχής. Όλα τα κράτη-μέλη υποστήριξαν την αλόγω ιδέα, παρόλο που δεν είναι ε, πλήρως σαφές το πώς θα οργανωθεί το όλο θέμα. Εν πάση περιπτώσει, στηρίζουν τα κράτη-μέλη την πρόταση, υπήρξαν σχόλια περί των χρηματοστικών μέσων και των δυνατοτήτων που παρέχουν αυτά στα κράτη-μέλη για να αυξηθούν οι ευκαιρίες που παρέχει η πολιτική συνοχής. Και κάποια σχόλια ακούστηκαν για την εκ των προτέρων ερεσιμότητα. Προς έκπληξή μου δεν υπήρξαν πολλά σχόλια περί του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Δεν ήταν ξεκάθαρα τα πράγματα για κανέναν. Τη δεύτερη μέρα την αφοσιώσαμε στο θεματολόγιο για τα αστικά ζητήματα και νέα ομάδα των Υπουργών συμμετείχε στη συνεδρίαση. Βλέπετε σε κάποια κράτη-μέλη υπάρχουν διαφορετικοί υπουργοί. Ένας υπεύθυνο στην πολιτική συνοχής και άλλος υπουργό είναι υπεύθυνο για το αστικό θεματολόγιο και την αστική ανάπτυξη. Τα κράτη-μέλη στο σύνολό τους υποστήριξαν την δήλωση που προετοίμασε η ε, Προεδρία Οπότε έχουμε τη διακήρυξη μάλλον της Ρήγας όσον αφορά το αστικό θεματολόγιο. Έχει διανεμηθεί από τη γραμματεία, αν δεν κάνω λάθος, έτσι. Μάλιστα. Και έχουμε αυτή την διακήρυξη. Αυτή αποτελεί τη βάση για συνεχή εργασία που θα αναλυφθεί από τις επόμενες προεδρίες την Προεδρία του Λουξεμβούργου που θα συνεχίσει να επεξεργάζεται τα θέματα του αστικού θεματολογίου και η Ολλανδική θα ολοκληρώσει το έργο αυτό παρουσιάζοντας τη διακήρυξη του Αμστερλοδάμου για το θεματολόγιο το αστικό. Αυτό λοιπόν είναι το θεματολόγιο το αστικό. Οι Προεδρίες, οι δύο, παρουσίασαν τα σχέδιά τους για την πολιτική συνοχής και το αστικό θεματολόγιο. Είναι σαφές ότι το αστικό θεματολόγιο θα αποτελέσει το βασικό τμήμα των δραστηριοτήτων των δύο προεδριών της Προεδρίας του Λουξεμβούργου και της Ολλανδίας. Το νέο σημείο των συζητήσεων μας αφορούσε το ρόλο των μικρομεσαίων αστικών περιοχών έχουμε αυτό το παράρτημα της διακηρύξεως που ετοιμάστηκε από την ε, Προεδρία της Λετωνίας που έγινε ε, αποδεκτό το κείμενο και υποστηρίχθηκε από τα κράτη-μέλη και από τους ε, εκπροσώπους του Λουξεμβουργού και της Ολλανδίας των δύο επομένων προεδριών έγινε αποδεκτό. Ο ρόλος των μικρών και μεσαίων αστικών περιοχών είναι σημαντικός είναι σημαντικό θέμα, συμφώνησαν όλοι οι Υπουργοί από αυτού. Είναι ζήτημα σημαντικό για την αστική πολιτική να δημιουργηθούν διασυνδέσεις μεταξύ της ανάπτυξης των μεγάλων αστικών κέντρων και των μικρών και μεσαίων αστικών περιοχών. Αυτό είναι το μήνυμα αναμένονται μελλοντικές εξελίξεις βάσει τη διακηρύξεως και βάσει των δραστηριοτήτων ε, των Προεδριών όσον αφορά το αστικό θεματολόγιο. Είχαμε συνεισφορά της Επιτροπής Ρέτζη, έκανα εγώ μια παρουσίαση για το έργο μας όσον αφορά το αστικό θεματολόγιο, την έκθεσή μας και την θέση των μελών της Επιτροπής Ρέτζη. Συνοψίζοντας, το θέμα είναι σημαντικότατο για μας Εξετάζουμε τις μελλοντικέ εξελίξεις στον τομέα, στηρίζουμε τις προσπάθειες των Προεδριών, στηρίζουμε ένθερμα τις προσπάθειες συνδυασμού όλων των εφισταμένων δραστηριοτήτων και εκθέσεων, να μην δημιουργηθούν νέε δικήσεις, νέε μονάδες, νέα έγγραφα, να είμαστε πιο ολιστικοί στην προσέγγιση, να χρησιμοποιήσουμε τα εφιστάμενα μέσα και έγινε άριστα αποδεκτή θέση μας από τα μέλη του Συμβουλίου. Ο κύριος Βανίσταλ Ρόι πήρε το λόγο κατά τη διάρκεια των ε, συζητήσεων. Αν θέλετε μπορεί να μας δώσει κάποιες ε, σχετικές πληροφορίες, αλλά πρόκειται περί της τύπου ε, συνεδριάσεως των Υπουργών υπευθύνων για τη συνοχή και το αστικό θεματολόγιο στην Ρήγα. Θέλετε να πείτε κάτι κύριε Βάνιστον. Ναι, νομίζω ότι υπήρξατε ακριβέστατοι στην παρουσίαση των συζητήσω. Υπάρχουν αυτά, αναφέρονται και σε, στα έγγραφα. Κάναμε μεγάλο βήμα στην Επιτροπή μέσω της εκθέσεώς μας, μέσω της διακηρύξεως της Ρήγας και με το θεματολόγιο ε, προς τα αποτελέσματα του Άμστερνταμ που νομίζω αυτό θα διεξαχθεί τέλος του Μαΐου του 2016. Έχουμε ένα πρόγραμμα, ένα θεματολόγιο. Ήταν υπέροχη η συμμετοχή μας που μπορέσαμε να συμμετάσχουμε παρόλο που επισκιαζόταν από την Ολομέλεια με τιμώρησαν στην ομάδα μου ότι δεν παρέστην σε μια ψηφοφορία. Ε, είναι πάντα δύσκολο να πηγαίνει κανείς σε αυτές τις εκδηλώσεις όταν ταυτόχρονα διεξάγεται η ολομέλεια του Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ όμως για την ενημέρωση και θα δούμε τελικά τι θα απορρεύσει από όλα αυτά. Ευχαριστώ λέει Πρόεδρος, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω να συνεχίσουμε με τη δημιουργική μας αυτή παράδοση, που να συμμετέχουμε στις συνεδριάσεις των Υπουργών, ακόμα και στις άτυπες, αλλά είναι σημαντικό να είμαστε στην πρώτη γραμμή, να ελέγχουμε τη θέση μας, να κατανοούμε και πώς βλέπει τα πράγματα η άλλη πλευρά, δηλαδή το Συμβούλιο. Αυτά λοιπόν όσον αφορά τις ανακοινώσεις, δεν έχω άλλες ανακοινώσεις, το επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης, στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ενώσεως για την Αδριατική και την, το Ιόνιο μετά από αίτημα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Ιουνίου του 2014, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνέταξε ανακοίνωση περί της Ευρωπαϊκής Ενώσεως για την Αδριατική και το Ιόνιο. Συνοδευόταν από σχέδιο δράσης αυτή η πρόταση. Είναι η τρίτη μακροπεριφερειακή στρατηγική και καλύπτει οκτώ χώρες. Οι μισές από αυτές είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, όπως η Κροατία, η Ελλάδα, η Ιταλία και η Σλοβενία. Και τα άλλα μισά κράτη είναι χώρες που είναι υποψήφιες χώρες Αλβανία, Μαυροβούνιο και Σερβία. Υποψ... Και η Βοσνία Ζεγοβίνη ενδεχομένω μπορεί να αποκτήσει θέση υποψηφίας χώρας. Θα υφετηθεί τέταρτη μακροπεριφερειακή ε, στρατηγική για την περιοχή των Άλπαιων, ανακοίνωσε Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτό το μήνα. Είναι στο πρόγραμμα, οπότε θα έχουμε νέα μακροπεριφερειακή στρατηγική Γενικό στόχο τη στρατηγικής για την Αδριατική και το Ιόνιο είναι η πρόθεση βιώσιμη οικονομική και κοινωνική ευημερία στην περιοχή μέσω αναπτύξεω και δημιουργίας θέσεων απασχόληση, διατηρώντας δε το περιβάλλον. Η, συνο... πολιτική συνοχή τη Ευρωπαϊκή Ένωση θα δραματίσει σημαντικό ρόλο όσον αφορά την υλοποίηση τη εν λόγω στρατηγικής. Στη συνεδρίαση τη Επιτροπή Ρέτζη τον Μάιο, ο εισηγητή μας, ο κύριος Γιάκοφτσιτς, περιέγραψε τι αρχικέ αμφιβολίε του σήμερα παρουσιάζει το σχέδιο εκθέσεώς του. Προτείνω προθεσμία για αποβολή τροπολογιών 12 το μεσημέρι της Παρασκευής 3 Ιουλίου. Παρασκευή 3 Ιουλίου, 12 το μεσημέρι. Θα ψηφίσουμε στη συνεδρίασή μας τις 17 Σεπτεμβρίου. Ε, θα ψηφίσουμε την τελική έκθεση. Αυτές είναι οργανωτικές λεπτομέρειες και θα δώσω το λόγο στον κύριο Γιάκοφ για να παρουσιάσει την έκθεσή του. Και έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Όσον αφορά το θέμα αυτό, πρέπει να πω καταρχάς ότι εύχομαι καλημέρα σε όλους και ευχαριστώ όλους σας για την συνεργασία των τελευταίων μηνών μετά την Ιταλική Προεδρία που ξεκίνησε η εφαρμογή, ε, η δρομολόγηση της Αττικής για το Ιόνιο και την Αδριατική δεν ε, θέμα ευγενία αυτά που λέω. Νομίζω ότι συνεργαστήκαμε πολύ φιλικά, πολύ επικοδομητικά. Ήταν πολύ καλή η ατμόσφαιρα και ευχαριστώ όλος την κυρία Τόμασιτς και τους άλλους συναδέλφους και όπως τον κύριο Φραντς Μπόγκοβιτς που δυστυχώς δεν είναι εδώ σήμερα που συνεργάστηκαν μαζί μου και που υπήρξαν συνεισηγητές για την ε, εν λόγω στρατηγική Ξεκινήσαμε λοιπόν καλά τις εργασίες μας. Τώρα έχουμε ένα έγγραφο στα χέρια μας, το οποίο πρέπει βέβαια να συζητηθεί περαιτέρω. Πιστεύω όμως ότι στο τέλος θα έχουμε ένα καλό έγγραφο και όλοι μας μπορούμε να υποβάλουμε τροπολογίες όσον αφορά το έγγραφο. Η έκθεση αυτή ε, έφτασε ένα σύνολο 6.000 λέξεων και γνωρίζουμε πόσο σημαντικός είναι ο τομέας αυτός για την Ευρώπη και η περιοχή για την Ευρώπη. Ε, θα προσθέσουμε λοιπόν κάποια στοιχεία μέσω των τροπολογιών. Όπως είπε και η Πρόεδρος, η προθεσμία είναι 3 Ιουλίου για τις τροπολογίες. Κυρίες και κύριοι, η έκθεση αυτή είναι περιπλοκότατη, διότι έχουμε τρία κράτη-μέλη της τέσσερα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως που καλύπτονται και τέσσερα κράτη που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, που είναι υποψήφιες. Αυτή η στρατηγική καλύπτει χώρες από μια περιοχή που πριν από 20 χρόνια είχαν και πόλεμο η πολιτική κατάσταση, η οικονομική κατάσταση, η κοινωνική κατάσταση ε, αντιμετωπίζουν προβλήματα. Τα προβλήματα είναι αποτέλεσμα της καταστάσεως που προανέφερα. Έχει όμως, υπάρχουν γειτονικέ χώρες που είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ενώσης, Κροατία, Σλοβενία, η Ελλάδα και η Ιταλία. Χώρες που πάντα συμμετείχαν πολύ στις όλες εξελίξεις της περιοχής Υπάρχει λοιπόν ένα πολιτικό φρέμιο και αυτό, ε, πλαίσιο συγγνώμη, και το πλαίσιο αυτό μπορεί να δώσει στην περιοχή μια οικονομική όθηση και αυτό μέσω διαφόρων μηχανισμών που ήδη υφίστανται εν μέρη. Γι' αυτό χωρίσαμε την έκθεση όπως προτάθηκε και στην αρχή σε τέσσερα κεφάλαια. Έχουμε τη γαλάζια ανάπτυξη, τις διασυνδέσεις της περιοχής, την ποιότητα του περιβάλλοντος με το τρίτο κεφάλαιο και βιώσιμο και ανταγωνιστικό τουρισμό. Ε, βέβαια, αυτά τα στοιχεία ε, είναι τα παρόντα, κάποια από αυτά είναι καινούργια και δεν συνδέονται άμεσα με αυτά που είχε προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά, αλλά τα στοιχεία αυτά και τα σημεία αυτά είναι κοντά στις αρχικές προτάσεις όλα αυτά τα στοιχεία ίσως να παράγουν και συνέργειες και πιστεύω ότι μέσω των τροπολογιών μας θα μπορέσουμε να ενισχύσουμε την έκθεση και ότι θα μπορέσουμε να πετύχουμε στο τέλος μια συνένεση όσον αφορά την έκθεση. Επιτρέψτε μου να υπογράψω δύο πολύ κρίσιμα στοιχεία. Δεν θέλω να διαβάσω το κείμενο που συνέταξα, αλλά θέλω να πω το εξή. Αν θέλουμε πραγματικά να βοηθήσουμε χώρες που δεν είναι ακόμα μέλη της Ευρωπαϊκής Ενώσεω και που έχουν όμως σχέσεις μαζί μας, η Παγκόσμια Τράπεζα και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα συγγνώμη, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων παρέχουν δανειοδοτήσεις και πόρους το Μαυροβούνιο, παραδείγματος χάρη, θέλει να εξαγάγει ενέργεια μέσω υποθαλασσίων καλωδίων. Αξιέπαινη πρόταση, αξιέπαινο έργο αυτό. Μια άλλη λεπτομέρεια που θα ήθελα να υπογραμμίσω. Πιστεύω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να συμμετάσχει και να εμπλακεί στους διοικητικούς φορείς που θα υλοποιούν τη στρατηγική το Ευρωκοινοβούλιο δεν εμπλέκεται ακόμα. Είναι έτοιμά μας αυτό να μπορέσουμε να εμπλακούμε και να συμμετάσχουμε. Αυτό είναι δικαιολογημένο και πρέπει να επιμείνουμε να συμμετέχει το Ευρωκοινοβούλιο στους διοικητικούς φορείς που θα ε, τα προγράμματα. Γαλάζια ανάπτυξη λοιπόν. Η γαλάζια ανάπτυξη είναι ένα από τα κεφάλαια της ε, εκθέσεως. αναφισβήτητα η, Αδριατική, η ακτή της Αδριατικής και του, η ακτή του Ιουνίου είναι περιοχές πολύ πλούσιες σε πόρους, φυσικούς πόρους και ανθρώπινους ε, πόρους. Έτσι αυτή η περιοχή γίνεται μια περιοχή από τις ομορφότερες στην Ευρώπη και στον κόσμο θα έλεγα. Επιτρέψτε μου να εκφράσω όμως και κάποια ανησυχία που έχω. Αυτή αφορά τη μείωση των αλλιευτικών αποθεμάτων στην Αδριατική θα πρέπει να ακολουθήσουμε το παράδειγμα των φίλων μας της Βαλτικής. Θα πρέπει να προστατεύσουμε όλα τα αλληλευτικά αποθέματα της Αδριατικής και του Ιωνίου Πελάγους. Και ένα άλλο στοιχείο που θα ήθελα να τονίσω είναι ότι στην Αδριατική εξακολουθούμε να έχουμε πολύ καλά ναυπηγεία να ναυπηγούμε πολλά ε, σκάφη αναψυχής, κουραζιερόπλια και είναι σημαντικό διότι απασχολεί ο τομέας χιλιάδες εργαζομένους, αλλά όχι μόνο αυτό, ο τομέας ε, συνδέεται ε, σχεδόν με όλες τις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης διότι χρειάζονται πολλά ανταλλακτικά και, κομμάτια για την αφήγηση των σκαφών και από άλλες χώρες είναι πολύ καινοτόμος τομέας ε, και θα πρέπει να στηριχθεί. Η διασυνδεσιμότητα της περιοχής είναι κάτι πολύ σημαντικό. Η διασύνδεση των μεταφορικών ε, διαδρομών, ε, η, επίσης ο ενεργειακός εφοδιασμός είναι σημαντικά στοιχεία που αφορούν και τις δυτικές και τις ανατολικές ακτές της Αδριατικής. Αυτό είναι σημαντικότατο στοιχείο. Οι διάδρομοι των δικτύων θα πρέπει να συνδέονται με, με άλλα κομμάτια των διευρωπαϊκών δικτύων. Πρόσφατα ξεκίνησαν εργασίες στο ΤΑΝΑΠ και έτσι φυσικό αέριο από το Αζερβαϊτζάν θα φτάνει στην Αλβανία και μέσω Αλβανίας θα εντάσσεται στη μακροπεριοχή αυτή, θα, πηγαίνει, θα καλύπτει και Ελλάδα και Αλβανία. Αναφέρομαι για το Τάνα, αναφέρομαι στο ΤΑΝΑΠ και στο ΤΑΠ. Και τερματική σταθμή για το υγροποιημένο αέριο θα κατασκευαστεί τερματικό θα κατασκευαστούν τερματικά και στην Κροατία και στην Αλβανία για το φυσικό αέριο. Είναι πολύ σημαντικά αυτά, τεράστια σημασία των ε, εγκαταστάσεων των υδροελεκτρικών στη Βοσνία Ζεγοβίνη, στο Μαυροβούνιο και τη Σερβία. Έχουμε πολλά προβλήματα ενεργειακά, ενεργειακής φύσης όπως γνωρίζετε. Ε, η υδροελεκτρική ε, παραγωγή ενέργειας είναι πολύ σημαντική, σημαντικότατη πηγή ενέργειας. Πρέπει να στηρίξουμε την ανάπτυξή της. Η προστασία του περιβάλλοντος ε, είναι και αυτή σημαντικότατη. Προσπάθησα να συμπεριλάβω κάποιες προτάσεις σχετικές. Σημαίνω ότι είναι σημαντικότατη η συνεχής παρακολούθηση της διασυνοριακής ρήπανσης που είναι σε πολύ ψηλά επίπεδα και πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο πρόβλημα αυτό. Μετά, άλλο στοιχείο, στην Αδριατική έχουμε πάρα πολλά υψηλά επίπεδα εκμετάλλευσης όσον αφορά ε, το φυσικό αέριο, το πετρέλαιο και θέλουμε και άλλα προγράμματα έρευνας για αυτές τις ενεργειακές πηγές. Δεν υπάρχει συντονισμένη προσπάθεια, δεν υπάρχει συντονισμός διακρατικός όσον αφορά τις έρευνες για τις ε, πλουτοπαραγωγικές αυτές πηγές. Δηλαδή να δημιουργηθεί ένα περιφερειακό κέντρο, μετά θέλουμε διαπεριφερειακό κέντρο για την αποφυγή των καταστροφών και το προτείνω αυτό δική μου ε, πρωτοβουλία. Ήμουν ομάρχης της περιοχής της Ίστρια και πάντα Είχαμε καλή συνεργασία με την Ιταλία όσον αφορά την πρόληψη των καταστροφών και παρεμβάσεις σε περιπτώσεις καταστροφών και η πρόληψη των καταστροφών και ένα κέντρο προλήψεως καταστροφών πιστεύω θα ήταν με χρησιμότατη προσθήκη στην όλη προσπάθεια που καταβάλλεται για την περιοχή. Η στην Διόζα επίσης αναφέρεται στην ε, έκθεση αυτά τα προβλήματα θα πρέπει να τονίζονται και να υπογραμμίζονται διότι μπορεί να βλάψουν την γεωργία μακροπρόθεσμα. Θα πρέπει επίσης να υπογραμμίσουμε και την αξία της πολιτιστικής κληρονομιάς που προστατεύεται από την UNESCO την Αδριατική ε, και στο Ιόνιο. Ε, ο ελληνικός πολιτισμός, ο ρωμαϊκός πολιτισμός συνέβαλαν τα μάλα στην παγκόσμια κληρονομιά και παρέχονται τεράστιες δυνατότητες για την ανάπτυξη του τουρισμού βάσει των μνημείων που υπάρχουν. Γι' αυτό προτείνω την ε, προετοιμασία μιας μελέτης ενδελεχούς όσον αφορά τις δυνατότητες που υπάρχουν για την εκμετάλλευση της πολιτιστικής κληρονομιάς που υπάρχει σε αυτή την περιοχή και να συμπεριληφθεί στη στρατηγική διότι πιστεύω ότι οι τουρίστες που επιθυμούν να επισκεφθούν αυτές τις περιοχές διαφέρουν. Έχουν διαφορετικές απαιτήσεις. Η πολιτιστική κληρονομιά σίγουρα όμως αποτελεί τον ε, βασικό κοινό παρανομαστή. Ε, αυτό που συζητούμε όσον αφορά τον τουρισμό πιστεύω δεν λαμβάνει υπόψη επαρκώς την πολιτική κληρονομιά όποτε συζητάμε τον τουρισμό. Έχουμε ελκυστική ύπεθρο, έχουμε ελκυστικά νησιά και όλα αυτά θα πρέπει να τα εκμεταλλευτούμε πλήρως. Στο τέλος θέλω να ευχαριστήσω όλους για τη συνεργασία τους και προσβλέπω σε περαιτέρω συζητήσεις οι οποίες θα ακολουθήσουν. Θα προσπαθήσουμε να εξετάσουμε τις τροπολογίες, θα προσπαθήσουμε να καταλήξουμε σε συμβιβαστικές τροπολογίες και το Σεπτέμβριο θα διεξαχθεί η ψηφοφορία. Σας ευχαριστώ πολύ για την υπομονή σας. Thank you. Thank you, Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Γιάκοφτσιτς για αυτή την παρουσίαση. Οι θα ήθελαν το λόγο για να ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Κυρία Τζουφρίντα. Ευχαριστώ Πρόεδρε και εγώ ήθελα να αναφέρω κάποιες σκέψεις. Πάνω απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την έκθεση αυτή που μόλις μας παρουσίασε και τον ευχαριστούμε και για τις προσπάθειες που κατέβαλε αυτά τα χρόνια και τις τελευταίες εβδομάδες πιο συγκεκριμένα που αφορούσε τη δημιουργία της στρατηγικής στην περιοχή. Αντιμετωπίζουμε μια πρόκληση. Η πρόκληση είναι της υλοποίηση της εν λόγω στρατηγική σε στενό συντονισμό με όλου τους εταίρου της περιοχής και σε αυτό το σημείο θα πρέπει να περάσουμε από τη φιλοδοξία που την έχουμε όλοι προς την ε, υλοποίηση διότι η διακυβέρνηση των μακροπεριφερειών είμαι πεπισμένη, σίγουρα είναι η πτυχή πιο κρίσιμη, αλλά ταυτόχρονα είναι η πτυχή που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τόσο ώστε να πετύχουμε στρατηγική, η οποία να είναι αποτελεσματική και να φροντίσουμε τόσο ώστε αυτή η έκθεση να καθορίσει τι απαιτείται, τι πρέπει να δημιουργηθεί, να δημιουργηθεί πραγματική διακυβέρνηση για να υλοποιηθεί ένα συντονισμός που αντιπροσωπεύει ένα είδος ή soft institution, ή ποιου θεσμού για την στρατηγική που συνεπάγεται ένα έλεγχο πραγματικό των επενδύσεων και τη διαθέση των πόρων, ότι προφανώ χρειάζεται κάτι τέτοιο. Είναι σαφέ ότι οι μακροπεριφερειακέ στρατηγικέ πάνω απ' όλα έχουν χαρακτήρα προσέγγιση ε, ε, εδαφική. Ε, είναι μια προσέγγιση πάρα πολύ ισχυρή και πρέπει να αντιστοιχεί στην επικουρικότητα και την αρχή τη εταιρική σχέση. Από την οπτική γωνία πρέπει να γνωρίσουμε ότι θεμελιώδη ρόλο παίζουν οι περιφέρειες για μια προσέγγιση που θα πρέπει να είναι πολυεπίπεδη διακυβέρνηση. Και είναι και το πνεύμα άλλωστε της στρατηγικής αυτό της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης. Πιστεύω ότι είναι θέμα και αξιοπιστία στρατηγικής που παίζει επί της δυνατότητας που έχει στρατηγική της ολοκλήρωση όσον αφορά τους πόρους, τη χρήση των διαθωτικών πόρων για το πρόγραμμα 2014-2020. Είπαν επανειλημμένα ότι η στρατηγική δεν διαθέτει του ίδιου πόρου. Θα πρέπει να καθορίσουμε ότι τα κράτη-μέλη και οι περιφέρειε θα πρέπει να ευθυγραμμίσουν τι πολιτικέ του και του σχετικού πόρου και θα πρέπει να συμπεριλάβουν τη στρατηγική στα προγράμματα συγχρηματοδοτήσεω Ευρωπαϊκή Ενώσεω. Εξασφαλίζοντα έτσι ότι οι στόχοι και οι δράσει στρατηγική τη μακροπεριφερειακή θα επικαιροποιούνται και θα τροφοδοτούνται μέσα των προγραμμάτων. Υπάρχουν μετά πτυχές ή εγκάρσεις που δεν συμπεριλαμβάνονται στους πυλώνες ε, που συζητήσαμε εκτενώς και το έκανε και ο συγκητής, δηλαδή που αποτελούν και τη βάση στρατηγική στα θεμέλια. Μία, ένας από τους πυλώνες είναι η πτυχή της επικοινωνίας, διότι δεν υπάρχει στρατηγική χωρίς αυτή να προωθείται επαρκώ. Χρειάζεται λοιπόν να εγγυηθούμε μια επαρκή ορατότητα σε επίπεδο εθνικό, σε επίπεδο περιφερειακό και πάνω από όλα σε επίπεδο τοπικό. Διότι στρατηγική θα πρέπει έτσι να γίνει αποτελεσματική, να αναπτυχθεί η επικοινωνία και να ευαισθητοποιήσουμε επί των στόχων και των επιτευχθέντων αποτελεσμάτων, να προωθήσουμε την ανταλλαγή των βελτίστων πρακτικών και να διοργανώσουμε και εκδηλώσει που θα εμπλέκουν το σημαντικό το στοιχείο που είναι ο πληθυσμό των εμπλεκομένων περιοχών δεν πρέπει να αφήσουμε όμως τις κοινωνικές πτυχές, την προστιθέμενη αξία της στρατηγικής που είναι ένας στόχος κοινό για την επίτευξη όλων των στόχων. Θα πρέπει να είναι το νήμα της αριάδνης για όλες τις δράσεις για να βελτιώσουμε τη συνεργασία των εργαζομένων, εγγυηθούμε την ισοτιμία των φύλων και την συμπερίληψη των ατόμων με αναπηρία τους πυλώνες για αφορούν τη μεταφορά και τον τουρισμό πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή ακριβώς στην άρση των αρχιτεκτονικών φραγμών και να μπορούν να χαίρονται τις υπηρεσίες και τα άτομα που έχουν κάποια αναπηρία. Ε, αυτό είναι ένα σημάδι της ευαισθησίας μας και τη ιδιαίτερη προσοχή που δίνουμε όσον αφορά τα άτομα που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση. Θα πρέπει να συμπεριλάβουμε επίση την επιχειρηματικότητα των νέων, τι νεοφυεί επιχειρήσει, μικρομεσαίε επιχειρήσει, διότι είναι ένα οικονομικό κόσμο αυτό που όλοι έχουμε μπροστά μα και προ αυτού τρέφονται πολλά μέτρα τα θεματικά, τα συναφή με αυτό. Πρέπει να προσέξουμε κυρίω και την πρόσβαση στι πιστώσει που θα πρέπει με κάθε τρόπο να διευκολύνουμε θα ήταν καλό και σκόπιμο να προβλέπουμε και μια ειδική κατάρτιση των υπαλλήλων της διοίκησης και της κοινωνίας των πολιτών που εμπλέκεται στην επεξεργασία κάθε προγράμματος και ακριβώς γι' αυτό είναι σημαντικό να εξασφαλίζουμε μια επαρκή ε, επαγγελματικότητα όσον αφορά αυτού του τύπου την προσπάθεια μακροπεριφέρειας. Δεν μπορούν να καθορίσουν εκ νέου τις προτεραιότητες που έχει καθορίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα προγράμματά της. Όμως Ιδιαίτερα οι περιοχές έχουν ένα καθήκον να προωθήσουν διάφορα προγράμματα που επιτρέπουν ε, να καλύψουν τις ελλείψεις και να προωθούν καινοτόμα προγράμματα, κυρίως εκείνα τα προγράμματα που οδηγούν στην ανάπτυξη. Προσθέτω μόνο κάποιες μικρές σκέψεις που θα μπορούσαμε να επεξεργαστούμε μαζί με τον εισηγήτη τις επόμενες εβδομάδες και αφορά τους πυλώνες. Όσον αφορά την γαλάζια ανάπτυξη, μου έρχεται στο μυαλό η ανάγκη μια ιδιαίτερη προσοχή που πρέπει να δοθεί όσον αφορά τις περιοχές τις τεχνικές και για τις θαλάσσιες τεχνολογίες. Όλος ο κόσμος της έρευνας σήμερα κοιτάει προς αυτή την κατεύθυνση. Τώρα όσον αφορά την περιβαλλοντική ποιότητα ε, θα πρέπει να χαρτογραφηθούν οι περιοχές, να υπάρξει ε, καθαρισμός των περιοχών που έχουν υποστεί υπερεκμετάλλευση τα χρόνια αυτά, να ελοποιηθεί ένα δίκτυο περιφερειακό ηλεκτροδότησης ε, υψηλής και πολύ ψηλής τάσος που θα διασυνδέεται με σωστή συνεργασία που θα γίνεται όσον αφορά τους, ε, με, τα δίκτυα ανανεώσιμων πηγών ενεργείας. Η αναδάσωση είναι σημαντικό, κυρίως σε κάποιες περιοχές. Ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό, πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Όσον αφορά τον πυλών τη διασύνδεση των περιοχών, συμφωνώ προφανώς με τον εισηγητή που εισάγει την ε, επέκταση βορρά-νότιου του διαδρόμου Σκανδιναβίας Μεσογείου από Πεσκάρα προς Μπάρι και κυρίως του διαδρόμου της Βαλτικής προς την ε, Αδριατική. Να χρησιμοποιηθεί διάδρομος της Μεσογείου η διασύνδεση μεταξύ της Ιβυρική Ιασονίσου Κεντρικής Ιταλίας και Βαλκανίων να συνδεθούν οι περιοχές. Βιώσιμος τουρισμός κατά την άποψή μου θα πρέπει να είναι στο επίκεντρο των προσπαθειών, διότι σίγουρα αποτελεί ένα κομμάτι της, ε, των περαιτέρω οικονομικών εξελίξεων και ανάπτυξης των περιοχών αυτών στο μέλλον και σε αυτόν τον πυλώνα θα προωθούσα πάρα πολύ τη στήριξη των πολιτιστικών βιομηχανιών και δημιουργικών βιομηχανιών. Λοιπόν, υπάρχουν προοπτικές όσον αφορά τις μακροπεριφέρειες αυτές, υπάρχουν μεγάλες προσδοκίες. Είναι ένα τεχνικό εργαλείο συντονισμού των πολιτικών, των διευθυντικών ταμείων της Ευρώπης και πέραν αυτού μπορεί να έχουμε δυτή και πιο φιλόδοξη λειτουργία με στο μακροπεριφερειών. Από τη μία πλευρά μπορούμε να προωθήσουμε την πολιτική περιφερειακή ολοκλήρωση, πολύ συχνά ε, βρίσκεται σε δεύτερη θέση εσείς με την κάθε ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα πρέπει να... Δεν, είναι, δεν ειρήνη σε όλη αυτή την περιοχή. Θα πρέπει να αναπτυχθούν ε, οικονομίες κλίμακα στη διαχείριση των Ευρωπαϊκών Κοινωνικών Ταμείων που μπορούν να χρηματοδοτήσουν ε, ε, κάποια μικρά στρατηγικά προγράμματα, λίγο, μικρό αριθμό στρατηγικών ε, προγραμμάτων και μπορούμε έτσι να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητα των ευρωπαϊκών πόρων. Ε, αυτό πρέπει να στηρίξουμε εμεί. Αυτή είναι η μικρή μα γονίτσα. Όλοι μπορούμε να συνεργαστούμε για να ελοπίσουμε η στρατηγική η οποία θα είναι πραγματικά αποτελεσματική και θα οδηγήσει αυτέ τι περιοχέ σε ευημερία. Ευχαριστώ. Um, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή Ιβαν Γιάκοφτσιτς. Πρόκειται για μια εξαιρετική έκθεση. Είχαμε πράγματι πολύ επιτυχημένη συνεργασία και με τους υπόλοιπους συναδέλφους για την εκπόνηση του σχεδίου έκθεσης. Η περιφέρεια Αδριατικής Ιωνίου αντιμετωπίζει μείζονες προκλήσεις, όπως υψηλά ποσοστά ανεργίας, κακές υποδομές στον τομέα των μεταφορών ε, και περιορισμένες διοικητικές ικανότητες, πολυπλοκότητα, γραφειοκρατία, οικολογικές καταστροφές. Προκειμένου να επιλύσουμε αυτά τα προβλήματα, πρέπει να ζητήσουμε και από ιδιωτικού φορείς και την κοινωνία των πολιτών να συμμετέχουν στην υλοποίηση αυτής της στρατηγικής. Οι πόροι πρέπει να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά στο πλαίσιο της διακυβέρνησης, της στρατηγικής. Το επίπεδο ευαισθητοποίησης για τα ζητήματα αυτά διαφέρει από χώρα σε χώρα. Είπαμε ότι τέσσερις από τις χώρες αυτές της στρατηγικής είναι μέλη της Ένωσης και τέσσερις όχι. Διαφορετικές εμπειρίες λοιπόν Άρα χρειάζεται μια στρατηγική που θα πρέπει να προσαρμοστεί και στο εδαφικό δυναμικό της κάθε μεμονωμένης χώρας. Θα ήθελα να υπογραμμίσω τον πρώτο πυλώνα της στρατηγικής και να μιλήσω για τον αλλιευτικό τομέα. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν πολλοί φραγμοί που καθιστούν αδύνατο να γίνει ε, εκμετάλλευση του πλήρους δυναμικού τομέα. Υπάρχει κατακαιρματισμένη βιομηχανία, περισμένη πρόσβαση και σε άδειες, περισμένη πρόσβαση στο κεφάλαιο. Δεν υπάρχουν επαρκείς πιστώσεις για την καινοτομία, οι διαδικασίες είναι δυσκίνητες. Καλό θα ήταν να υπάρξει συνεργασία με άλλους οικονομικούς τομείς όπως είναι η γεωργία και ο τουρισμός. Αυτό θα πρέπει να απλοποιηθεί και να δραστηριοποιηθούν οι τοπικές ομάδες δράσης έτσι θα υπάρξει μεγαλύτερη διαφοροποίηση. Με τον τρόπο αυτό, ο τοπικός πληθυσμός θα παραμείνει και στα νησιά, που είναι ιδιαίτερα ευάλωτα και οι κοινωνίες τοπικές εκεί είναι ευάλωτες. Πρέπει επίσης να διατηρηθεί η παραδοσιακή πολιτιστική κληρονομιά των τοπικών κοινωνιών που συνιστά προστιθέμενη αξία και μπορεί να προωθηθεί με την ανάπτυξη τοπικών εμπορικών σημάτων και προϊόντων τοπικών. Εν κατακλείδη. Θα ήθελα να θέσω ένα ερώτημα στον εκπρόσωπο της Κομισιόν. Η έλλειψη ε, ανθρώπινου δυναμικού ε, και οι περιορισμένοι πόροι και μέσα μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα και αν ναι, τι ε, μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό. Πρόεδρος να έρθω στους επόμενους ε, σκιώδες. Νομίζω ο επόμενος είναι ο κύριος Μπόκοβιτς. Ναι, ευχαριστώ και ζητώ συγγνώμη που καθυστέρησα. Ουσιαστικά μόλις γύρισα από την περιφέρεια Αδρατικής και Ιωνίου. Ήμουν σε ένα επιχειρηματικό συνέδριο διευθυντών από τη Σερβία, εξού και καθυστέρησα. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον εισηγητή και τους συνεργάτες του. Η έκθεση του κυρίου Γιάκοφτσιτς είναι αρτιότατη, καλύπτει το θέμα της ε, περιοχής αυτής, στρατηγικής και της περιφέρειας Ανδριατικής Ιωνίου. Η περιφερειακή ανάπτυξη ασφαλώς και είναι πολύ σημαντική αναφέρονται και άλλες περιφέρειες που και αυτές είναι σημαντικές. Είμαι βέβαιος ότι οι συνάδελφοι και οι υπόλοιπες επιτροπές που θα καταρτήσουν γνωμοδότηση θα εμπλουτίσουν την έκθεση ακόμη περισσότερο. Όπως προείπα, επισκέφθηκα αυτή την περιφέρεια μόλις επέστρεψα σήμερα το πρωί από εκεί τέσσερις χώρες της περιφέρειας είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τέσσερις όχι. Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα, μία από τις σημαντικότερες ελλείψεις είναι ότι οι χώρες αυτής της ε, περιφέρειας ε, δεν ε, εμπιστεύονται παρκώς η μια την άλλη και το ίδιο ισχύει και τους πολίτες, τους υπηκόους των χωρών αυτών. Και βέβαια αυτό επηρεάζει το συντονισμό και τη συνεργασία μεταξύ των χωρών. Βλέπουμε ότι στην περιοχή της Βαλτικής υπάρχει καλή συνεργασία. Γι' αυτό και θεωρώ ότι η στρατηγική για την περιφέρεια Αδριατικής Ιωνίου θα είναι μια ευκαιρία για την ε, σύμπηξη πιο στενών σχέσεων και επαφών. Ελπίζω να ενδυναμωθεί η διοικητική ικανότητα των περιοχών και των χωρών, ώστε και οι κυβερνήσεις αλλά και οι υπόλοιποι φορεί να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν τις προκλήσει που αναφέρονται στην έκθεση. Ακούσαμε επίσης πολλά για τις οργανωτικές πτυχές. Φυσικά τα κράτη-μέλη είναι σε διαφορετικό επίπεδο οργάνωσης από τις υπόλοιπε τέσσερις χώρες που δεν είναι μέλη της Ένωσης. Με την ανταλλαγή πληροφοριών και καλών πρακτικών και οι υπόλοιπε χώρε τη περιφέρεια πιστεύω θα μπορέσουν να βελτιώσουν τι διοικητικέ του ε, ικανότητε αξιόπεντα τη δική μα τεχνογνωσία. Στο σημείο 7 γίνεται λόγο για την ε, μεγαλύτερη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα διευθυντικά όργανα αυτή τη ε, περιφέρεια. Πώ θα γίνει αυτό, πώς θα μπορέσουμε να συμμετέχουμε σε αυτές τις δομές. Θα πρέπει να τα εξετάσουμε, να τα συζητήσουμε. Στον τομέα του τουρισμού τώρα, θεωρώ ότι οι δυνατότητε είναι τεράστιες, πρέπει να ενισχυθεί όμως το έγγραφο περισσότερο. Σε αυτό το τομέα, το τομέα του τουρισμού, θα πρέπει να προωθήσουμε περιφερειακά προϊόντα που θα σχετίζονται με τον τουρισμό στην Αντριατική, είναι πολύ σημαντικός ο τομέας αυτός. Η χώρα, μεγάλου μεγαλοπόλεις, επίσης μπορούν να έχουν μεγάλη σημασία. σε αυτή την προσπάθεια προώθησης σημαντικών τοπικών προϊόντων. Σε ό,τι αφορά τον τουρισμό, θα πρέπει πιστεύω να υπογραμμίσουμε το γεγονός ότι η Σλοβενία και η Κροατία έχουν το 40% της επικράτειάς τους στο δίκτυο Natura, άρα θα πρέπει να έχουν ακόμη μεγαλύτερες προστασίες στις περιοχές αυτές. Θα πρέπει επίσης οι οικονομικές δραστηριότητες αλλά και οι άλλες δραστηριότητες που έχουν στόχο την προστασία των περιοχών Natura να συνδυαστούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Υπάρχει μεγάλο δυναμικό κάτι ακόμη για τον τουρισμό. Πρέπει να τονίσουμε το γεγονός ότι η τουριστική περίοδος είναι περιορισμένη χρονικά. Είναι εκεί. Θα πρέπει, πιστεύω, και το φθινόπωρο και την άνοιξη να γίνουν πράγματα. επί πολιτικές ναυτιλία συνδέονται με τις παραδόσεις μας, είναι σημαντικές και αυτές οι δραστηριότητες. Θα πρέπει, πιστεύω, να δοθεί μεγαλύτερη σημασία και στον ε, τομέα της αλίας, ιδίως στη μικρή κλίμακα αλίας και τα παραδοσιακά προϊόντα. Θα πρέπει να δοθεί, επαναλαμβάνω, μεγαλύτερη έμφαση στον τομέα αυτό της αλίας. Τώρα, ενέργεια. Φυσικά και θα πρέπει να βελτιωθούν οι υποδομές. Οι περιφέρειε, χώρε περιφέρεια, θα πρέπει να αρχίσουν να σκέφτονται το ενδεχόμενο μια ενεργειακή ένωση. Ο εφοδιασμό σε φυσικό αέριο δεν είναι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Υπάρχουν προβλήματα. Πρέπει να ενισχυθεί η σύνδεση, η ενεργειακή σύνδεση, να βελτιωθούν οι σχετικέ υποδομέ Ο συγκεκριτής αναφέρει δύο χώρες, αλλά νομίζω όλες θα πρέπει να αναφέρονται σε ό,τι αφορά το ενεργειακό δυναμικό. Επίσης, ε, η εξόριξη αναζήτηση πετρελαίου στην Αδριατική επίσης είναι ένα θέμα, θα πρέπει όμως να γίνεται με φιλοπεριβαλλοντικές τεχνολογίες και σε ό,τι αφορά την παροχή ενέργειας. Επίσης έχουμε τις υλικοτεχνικές υποδομές, logistics, Έχουμε τη Ριέκα, την Τεργέστη και το ΚΟΠ που είναι τρία λιμάνια πολύ σημαντικά στη Βόρεια Αδριατική, τρία σημεία εξόδου από την Ευρώπη στα άλλα πελάγια, στις άλλες θάλασσες, θα πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα τις λιμενικές υποδομές, θαλάσσιες υποδομές και σίγουρα θα πρέπει να υπάρξουν συνέργειες μεταξύ των λιμένων. Νομίζω ότι και με τις τροπολογίες μας θα συνεισφέρουμε στο να έχουμε τελικά μια εξαιρετική έκθεση για τη στρατηγική της Περιφέρειας Ανδρετικής Ιωνίου. Η Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Ολοκληρώσαμε με τους κοιόδους. ο Παδημούλης τώρα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Γιάκοφτσης ε, για την εργασία που έχει κάνει. Είχαμε μια εξαιρετική συνεργασία και με μένα ως κοιόδη εισηγητή της πολιτικής μου ομάδας ε, και πιστεύω ότι και με τη σημερινή συζήτηση και με τις τροπολογίες που θα κατατεθούν μπορούμε να καταλήξουμε σε ένα κείμενο που να, δώσει, να δώσει όθηση σε αυτή την ε, στρατηγική συνεργασία στην περιοχή της Αδριατικής και του Ιωνίου. Έχουμε άλλωστε ένα θετικό παράδειγμα. Το παράδειγμα των χωρών της Βαλτικής που εξασφάλισαν μια αποδοτική συνεργασία και έχουν πετύχει θετικές συνέργειες εποφελία της ανάπτυξης ε, των χωρών του. Θα ήθελα πριν περάσω σε θετικές επισημάσεις να υπογραμμίσω ορισμένες δυσκολίες που έχει το εγχείρημα γιατί με αυτές αναμετριόμαστε. Μην ξεχνάμε ότι είναι μια έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που θέλει να δώσει όθηση σε κάτι που είναι αναγκαίο όσοι προηγήθηκαν και ο κ. Γιάκοφτης και οι σκιώδεις ηγητές των άλλων πολιτικών ομάδων επεσήμαναν σωστά και αυτονόητα πράγματα. Ότι εδώ χρειάζεται συνεργασία, οικονομίες κλίμακας, συνέργειες, με στόχο το κοινό και την ανάπτυξη μιας περιοχής που έχει σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα και δυνατότητες συνανάπτυξης. Θα ήθελα εγώ να σταθώ στις δυσκολίες η πρώτη δυσκολία υπόθηκε ήδη. Είναι τέσσερις χώρες που είναι ήδη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τέσσερις χώρες που δεν είναι. Μεγάλες διαφορές επιπέδων ικανότητας στη διοίκηση. Ιστορικά κληρονομημένες δυσπιστίες. Περιορισμένοι πόροι. Δεν υπόθηκε, αλλά όλοι το ξέρουμε δεν υπάρχει καινούριο φρέσκο χρήμα για την ενίσχυση αυτής της πρωτοβουλίας. Θα πρέπει να αξιοποιηθούν οι υπάρχοντες πόροι, τα υπάρχοντα χρηματοδοτικά εργαλεία. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να γίνει πολύ αυστηρή ιεράρχηση και επιλογή από κοινού, από όλες τις χώρες, των επενδύσεων που θα πραγματοποιηθούν, που θα πάνε τα χρήματα. Και αυτό απαιτεί καλή συνεργασία και ικανότητα επιλογών. Γιατί εάν προγραμματιστούν περισσότερα από αυτά που μπορούν να χρηματοδοτηθούν, θα μείνουν μισοτελειωμένα έργα. Και αυτό δεν θα βοηθήσει καθόλου ε, στην ε, ανάπτυξη. Νομίζω ότι θα πρέπει να εστιάσουμε ιδιαίτερα και το κάνει ο κ. Γιάκοφτης στους τομείς όπου είναι ολοφάνερο ότι η συνεργασία δημιουργεί ε, οικονομίες κλίμακας και οθεί την ανάπτυξη. Μεταφορές, ενέργεια, τουρισμός, προστασία του περιβάλλοντος που δίνει και βιωσιμότητα στα θέματα της ανάπτυξης. Μην ξεχνάμε ότι μιλούμε για μια περιοχή που και οι χώρες που είναι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οι χώρες ακόμη περισσότερο που είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης αντιμετωπίζουν μεγάλα προβλήματα περιορισμού πόρων, υψηλής ανεργίας, χαμηλού επίπεδου όχι μόνο την ε, ανάπτυξη των υποδομών τους αλλά και στο βιωτικό επίπεδο των λαών τους. Και έχει σημασία αν θέλουμε να ξεπεράσουμε τις δυσπιστίες οι επενδύσεις που θα γίνουν να δημιουργούν την αίσθηση στους πολίτες ότι πιάνουν τόπο τα λεφτά. Αλλά για να γίνει αυτό πρέπει να βοηθήσουν περισσότερο και αυτοί που έχουν επιπλέον χρήματα. Και έχει σημασία και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το νέο ταμείο που δημοσιογραφικά ονομάζεται Ταμείο Juncker, το EFSI, να ενισχύσει αυτές τις προσπάθειες. Και νομίζω κύριε Γιάκοβιτς ότι πρέπει να βρούμε τρόπο να εξασφαλίσουμε, και αυτό απαιτεί πιο συγκεκριμένη πρόταση, την συμμετοχή του Ευρωκοινοβουλίου στη διοίκηση αυτού του σχήματος, ειδικά στα πρώτα βήματα, έτσι ώστε να μπει σε μια σειρά, να μπει το νερό στα βλάκι, να δρομολογηθούν τα πράγματα. Ορισμένες τώρα επιμέρους παρατηρήσεις θα ήθελα να κάνω. Η πρώτη είναι ότι θεωρώ εξαιρετικά καλή την ιδέα να υπάρξει, να καθιερωθεί ένα ευρωπαϊκό έτος νησιωτικών και ορεινών περιοχών που υπάρχει ε, στην, ε, στην έκθεση και θα ήθελα σε αυτό το θέμα, μιας και η πρόταση αφορά και προς την Κομισιόν, να ακούσω και τη γνώμη της Κομισιόν. Ένα δεύτερο θέμα είναι ότι κάνετε μια αναφορά στην έκθεση, κύριε Γιάκοφ, στο θέμα των μεταναστευτικών ροών. Χώρες όπως η Ιταλία και η Ελλάδα δέχονται μεγάλη πίεση μεταναστευτικών ροών και πρέπει να ενταχθεί ε, συμπληρω... Ε, στον τομέα αυτό να συμπληρώσουμε με την ανάγκη δημιουργίας δομών υποδοχής ε, των, των μεταναστών με ευρωπαϊκή στήριξη. Επίσης θα προτείνω και μέσω τροπολογιών να ενισχύσουμε στην ισορροπία του κειμένου τους στόχους μιας βιώσιμης ανάπτυξης και της δημιουργίας θέσεων εργασίας και ιδιαίτερα της, του περιορισμού της ανεργίας των νέων. Και τέλος, επειδή μιλάμε για μια συνεργασία που είναι έχει δυσκολίες να ξεκινήσει, τέσσερις χώρες μέλη, τέσσερις χώρες μη μέλη, νομίζω ότι η όποια διεύρυνση πρωτοβουλειών ε, της στρατηγικής αυτής συνεργασίας και με άλλες χώρες πέραν των οκτώ γειτονικέ θα πρέπει να γίνει με προσοχή αφού έχουν δρομολογηθεί τα πρώτα βήματα και έχει προχωρήσει αυτή η υλοποίηση της συνεργασίας με σύμφωνη γνώμη όλων των χωρών για να αποφύγουμε τα προβλήματα μιας βιαστικής ε, που θα δυσκολέψει την υλοποίηση των στόχων που θέτει η έκθεση ε, ε, θα περιοριστώ σε αυτές τις παρατηρήσεις, θα καταθέσουμε τροπολογίες και πιστεύω ότι όπως είχαμε μέχρι τώρα μια πολύ επικοδομητική συνεργασία και στη σύνταξη της έκθεσης, με τον ίδιο τρόπο θα διαχειριστούμε και τις ε, τροπολογίες που θα κατατεθούν από όλες τις πολιτικές ομάδες προκειμένου να έχουμε ένα ντοκουμέντο που και θα εγκριθεί με μια ευρύτατη συμφωνία και θα πιέσει και άλλους θεσμούς όπως η Κομισιόν, η Ευρωπαϊκή ε, Τράπεζα Επενδύσεων, το EFSI να δώσουν μεγαλύτερη προσοχή και χρηματοδοτική στήριξη στα επενδυτικά σχέδια αυτής της στρατηγικής συνεργασίας. Ευχαριστώ. Thank you. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Ρισκλέρκ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή κύριο Γιάκοφτιτς για την εξαιρετική βάση που δημιούργησε και επεξεργάστηκε και είμαι σίγουρος ότι η τροπολογίες μας θα εμπλουτίσουν και θα βελτιώσουν ακόμα περισσότερο το σχέδιο έκθεσης. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω και ε, τους ε, ηγητές για την εξαιρετική συνεργασία που είχαμε στις τελευταίες συναντήσεις. Τώρα, ως προς το περιεχόμενο, θα σας αναφέρω τις ε, τροπολογίες που σκοπεύουμε να υποβάλουμε. Θεωρώ ότι κύριο μέλημά μας πρέπει να είναι η φροντίδα της συνεργασίας και του συντονισμού. Ε, είδαμε ότι στην περιοχή της Βαλτικής και στην ε, περιοχή του Δούναβη είχαμε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία και μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε ως ε, καλό παράδειγμα και βέλτιστη πρακτική. Οι μακροπεριφέρειες μας δίνουν τη δυνατότητα να ακολουθήσουμε ε, κοινούς στόχους. Τώρα σχετικά με την ε, χρηματοδότηση και τα κονδύλια φυσικά θα μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε και θα έπρεπε να χρησιμοποιήσουμε το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Επίσης σημαντικό είναι η διασυνοριακή συνεργασία να τονιστεί. Υπάρχουν σχετικά ταμεία που προωθούν την συνεργασία και πιστεύω πως εδώ θα μπορούσαμε να τα χρησιμοποιήσουμε έτσι ώστε να βελτιώσουμε την στρατηγική μας αντιμετώπιση. Και έπειτα, ενεργειακή ένωση. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ενεργειακή απόδοση είναι όροι πάρα πολύ σημαντική για την περιοχή και πιστεύω πως χρειάζονται επενδύσεις για συγκεκριμένα στρατηγικά προγράμματα και εδώ η συνεργασία είναι αναπόσπαστο κομμάτι της στρατηγικής μας. Είναι σημαντικό επίσης να προσελκύσουμε ιδιωτικές επενδύσεις και εδώ πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το σχέδιο Juncker διότι σε τελική ανάλυση για την ολοκλήρωση των προγραμμάτων χρειάζονται οι ιδιωτικές επενδύσεις. Επίσης θα ήθελα να αναφέρω ότι οι μακροπεριφέρειες αυτές έχουν τεράστιο δυναμικό και σε φυσικούς πόρους. Γι' αυτό λοιπόν είναι πολύ σημαντική η στρατηγική Ευρώπη 2020 και υπάρχει η γαλάζια ανάπτυξη, ένας πολύ σημαντικός πυλώνας αυτής της στρατηγικής. Ας μην ξεχνάμε όμως και την πράσινη ανάπτυξη που μπορεί να φέρει καινοτομία και πρόοδο στην ε, περιφέρεια αυτή, μέρος της οποίας είναι και η αλληλεία. Υπάρχουν διάφορες δυνατότητες στήριξης και προώθησης ε, της ε, αλληλείας σε συνδυασμό πάντα με την προστασία του περιβάλλοντος, την προώθηση και τη στήριξη της επιχειρηματικότητας. Είναι δηλαδή πάρα πολύ σημαντικό η αλληλεία να είναι και βιώσιμη και να ακολουθεί την παράδοση των περιφερειών αυτών. Το 40% των αλλιευμάτων που καταναλώνονται στην Ευρώπη προέρχεται από ε, εισαγωγές. Γι' αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντική προώθηση της βιώσιμης αλληλείας για μια πιο υγιεινή διατροφή. Σχετικά με την γαλάζια ανάπτυξη τώρα, χρειάζεται προσοχή για την ε, παραγωγή καθαρής ενέργειας και καθαρών ε, τροφίμων. και τα προϊόντα που θα παράγονται στις ε, περιοχές αυτές, στις παράκτιες περιοχές αυτές θα μπορούν να ε, χρησιμοποιηθούν και να εξαχθούν και στις ε, χώρες που βρίσκονται στην ενδοχώρα, που δεν έχουν πρόσβαση στη θάλασσα. Και είναι πολύ σημαντικό επίσης να στηρίξουμε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Τώρα, όσον αφορά την, υποδομέ, ε, τις υποδομές, χρειάζεται φυσικά ε, μεγάλη προσοχή στην ε, βελτίωση του δικτύου μεταφορών. Ένα πολύ αδύναμο σημείο της περιοχής είναι η έλλειψη σιδηροδρομικής σύνδεσης υψηλής ταχύτητας. Και χρειάζεται επίσης βελτίωση του δικτύου αυτοκινητοδρόμων. Περιβάλλον τώρα. Η διαχείριση των απορριμμάτων είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Όμως έχουμε το παράδειγμα της Βαρκελόνης, η οποία είναι μια πάρα πολύ καθαρή πόλη και έχει να μας διδάξει πάρα πολλά σε σχέση με την περιβαλλοντική χρηστή διαχείριση των απορριμμάτων. Και στο σημείο αυτό θα ήθελα να τονίσω πως δεν πρέπει να ξεχνάμε τα νησιά της ε, περιοχής Αδριατικής Ιωνίου. Εκεί χρειάζονται περισσότερες επενδύσεις από τις ε, υπάρχουσες και γι' αυτό λοιπόν πρέπει να κοιτάξουμε καλύτερα το θέμα της χρηματοδότησης. Σχετικά με το περιβάλλον, πρέπει επίσης να μην ξεχνάμε ότι εκτός από τις θάλασσες υπάρχουν και οι λίμνες. οι οποίες είναι ε, εξίσου σημαντικές και έχουν μεγάλο δυναμικό ε, για την ε, περιφέρεια. Χρειάζεται επίσης να δοθεί προσοχή στην προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Χρειάζεται αύξηση της αποδοτικότητας των πηγών αυτών. διότι έτσι θα αυξηθεί η ενεργειακή ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και μπορούμε να δούμε ότι στα προγράμματα κοινού ενδιαφέροντος περιλαμβάνονται μόνο η Ελλάδα και η Κροατία, αλλά όχι η Αλβανία, η οποία δεν ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και όταν γίνεται λόγος για αυτούς τους πόρους, πρέπει επίσης να μην ε, ξεχάσουμε να αναφέρουμε κάποια προγράμματα για την ε, διερεύνηση των ε, δυνατοτήτων που έχουμε για φυσικό αέριο και στην Ιταλία και στην Κροατία, αλλά και στην ακτή της Ελλάδας και της Αλβανίας. Φυσικά, τηρώντας πάντα την αρχή της βιωσιμότητας. Και επίσης χρειάζεται προσοχή στις ευάλωτες περιοχές, σε κάτι που συνδέεται και με τη γαλάζια ανάπτυξη. Υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια για την ε, διερεύνηση δυνατοτήτων εξαγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου και πρέπει να, αερίου και πρέπει να τα ακολουθήσουμε. Ε, αναφέρθηκαν επίσης οι ικανότητες για την μακροπεριφερειακή στρατηγική από την προηγούμενη σκιώδη γήτρια. Θεωρώ πως όταν θα φτάσουμε στο σημείο να ψηφίσουμε την οδηγία αυτή, πρέπει να λάβουμε υπόψη όλα τα προγράμματα τα οποία έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή. Και πρέπει να ξέρουμε πώς ακριβώς θα συνεχιστούν αυτά τα προγράμματα. εργοστάσια παραγωγής ενέργειας στα κράτη-μέλη και στα μη κράτη-μέλη είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικά και όλοι πρέπει να δεσμευτούν για την καταπολέμηση της ε, κλιματικής αλλαγής. ιδιαίτερα εν ώψη των ε, αλλαγών που πρέπει να γίνουν μέχρι το 2030. Γι' αυτό λοιπόν προτείνω να καταρτιστεί μια μακροπεριφερειακή στρατηγική η οποία θα δεσμευτεί για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και θα έπρεπε ίσως να δημιουργηθεί ένα ταμείο αλληλεγγύης το οποίο θα συντράμει όχι μόνο στην ε, πρόληψη της κλιματικής αλλαγής και στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, αλλά και στην βοήθεια των κρατών που θα υποφέρουν περισσότερο από την κλιματική αλλαγή. Και τέλος, σχετικά με τον τουρισμό. Εγώ δεν θα ε, χρησιμοποιούσα την αναφορά στις, ε, στους διαφορούς ε, τρόπους διασκέδασης που θα πρέπει να παρέχονται στους ε, τουρίστες. Οι τουρίστες έχουν υψηλή κινητικότητα όταν κάνουν διακοπές. Γι' αυτό λοιπόν ίσως θα έπρεπε να προωθήσουμε τις ε, μεταφορές και την κινητικότητα στα πλαίσια του τουρισμού, την ε, μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος. Επίσης, στην Αδριατική και στο Ιόνιο βρίσκονται πολλά νησιά και υπάρχουν πάρα πολλά προγράμματα που έχουμε αυτή τη στιγμή για να ενισχυθεί η ανεξαρτησία των ε, νησιών αυτών και πρέπει να συμπεριληφθούν και οι τοπικές ε, κοινότητες ε, για την επίτευξη του στόχου της ενεργειακής ανεξαρτησίας. εκπαιδευτικά προγράμματα θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην ευαισθητοποίηση και την ενημέρωση του κοινού για την προστασία του περιβάλλοντος. Αυτές είναι εν ολίγης οι τροπολογίες που θα προτείνω. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ανταμάτο. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για το σχέδιο έκθεσης που αφορά την στρατηγική η οποία αφορά μια περιφέρεια με πολλά εκατομμύρια κατοίκους και τέσσερις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα ήθελα και εγώ να τονίσω πως είναι πάρα πολύ σημαντική αναφορά στον ε, τουρισμό, στην ανάπτυξη των υποδομών και των μεταφορών και την προστασία του περιβάλλοντος. Είναι θέματα τα οποία ε, συνδέονται στενά μεταξύ τους και πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε ως ε, σύνολο. θα μπορούσαμε να προτείνουμε κάποια προγράμματα ε, για την ενέργεια, για παράδειγμα, ε, για την διασύνδεση ενεργειακών προγραμμάτων, προγραμμάτων μεταφορών και προγραμμάτων προστασίας του περιβάλλοντος. Και να προσπαθήσουμε να συνδυάσουμε στο σχέδιο έκθεσης όλες αυτές τις ε, πτυχές. Επίσης, ε, ενεργειακή ανεξαρτησία. Είναι πολύ σημαντικό να τονιστεί η ενεργειακή ανεξαρτησία ιδιαίτερα χρησιμοποιώντας φυσικό αέριο. Γι' αυτό λοιπόν και εγώ συμφωνώ πως πρέπει να ε, διεξάγουμε έρευνες για την δυνατότητα εξαγωγής φυσικού αερίου ή πετρελαίου. Αλλά χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή για να μην ε, καταστραφεί το περιβάλλον και η αλληλεία ιδιαίτερα στην περιοχή αυτή η οποία ήδη αντιμετωπίζει προβλήματα. Χρειάζεται λοιπόν μια βιώσιμη ενεργειακή πολιτική. Και αναφέρομαι κυρίως στην ακτή της Αδριατικής, όμως και στο Ιόνιο. Χρειάζεται προσοχή. ο αγωγός φυσικού αερίου θα εξυπηρετήσει όλη την περιοχή, θα καταλήξει στην περιοχή της Πούλια στην Ιταλία και χρειάζονται επενδύσεις. Επενδύσεις όμως που θα ε, επικεντρώνονται σε ένα αποκεντρωμένο ε, μοντέλο διοίκησης που θα δίνει προσοχή στις επιμέρους περιοχές της ε, μακροπεριφέρειας και χρειάζεται επίσης να βρεθούν εναλλακτικές λύσεις ε, για την ε, ενεργειακή αλλαγή και την ενεργειακή ασφάλεια. Γι' αυτό λοιπόν ε, πιστεύω πως πρέπει επίσης θα πρέπει να δούμε τι κάνουμε με την Γεωργία. Θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι λοιπόν, όχι μόνο σε επίπεδο των 100 μελών που εμπλέκονται, αλλά σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, προτείνοντα και εδώ κάποιε λύσει, παραδείγματο χάρη, το δρόμο της βιολογικής γεωργίας και της βιώσιμης ε, γεωργίας. Κάτι τελευταίο, εγώ θα συμφίλω να, θα πρότεινα να, το, την οικοδόμηση της γέφυρας της Μεσίνης να το αφήσουμε. δεν είναι από τα θεμελιώδη σημεία. Ε, είναι ένα πρόγραμμα, πώς να το πω, που δεν μπορούμε καν να το παρουσιάσουμε. Προτείνω και στους συναδέλφους να μελετήσουμε λίγο μαζί ε, την διαγραφή αυτής της προτάσεως στις ε, κατευθύνες γραμμές. Ουσιαστικά οι προκλήσεις, κρίσιμα στοιχεία και οι δυνατότητες που αφορούν ε, την περιοχή αυτή είναι τεράστιες. Θα πρέπει να συνεργαστούμε και αν συνεργαστούμε θα κάνουμε μια πάρα πολύ καλή δουλειά. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Μάλετιτς έχει το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Για να είμαστε πιο γρήγοροι θα μιλήσω αγγλιστή. Ευχαριστώ τον εισηγητή για το σχέδιο εκθέσεως και όλους τους ε, σκιώδεις ε, έχουν κάνει έξοχα σχόλια. Θα ήθελα να τονίσω τη σημασία που έχει η εφαρμογή και η υλοποίηση της ε, στρατηγικής και θα πρέπει να σκεφτούμε το πώς η εφαρμοστική δομή θα δημιουργηθεί και νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να κινηθούν ταχύτερα και να εργαστούν σκληρότερα στον αυτό το θέμα. Υπάρχουν πολλές ανησυχίες, πολλές από τις ανησυχίες που αφορούν την εφαρμογή και υλοποίηση ήδη έχουν ε, αναφερθεί. Μιλήσατε για διοικητικό δυναμικό που αν δεν είναι καλό οδηγεί σε κακή εφαρμογή, αδύναμη εφαρμογή και είναι δυσκολότατο να καθορίσουμε κοινούς στόχους στις χώρες που είναι σε διαφορετικό επίπεδο αναπτύξεως, έχουν διαφορετικές ανάγκες και εξ αυτού ο κοινός στόχος, η υλοποίηση των κοινών στόχων δεν είναι και τόσο εύκολο στην πράξη και εγώ γι' αυτό μιλώ κυρίως για την υλοποίηση. Δεν έχουμε επίση συγκεκριμένους κανόνες και διαδικασίες σε όλες τις χώρες διότι έχουμε τεράστια ποικιλία στις χώρες και θα πρέπει αυτό να το επεξεργαστούμε και να δούμε πώς μπορούμε να υλοποιήσουμε τις προσεγγίσεις στις χώρες και ε, ε γι' αυτό είναι και πιο δύσκολη η εφαρμογή λόγω των διαφορών. Αυτό που χρειαζόμαστε για έγκαιρη και σωστή εφαρμογή είναι καλά δομημένα έργα και προγράμματα τα οποία θα οδηγήσουν σε εκπλήρωση των καθοριστέντων στόχων της στρατηγικής και μπορούμε να πούμε ότι έχουμε κατάλογο προγραμμάτων. Το πρόβλημα είναι έχουμε καλά δομημένα και έτοιμα προς εφαρμογή προγράμματα. Από εκεί θα πρέπει να ξεκινήσουμε. Όταν λέω καλά δομημένα έργα και προγράμματα θεωρούμε ότι με τα προγράμματα που έχουμε στον κατάλογο εκπληρώνουμε στόχους που είναι σημαντικοί για τη μακροπεριφέρεια στο σύνολό τη ή εξακολουθούμε να πιστεύουμε ε, να έχουμε απόψεις που βασίζονται σε εθνικά συμφέροντα πρώτα και μετά στα συμφέροντα της μακροπεριφέρειας. Αυτά πρέπει να τεθούν και όσον αφορά την πηγή της ε, χρηματοδότησης θα πρέπει και εμείς και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή μάλλον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τελευταία, και αυτοί και εμείς σκεφτόμαστε για νέα χρηματοδοτικά μέσα και πώς να βρούμε πηγές ε, χρηματοδότησης και να ανοίξουμε τη χρηματοδότηση για τους επιχειρηματίες. Ίσως μπορούμε να σκεφτούμε πώς μπορούμε να δομήσουμε και να δημιουργήσουμε συγκεκριμένο ταμείο για προγράμματα στη μακροπεριφέρεια, όπως για τις χώρες της Βαλτικής έχουν ένα κοινό ταμείο για την ε, χρηματοδότηση ε, έργων του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα και το συνδυασμό αυτών των έργων από αυτό το ταμείο. Θα ήταν καλό λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε και τις πηγές της συνοχής και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και οι πηγές να συνδυαστούν στο νέο χρηματοδοτικό αυτό ε, μέσο. Νομίζω ότι είναι σημαντικότατο να έχουμε συγκεκριμένο ταμείο, πόρο που θα βοηθά την υλοποίηση των έργων. Πρώτα απ' όλα όμως χρειαζόμαστε έναν κατάλογο καλά δομημένων έργων. Θα έπρεπε μετά να δούμε πώς μπορούμε να στηρίξουμε τις αλλαγές και τις μεταρρυθμίσεις και ταχύτερη ανάπτυξη στις χώρες ε, που είναι λιγότερο ανεπτυγμένες και έχουν κάποια διαφορετικές απόψεις για κάποιες κοινέ πολιτικές που ήδη έχουν καθιερωθεί στα κράτη-μέλη, αλλά όχι στις χώρες που δεν είναι μέλη. Αυτή η ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών θα πρέπει να λάβει χώρα και στην πράξη. Στο τέλος, όταν μιλούσα για νέα χρηματοδοτικά εργαλεία και πώς μπορούμε να εξετάσουμε το ενδεχόμενο νέου ταμείου, θα ήθελα να πω ότι στις 8 χώρες αυτές έχουμε τεράστιο κατακαιρματισμό των χρηματοπιστωτικών αγορών. Εξ αυτού δεν έχουμε επιχειρηματίες που έχουν τις ίδιες ευκαιρίες. Δεν έχουν τις ίδιες ευκαιρίες όσον αφορά την υλοποίηση των έργων και των προγραμμάτων, διότι έχουμε τεράστιες διαφορές που υπάρχουν όσον αφορά τα επιτόκια, τις δυνατότητες χρήσεως της χρηματοδοτήσεως για τα διάφορα έργα υπάρχουν πολλά εμπόδια στα μη κρατη αλλά και σε κάποια όπως στην Κροατία παραδείγματο χάρη. Και αυτό θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ο κύριος Ανδρέα Μέιρέιτ αν το προφέρω σωστά είστε εδώ Ορίστε. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα θέλαμε να καλωσορίσουμε την έκθεση του αξιότιμου μέλους του Κοινοβουλίου, του κυρίου Τζάκοτσιτς και συμφωνούμε με το μεγαλύτερο τμήμα του περιεχομένου της εκθέσεως θα θέλαμε να προβούμε σε τρία σχόλια. Το πρώτο. Στη διακυβέρνηση θα πρέπει να φέρουμε και τα εθνικά κοινοβούλια. Πρέπει να ενισχυθούν οι σχέσεις με τα εθνικά κοινοβούλια. Γιατί, διότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει σημαντικό ρόλο για το στατηγικό συντονισμό της στατηγικής, αλλά εξαρτάται και από τα κράτη-μέλη η απόφαση περί των βασικών στοιχείων της στρατηγικής, ούτω ώστε να εξασφαλίζεται η ανάληψη των ευθυνών για τη στρατηγική. Πιστεύουμε ότι τα Εθνικά Κοινοβούλια μπορούν να παίξουν και σημαντικό ρόλο όσον αφορά την ευαισθητοποίηση περί της στρατηγικής. σε πολιτικό επίπεδο και να αυξήσουν επίσης την ορατότητα των προσπαθειών σε κάθε χώρα. Είναι σημαντικό αυτό για την ευθυγράμμιση των εθνικών πολιτικών, των επενδυτικών σχεδίων και των προγραμμάτων, κυρίως στις υποψήφιες και δυνάμει υποψήφιες χώρες, ε, για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής. Και είναι σχετικό και με την ευθυγράμμιση των χρηματοδοτήσεων, της χρήσης των εθνικών και περιφερειακών πόρων και των επιχειρησιακών προγραμμάτων των χωρών και των περιοχών που είναι βασική πηγή χρηματοδοτήσεως. Η χρηματοδότηση μπορεί να ευθυγραμμιστεί και να στηρίξει και τη στρατηγική και τους σχετικούς στόχους. Δεύτερον, διοικητικό δυναμικό. Αναφέρθηκε αυτό. Και μάλιστα από αρκετά μέλη. Θα θέλαμε να τονίσουμε το εξής. Έχουμε υπερεθνικό πρόγραμμα, το Adrian, που καλύπτει την ίδια γεωγραφική περιοχή. Μπορεί αυτό να στηρίξει το διοικητικό δυναμικό μέχρι μέσω ειδικού μέσου που θα βρίσκεται το σημείο το αρμόδιο στη Σλοβενία και θα διαθέτει το 10% του προϋπολογισμού, δηλαδή 10 εκατομμύρια για τη στήριξη του διοικητικού δυναμικού, της διακυβερνήσεως και της ε, υλοποίησεως της στρατηγικής. Θα θέλαμε επίσης να τονίσουμε και κάτι άλλο. Κάθε συμμετέχουσα χώρα υπέχει ευθύνη. Ευθύνη να εξασφαλίσει επαρκής και ικανούς διοικητικούς πόρους για την υλοποίηση της στρατηγικής για την Αδριατική και το Ιόνιο. Νομίζω ότι αυτό είναι ουσιαστικό αν θέλουμε να εξασφαλίσουμε επαταλεσματική εφαρμογή και υλοποίηση της στρατηγικής. Τρίτο σημείο που θα ήθελα να τονίσω. Σε προηγούμενες στρατηγικές, στη στρατηγική για τη Βαλτική, για, στη στρατηγική για το Δούναβι επίσης, υπήρξε διαθέσιμη χρηματοδότηση για την έναρξη της εφαρμογής για τη δρομολόγηση προπαρασκευαστικών μελετών. Θα θέλαμε, λοιπόν, ή δυνατόν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να στηρίξει επίσης παρομοίως την υλοποίηση της στρατηγικής για την Αδριατική και το Ιόνιο. Με τον ίδιο τρόπο να τονωθεί η εφαρμογή και η υλοποίηση και να υπάρξει μια στέρεη βάση για ιδιωτικοποιήσει, επιλογή προγραμμάτων και έλεγχο της υλοποίησης της στρατηγική. Αυτά και ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Γιάκοφτσιτ θα ήθελε να δώσει κάποιε απαντήσεις ενδεχομένω. Yes, okay. Μάλιστα. Πρώτα απ' όλα θέλω να σας ευχαριστήσω όλους τους αγαπητοί συνάδελφοι για την συμμετοχή σε στη συζήτηση. Θα είμαι πολύ σύντομος. Να ευχαριστήσω και τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Γιατί συναντηθήκαμε και με την Κομισιόν και ήταν καλή συνεργασία που είχαμε. Και πολύ σωστά τα είπε μόλις πριν ο εκπρόσωπος της Κομισιόν. Ελπίζω ότι θα δοθούν τα αρχικά κονδύλια για την υλοποίηση της στρατηγικής. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους που συνεργάστηκαν μαζί με την κατάρτιση του σχεδίου έκθεσης. Είναι εδώ η κυρία Ρώσα Νταμάτο. Συνεργάστηκα πολύ με το γραφείο της. Υπάρχουν βέβαια κάποιες ε, μικροδιαφορές και μικροδιαφωνίες μεταξύ μας, αλλά νομίζω ότι θα καταλήξουμε στο τέλος ένα πολύ καλό έγγραφο. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη σίγουρα το πρόβλημα της μετανάστευσης. Είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, ένα πρόβλημα που το έχουμε συζητήσει πολλές φορές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. και τα όσα ανέφερε ο κ. Παπαδημούλη σίγουρα θα πρέπει να τα συμπεριλάβουμε στην έκθεση. Τουρισμός, περιβάλλον. Αναφέρθηκαν πολλά, τα οποία είναι σίγουρα σημαντικά, απλά δεν μπορούσα όλα να τα αναφέρω, γιατί είχα περιορισμό στις 6.000 λέξεις. Δεν νομίζω όμως ότι είναι ανυπέρβλητα τα εμπόδια και οι διαφορές μας χωρίζουν. Θα ήθελα λοιπόν να ζητήσω από όλους και δύο από τους κοιόδης να μου δώσουν τροπολογίες για να δω ακριβώς ε, στο χαρτί ποιες είναι οι ιδέες σας και να μπορέσω να τις συμπεριλάβω στην έκθεσή μου. Ολοκληρώνοντας, θα ήθελα να πω ότι στο εισαγωγικό κομμάτι και συγκεκριμένα στο σημείο 5 αναφέρω την ΕΤΕΠ, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα σε συνεργασία με την ΟΠΤΡΕΠΗ, να εξετάσει τη δυνατότητα δημιουργίας ειδική επενδυτικής πλατφόρμας για τη στρατηγική. Δεν μιλάω συγκεκριμένα για κάποιο ταμείο, μιλάω όμως για την ΕΤΕΠ και τη δημιουργία μιας επενδυτικής πλατφόρμας. Δεν ξέρω, μπορούμε να το πούμε κάπως αλλιώς. Ήταν λίγο πιο γενικός όρος που χρησιμοποίησε. Υπάρχει σίγουρα μεγάλο πρόβλημα ανεργίας και στις χώρες μέλη αλλά και κυρίως αυτές που δεν είναι μέλη της Ένωσης. Οπότε νομίζω ότι θα ήταν καλό να δούμε πώς μπορεί να προσελκυστεί το ιδιωτικό κεφάλαιο. Βασίζομαι και στη δική σας συνεργασία λοιπόν, Πρόεδρος. Σας ευχαριστώ και εγώ για την πολύ αναλυτική αυτή συζήτηση. Προθεσμία κατάθεση τροπολογιών Παρασκευή 3 Ιουλίου 12 το μεσημέρι. Ψηφοφορία στην Επιτροπή μας στις συνεδρίες του Σεπτεμβρίου. Περνάμε τώρα στο επόμενο σημείο της μερισιάς διάταξης που είναι ανταλλαγή απόψεων με τη διάσκεψη των παράκτιων περιφερειακών περιοχών της Ευρώπης. Η διάσκεψη των παράκτιων περιφερειακών περιοχών της Ευρώπης η 1973 είναι μια ομάδα προβληματισμού, μια δεξαμενή σκέψης που εκπροσωπεί 160 περιφέρειες από 28 χώρες και μέλη της Ένωσης και όχι μέλη της Ένωσης. Η... Οργα... Οργανώνεται σε ε, έξι γεωγραφικές περιοχές, σε επιτροπές. Η κάθε μία έχει τη δική της δομή και προωθεί σχέδια συνεργασίας μεταξύ των μελών της. Σήμερα έχουμε ανταλλαγή απόψεων για το έργο της οργάνωσης. Ο κύριος Ενερίκο Ρώση είναι εδώ, πρόεδρος της ε, περιφέρειας της Τοσκάνης. Και έχουμε και τον κύριο Πέλκαρσκιντ από τη Βρετάνη ή κάπως έτσι τέλος πάντων είναι τα ονόματα. Σας ευχαριστώ που ήρθατε. Θα σας δώσω το λόγο και στους δύο για μια σύντομη παρέμβαση και θα προσπαθήσω κάπως να περιορίσω το χρόνο αγόρευσης. Σίγουρα θα είναι ενδιαφέροντα αυτά που ήθελα να μας πείτε. Θα ήθελα όμως να έχουμε και λίγο χρόνο για ανταλλαγή απόψεων, να έχουμε και μια συζήτηση με τα μέλη της Επιτροπής ΡΕΚ. Κύριε Ρώση, έχετε το λόγο. Ε, αγαπητοί Πρόεδρε, αγαπητοί Προβουλευτές, κύριε και κύριοι, θα αφήσω τις ε, προσωπικές παρουσιάσεις και του φορέα που εκπροσωπώ. Ήδη κάνατε την παρουσίαση, εσείς άριστα κυρία Πρόεδρε. Εμείς συνεργαζόμαστε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Παρακολουθήσαμε προσεκτικότατα όλο την νομοθεσία για τον κανονισμό για τα ταμεία και για τις επενδύσεις. Υπάρχουν κάποιες προτάσεις δικές μας που συμπεριλήφθησαν στο κείμενο το οποίο ενεκρίθη. Τώρα θέλουμε αναγνώριση των χαρακτηριστικών, των ιδιαιτεροτήτων των περιοχών, των περιφερειών, των μεταβατικών επίσης. Από το 2008 μέχρι τώρα η κρίση οδήγησε σε αναπόφευκτη αύξηση των περιφερειακών διαφορών και παρήγαγε ένα νέο ε, παράδειγμα κέντρου κατά περιφέρειας. Και επιτρέψτε μου να αναφέρω ε, την ε, London School of Economics μελέτη για τη συνέπεια της κρίσης στην κοινωνική συνοχή που ανετέθη αυτή η μελέτη από το Ευρωκοινοβούλιο και την έκτη έκθεση όσον αφορά την συνοχή και είναι προφανές ότι όλες οι πρόσφατες μελέτες και στατιστικές του Ευρωστάτ έχουν δείξει αυτή την αλλαγή. Όλα αυτά θα μας επιτρέψουν και θα μας ευκολύνουν να κάνουμε προβληματισμό. Χρειάζεται ευρωπαϊκή πολιτική συνοχής, χρειάζεται περισσότερο από ποτέ αν δεν θέλουμε να μείνουν πίσω κάποιες περιοχές και να κινδυνεύσουμε να ε, υπονομεύσουμε το ευρωπαϊκό εγχείρημα. Κατά την άποψή μου, ένα από τα σοβαρότερα παράδοξα της πολιτικής συνοχής είναι η παρούσα κατανομή των πόρων που εδράζεται επί δικτών και κριτηρίων που δεν συνδέονται με την κοινωνικονομική πραγματικότητα των περιοχών, αλλά αποκλειστικά στις παραμέτρους του ΑΕΠ της περιοχής, της περιφερειακής, του περιφερειακού ΑΕΠ και η περίοδος αναφοράς που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της κατανομής των θετικών ταμείων δημιουργεί πρόβλημα, εδράζεται επί στατιστικών στοιχείων που είναι απειρχιωμένα πρώτης κρίσης. Ένα παράδειγμα συγκεκριμένο, οι ελληνικές περιοχές να, βλέπουν να μειώνεται κατά 20% το υπόρριο του θετικό ταμείου σε σχέση με τις προηγούμενες περιόδους. Γι' αυτό η κατανομή των πόρων θα πρέπει να εδράζεται επί ευρύτερου φάσματος και επί κριτηρίων ε, εδαφικών και κυρίως επί επικαίρων στατιστικών στοιχείων. Είμαι σίγουρος ότι οι ευρωβουλευτές που εργάστηκαν όσον αφορά το πακέτο συνοχής θα συμφωνούν ότι η κατανομή των διαθεωτικών πόρων είναι καρπός που χρειάζεται επι, επι, γεννήθηκε επιβάσεις ευρύτερη συζητήσεω για τον ευρωπαϊκό προπολογισμό και δυστυχώς δεν είχε άμεσα εμπλακεί σε αυτές τις συζητήσεις το Ευρωκοινοβούλιο. Αντίθετα, αν θέλουμε η πολιτική συνοχής να επιβιώσει, κατά την άποψή μου το Ευρωκοινοβούλιο από τούδε και στο εξή θα πρέπει πάντα να εμπλέκεται σε τέτοιε συζητήσει. Άλλη πτυχή. Οι πόροι για την πολιτική συνοχής διανέμονται βάσει ε, εθνικών κριτηρίων παρόλο που πρόκειται περί περιφερειακών πολιτικών για να διευκολύνουμε πιο πλήρη προβληματισμό για την μέθοδο της κατανομής η οργάνωσή μας δημιούργησε μια ομάδα κρούσης, task force για τους δείκτες. Ποια ήταν η κεντρική ιδέα, να ξεκινήσει ένας προβληματισμός όσον αφορά τη μεθοδολογία διανομής να υπάρχει ανταλλαγή πληροφοριών και γνώσεων μεταξύ των περιφερειών και να προετοιμάσουμε επ' αυτή τη βάση τις προβλέψεις που θα μπορούσαν να είναι χρήσιμες για μια εμβάθυνση της αναλύσεως. Είμαστε στην αρχική φάση των εργασιών, αλλά ήδη βλέπουμε ενδιαφέροντα στοιχεία και με τα χαράς μπορούμε να σας δώσουμε αυτά τα στοιχεία και ε, να μοιραστούμε μαζί σας τα αποτελέσματά μας που πιστεύω ότι θα δημοσιοποιηθούν μέχρι το Δεκέμβριο νεστότος έτους. Οι συνθήκες καθορίζουν ότι στόχος της πολιτικής συνοχής είναι η μείωση των διαφορών όσον αφορά την ανάπτυξη των περιοχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως με την πάρα του χρόνου αυτή η πολιτική έγινε ε, προσπαθεί να μειώσει διαφορά μεταξύ των περιοχών αλλά να πετύχει ταυτόχρονα και τους στόχους στρατηγικής για την Ευρώπη για το 2020. Πιο γενικόλογη δηλαδή προσέγγιση και η μακροοικονομική ρεσιμότητα ε, και η διακυβέρνηση οικονομική της Ένωσης δεν χρησιμοποιούνται πλήρως. Αν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε τις μεγαλύτερες ανάγκες παρεμβάσεων και αυτό ίσως είναι σωστό, τότε θα πρέπει να είμαστε συνεκτικοί και συνεπείς. Θα πρέπει να αυξήσουμε τους πόρους που αφορούν την πολιτική συνοχής και συνεπώς εν γέννη να αυξηθεί ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός να επανεξεταστεί προς τα άνω ευρωπαϊκός προπολογισμός. Πρέπει να το πούμε σαφώς. Η πολιτική συνοχή θα πρέπει να επικεντρωθεί επί της οικονομικής περιφερειακής ανάπτυξης και να μην είναι όμοιρος για να εξασφαλίζει μακροοικονομικές συγκλήσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Διότι εφαρμόζοντας αυτόματα την αρχή της αιρεσιμότητας της μακροοικονομικής κινδυνεύουμε να θέσουμε σε δύσκολη θέση τις, περιοχές, τις περιφέρειες, κυρίως εκεί όπου η συνοχή εξασφαλίζει σχεδόν όλες τις χρηματοδοτήσεις για την ανάπτυξη. Για να επιτρέψουμε λοιπόν μια επικαιροποίηση οικονομική ως πρέπει, θα πρέπει η συγχρηματοδότηση περιφερειακό εθνικό επίπεδο των διαθετικών τομέων να μην εντάσσεται στον υπολογισμό των δεσμεύσεων που τίθεται από το Σύμφωνο Σταθερότητας. Τουλάχιστον αυτό θα πρέπει να ε, επιτραπεί. Εάν επιτραπεί αυτό, η περιοχή μου θα μπορούσε να έχει πρόσθετους πόρους για πράγματα όπως τα 62 εκατομμύρια ευρώ το έτος για την επταετία και 400 εκατομμύρια συνολικά που ε, βεβαίως μπορούμε να τα δαπανίσουμε και θέλουμε να τα δαπανίσουμε για να αυξήσουμε τις επενδύσεις που προβλέπονται όσον αφορά την πολιτική συνοχής για να χρησιμοποιήσουμε τα χρήματα για την επίτευξη των στόχων. Υπενθυμίζω μεταξύ άλλων ότι σαν το Σκάνα, α, στο Σκάνι αλλά όχι μόνο εμείς, 82 εκατομμύρια ευρώ έχουμε προβλέψει σαν πόρους εν αναμονή των ευρωπαϊκών πόρων για την επταετία 2014-2020 που έχουν καθυστερήσει και έχουν καθυστερήσει να εγκριθούν. Αυτό δείχνει πολύ καλά όχι μόνο η τη δική μου περιφέρεια αλλά και πολλές άλλες περιφέρειες ότι είμαστε πεπισμένοι για τη χρησιμότητα της πολιτικής συνοχής. Η περιφερειακή οικονομική ανάπτυξη δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς οι περιφέρειες να είναι στο επίκεντρο της εν λόγω πολιτικής και θα πρέπει να παίξουν σημαντικό ρόλο για την επίτευξη στρατηγικής της Ευρωπαϊκής για το 2020 στις διάφορες ε, περιφέρειες και για τον ορισμό και την εφαρμογή των λειτουργικών προγραμμάτων. Όσον αφορά αυτό, η οργάνωσή μας πάντα πρότεινε ότι πρέπει στις περιφέρειες να δοθεί μεγαλύτερος ρόλος στη διαχείριση και υλοποίηση της πολιτικής συνοχής. Και χάρη στο Ευρωκοινοβούλιο η ενίσχυση των διαφόρων διατάξεων όσον αφορά τη διακυβέρνηση την πολυεπίπεδη και την αρχή της εταιρικής σχέσης έχουν αυτά εισαχθεί και στους διάφορους κανονισμούς που διέπουν τα διευθυντικά ταμεία. Η οργάνωσή μας ε, κάνει μια δημοσκόπηση μεταξύ των περιφερειών για να δούμε πώς μπορούν και να υλοποιούνται αυτοί οι στόχοι και να γίνονται σεβαστές οι αρχές και αυτή τη δειγματοληψία, άμα θέλετε, τη δημοσκόπηση μπορούμε να τη μοιραστούμε μαζί σας και τα συμπεράσματα. Σήμερα βρισκόμαστε στην αρχή της περίοδου προγραμματισμού 2014-2020, αλλά το μέλλον της πολιτικής συνοχής μετά το 2020 ήδη έχει τεθεί επιτάπητος. Πιστεύω ότι ο συνάδελφος Πιέρ Καλσκίντ, αντιπρόεδρος της περιοχής της Βρετάνης και μέλλον του Προεδρείου του φορέου μας μπορεί να αναπτύξει άλλα ενδιαφέροντα σημεία προς προβληματισμό. Σας ευχαριστώ για μια ακόμη φορά που με επιτρέψατε να έρθω να σας μιλήσω. Thank you. Thank you very much. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Κάρλε Κίντ. Καλά το είπα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές. Λέγομαι πια Κάρλε Κίντ, είμαι αντιπρόεδρος της Περιφέρειας Βρετάνης, προσωπώ όπως είπε και ο κύριος Ρώση, την ε, διάσκεψη των παράκτιων περιφερειακών περιοχών ε, σήμερα. Σας ε, μετέφερε κάποια μηνύματα και κάποια ερωτηματικά δικά μας ο κύριος Ρώση. Εγώ από την πλευρά μου θέλω να σας ευχαριστήσω κυρία Πρόεδρε για την υποδοχή που μας επιφυλάξατε στη συνεδρία της Επιτροπής σας, της Επιτροπής Ρέτζη. Θα ήθελα επίσης να σας ευχαριστήσω για τη διάσκεψή μας. Τα τελευταία χρόνια έχει συνεργαστεί με τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Συγκεκριμένε συγκεκριμένα σε διαπραγματεύσεις ε, για το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο και βέβαια και για το νομοθετικό πακέτο της πολιτικής συνοχής. Έχουμε δώσει κοινέ μάχες, το είπε ο κ. Ρώση, παραδείγματο χάρη σε ό,τι αφορά την ε, μεγαλύτερη ευελιξία για τις προτεραιότητε τις επενδυτικέ στο ΕΤΠΑ, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακή Ανάπτυξη. όπως επίσης αναφέρθηκε το όχημα στην μακροαιρεσιμότητα η δύναμη, ισχύ της διάσκεψής μας είναι ότι μπορούμε τις σκέψεις μας, τις απόψεις μας από τις διαφορετικές περιφέρειες να τις διαθρώνουμε σε πολιτικό λόγο. Είμαστε άλλωστε οι άνθρωποι που βρισκόμαστε επί τόπου και θέλουμε να μεταφέρουμε κάποια μηνύματα προς τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και σε εσά μεταξύ άλλων στους Ευρωπαίους βουλευτές. Αν μιλάμε για περιφερειακές πολιτικές, για το μέλλον της περιφερειακής πολιτικής εν γέννη, νομίζω ότι ε, εσείς οι ευρωβουλευτές και τα μέλη της Επιτροπής ε, Ρέτζι είστε οι τύχη, αν θέλετε, που έχουμε, ε, η τύχη να έχουμε σας ως συνομιλητές. Ποια είναι η εμπειρία μας ότι αφορά την υλοποίηση των προγραμμάτων της περίοδου 2014-2020 πριν συμπληρώσω αυτά που είπε ο κύριος ε, Ρώση για το μέλλον της ε, περιφερειακής πολιτικής εξέφρασε κάποια ερωτηματικά, κάποιες ανησυχίες, θα ήθελα να πω δύο λόγια για την εμπειρία των περιφερειών σε ό,τι αφορά την υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων της περίοδου 14-20. Η διάσκεψή μας υιοθέτησε μια πολιτική θέση στις 27 Φεβρουαρίου όταν συνεδρίασε το πολιτικό προεδρείο το πρώτο μήνυμα που θα ήθελα να σας μεταφέρω είναι η πολιτική νομιμοποίηση των περιφερειών. Ουσιαστικά είμαστε μια αρχή διαχείρισης, ή ε, μεσολαβητές, ε, οι εντεταλμένοι ε, για το ρόλο αυτό της διαχείρισης. Είμαστε και εμείς δηλαδή ε, εκλεγμένοι, οι περισσότεροι τουλάχιστον, είμαστε αιρετοί και είμαστε και ένας πολιτικός θεσμός Άρα ουσιαστικά είμαστε ο συνδετικός ε, κρίκος μεταξύ του τεχνικού επίπεδου, του πολιτικού οράματος ε, και της δικής σας, ε, του δικού σας ρόλου που είναι η εφαρμογή των πολιτικών. Καλούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προβεί σε ένα καλύτερο συντονισμό μεταξύ των κανονισμών της πολιτικής συνοχής, των συστάσεων των χωρών, των συμφωνιών εταιρικής σχέσης και των επιχειρησιακών προγραμμάτων. Η ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ Ρέγγιο επίσης πρέπει να παίξει ένα πιο σημαντικό και πιο στρατηγικό ρόλο συντονισμού στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κάποια άλλα ζητήματα τα οποία ετέθησαν, να σας πω ότι έχουμε τονίσει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε για την εκπόνηση αυτών των επιχειρησιακών προγραμμάτων και συγκεκριμένα για να δικαιολογήσουμε την ε, χρηματοδότηση υποδομών με κρίση κλίμακας, παρά το ότι το επιτρέπει το ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο. Είναι πραγματικά παράδοξο και το λέω τα λόγω γνώσεως, γιατί η Βρετάνη, δική μου περιφέρεια, μεταξύ αυτών ε, που επλήγησαν κατά κάποιο τρόπο το ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την ε, ψηφιακή στρατηγική τη βάζει πάνω-πάνω ε, στις προτεραιότητες ενώ εμείς πρέπει να κινήσουμε και ουρανό για να αιτιολογήσουμε τις επενδύσεις που θα πρέπει να γίνουν από το πρόγραμμα ΕΤΠΑ στις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνία και εν γέννη για τις αναπτυγμένες όπως λένε περιφέρειες. Εμείς κινητοποιούμεθα για να καθορίσουμε το μέλλον της πολιτικής συνοχή για την περίοδο μετά το 2020. Στα λίγα λεπτά λοιπόν που μου απομένουν θα ήθελα να σας μεταφέρω κάποια μηνύματα και κάποια ερωτηματικά. Ένα ερωτηματικό. Ποιο είναι ο ρόλος ε, ο δικός μας ε, της πολιτικής, για το μέλλον της περιφερικής πολιτικής. Υπήρξε μεγάλη υποστήριξη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και έτσι σώθηκε ο προπολογισμό τη Περιφερειακή Πολιτική για τα έτη 14-2020. Είναι θετικό αυτό. Πρέπει όμω να έχουμε υπόψη μα ότι είναι πολύ σημαντική αυτή η χρηματοδότηση γιατί τη να σα πω συγκεκριμένα, στο, στην επικράτειά μα. Είδαμε να φτάνουν περίπου 900 εκατομμύρια ευρώ από το Κοινωνικό Ταμείο, από το Ταμείο ανάπτυξη Ανάπτυξης, το Ταμείο για τα για τις θαλάσσιες ε, και βέβαια από το ΕΤΠΑ. 900 εκατομμύρια λοιπόν. 1,4 δις όμως είναι ο ετήσιος προπολογισμό του Περιφερειακού Συμβουλίου της Βρετάνης. Άρα δεν είναι διακοσμητικό ο ρόλο μα. Καταλαβαίνετε ότι είμαστε ένα μοχλό, είμαστε ένα πολύ σημαντικό ε, παράγοντα. Και βέβαια αυτό εντάσσεται και στι αναπτυξιακέ, μακροπρόθεσμε αναπτυξιακέ μα στρατηγικέ είδαμε ότι κάποιες φορές ετέθη το ζήτημα κατά πόσο η πολιτική συνοχή μπαίνει σε ε, δεύτερο ρόλο. Ο κύριος Γιούνκερ λίγο παραπάνω από ένα χρόνο πριν ε, παρουσίασε τις πολιτικές του κατευθύνσεις. Δυστυχώς αυτές δεν αναφέρεται η πολιτική συνοχή. Ούτε η ανάγκη να ενισχυθεί η οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή. Παρότι αναφέρονται ρητός στη συνθήκη της Ένωσης αυτές οι τρεις συνοχές, οικονομική, κοινωνική και εδαφική. Έχει υπαχθεί λοιπόν ε, ε, και υποβαθμιστεί κατά κάποιο τρόπο η περιφερειακή πολιτική, ε, έχει υποτιμηθεί η σημασία, έχει μπει σε δεύτερο πλάνο. Όμως, αν δεν υπάρχει η, η αλληλεγγύη σε επίπεδο οικονομικό, κοινωνικό και περιφερειακό δεν μπορεί να εφαρμοστεί επιτυχημένα με οικονομική πολιτική. Αν αναπτυχθούν δε και οι πιο φτωχές περιφέρειες, θα μπορέσει να δημιουργηθεί μια οικονομική ζώνη που θα ευημερεί περισσότερο, παρότι βλέπουμε περισσότερες ε, ε, διάφορες και το χάσμα να διευρύνεται στην Ευρώπη. Τώρα, η επενδυτική πολιτική βασίζεται στις χρηματοοικονομικές επενδύσεις. Ο κύριος ε, Γιούνκερ πολύ σωστά είπε ότι θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τη μεγάλη έλλειψη επενδύσεων στην Ευρώπη. Θα θέλαμε βέβαια πιο φιλόδοξο το ευρωπαϊκό πρόγραμμα επενδύσεων. Θέλω να συγχαρώ το Κοινοβούλιο και κυρίως τον κύριο Φανίστελ που κατέθεσε την γνωμοδότηση της Επιτροπής ΡΕΚΙ για το σχέδιο κανονισμού. Θέλω να σας ευχαριστήσω λοιπόν. Ε, πιστεύω ότι το σχέδιο Γιούνκερ πρέπει να είναι απλά συμπληρωματικό εργαλείο, όχι να υποκαταστήσει την πολιτική συνοχή. Η Κομισιόν ε, θέλει να ξεκινήσει ξανά την ανάπτυξη με χρηματοπιστωτικά μέσα. Μας ε, Δημιουργεί κάποια ερωτηματικά η επιλογή αυτή. Θα πρέπει να δούμε τι αντίκτυπο θα έχουν αυτά τα μέσα στην περιφερειακή ανάπτυξη και στην οικονομική, κοινωνική, εδαφική συνοχή. Εμεί θα είμαστε πολύ προσεκτικοί, θα παρακολουθούμε και του σύνεγγυ και βέβαια και στη διάθεσή σα ώστε μαζί με εσά στην Επιτροπή Ρέγγι να επιληφθούμε αυτού του ζητήματο και να συνεργαστούμε. Εμεί έχουμε να σα δώσουμε παραδείγματα, που να σα δώσουμε τις ιδέες μας για τη χρήση των χρηματοπιστωτικών αυτών μέσων. Ολοκληρώντα εν συντομία να σας δώσω κάποιες ε, σκέψεις, κάποιες πίστες για το μέλλον της πολιτικής συνοχής. Πιστεύω ότι θα πρέπει να υπερασπιστούμε τα ωφέλη που έφερε η περιφερειακή πολιτική σε όλες τις περιφέρειες της Ένωσης και ως διάσκεψη και ένωση περιφερειών θέλουμε να σας παρουσιάσουμε και να αναπτύξουμε κάποια παραδείγματα ε, και επιτυχημένες ε, περιπτώσεις. Μέχρι το 2016 θα έχουμε δημοσιεύσει ε, κάποια στοιχεία τα οποία πιστεύουμε ότι μπορούν να σας βοηθήσουν για την αναθεώρηση, την ενδιάμεση του δημοσιονομικού πλαισίου. Επίσης πρέπει να σας πω ότι παίζουν πολύ θεμητό ρόλο οι περιφέρειες της πολιτικής συνοχής. Δεν εφαρμόζουμε απλά τα τεχνικά, έχουμε και πολιτικές προτάσεις να διατυπώσουμε για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της πολιτικής αυτής. Τέλος, πιστεύω και το προείπα, η εγκάρσια πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η περιφερικη πολιτική. Θα πρέπει να το λέμε και θα πρέπει να φροντίσουμε να μην υπαχθεί ε, σε άλλες ε, πολιτικές της Ένωσης. Άρα θα πρέπει να διατηρήσει έναν επαρκή προϋπολογισμό. Μίλησα για τα χρηματοπιστωτικά μέσα, δεν επανέρχομαι. Τέλος, Ολοκληρώνω υπενθυμίζοντας ότι η οικονομική, η κοινωνική, εδαφική συνοχή, το εδαφικό κομμάτι, η πτυχή αυτή δεν θα πρέπει να ξεχαστεί. Για μας είναι πολύ σημαντική αυτή η εδαφική διάσταση και ξέρουμε ότι και τα νησιά, οι νησιωτικές περιφέρειες ε, ε, έχουν ε, κάπως μεγαλύτερο εδαφικό κόστος. Αυτά λοιπόν είναι τα μηνύματά μας και σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Thank you. Thank you very much. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη διαφορετική προσέγγιση στην παρουσίασή σας και για τις πολύ ενδιαφέρουσες ερωτήσεις που θέσατε. Τώρα θα γίνει μια συζήτηση με τα μέλη, ίσως λάβουμε και μερικές απαντήσεις, ίσως κάνουμε και μερικές παραπάνω ερωτήσεις. Ο κύριος ε, Ραμανζέ ζήτησε πρώτα στο λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε κύριε Πρόεδρε Ρώση, κύριε Αντιπρόεδρε του Περιφερικού Συμβουλίου της Βρετάνης. Ευχαριστώ όλους σας που θέσατε τις ερωτήσεις της θεμελιώδης όσον αφορά την πολιτική συνοχής. Ερωτήσεις που θέτουμε κι εμείς. Αν μου επιτραπεί χρονικά θα ήθελα να επανέλθω σε κάποια στοιχεία. Όπως ο κύριος Κακασίν ε, και εγώ εκφράζω ανησυχίες Έχουμε ανησυχίε όσον αφορά το μέλλον το ίδιο της περιφερειακής πολιτικής μετά το 2020. Καταρχάς, χαιρετίζω την αποτελεσματική δράση και τη σημαντική συνεισφορά ε, της διάσκεψης ε, των παρακτήων περιφερειακών περιοχών όσον αφορά τη δράση για τις πολιτικές συνοχής. Θα ήθελα να προβώ και σε ένα σχόλιο όσον αφορά τη σημασία της διάσκεψης παρακτήων περιφερειακών περιοχών. Λοιπόν, ο φορέας μας, αυτή η διάσκεψη των παρακτήων περιφερειών και θαλάσσιων περιοχών ε, και εμείς σαν Επιτροπή Ρέζη δεν πρέπει να λησμονούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια θαλάσσια ισχύς, μια θαλάσσια δύναμη και η Ευρώπη είναι η Ήπειρος εκείνη που είναι η πιο αποκομμένη από όλες τις υπήρους του κόσμου με ανοίγματα προς τη θάλασσα ε, πάρα πολύ μεγάλα. Λοιπόν, ξέρουμε το ρόλο που θα παίξουν οι θάλασσες στο μέλλον και οι ωκεανοί. Είναι σημαντικό λοιπόν να έχουμε την υποστήριξη της διάσκεψης των παρακτήων περιφερειακών περιοχών για να κινητοποιούμε ε, την Ευρωπαϊκή Ένωση για να εφαρμόζει μια πραγματική θαλάσσια πολιτική, ωκεανική και λιμενική πολιτική ενοποιημένη. Κάτι εποφελές για όλες τις περιφέρειες της Ευρώπης. Τούτων λεχθέντων. Πράγματι θέσατε θεμελιώδη ερωτήματα. Ίσως όσον αφορά την αποδυνάμωση της περιφερειακής πολιτικής η οποία συνεπάγεται ανησυχίες όσον αφορά και την διόνυση της πολιτικής. Εξεπλάγει, διότι στη συζήτηση ευρωπαϊκό επίπεδο ελάχιστα αναφέρουμε τη γεωργική πολιτική και την πολιτική συνοχής. Θυμάμαι την παρουσίαση που έκανε ο πρόεδρος Γιούνκερ όταν παρουσίασε το πρόγραμμά του στους ευρωβουλευτές πριν αναλάβει τα καθήκοντά του και έπρεπε να ψάξω να βρω γραμμή για την αγροτική πολιτική. Δεν τη βρήκα Και γραμμή όσον αφορά την πολιτική συνοχής ενώ πρόκειται για δύο μεγάλες πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Όσον αφορά την πολιτική συνοχής, είναι η πολιτική της αλληλεγγύης, της σύγκλησης, το θυμήσατε, η αλληλεγγύη αναφέρεται στις συνθήκες. Είναι κάτι που υποχρεώνει ε, να συμμορφωθούν με αυτή την αρχή όλες οι ευρωπαϊκές πολιτικές και εκφράζουμε μια ανησυχία, μάλλον δύο ανησυχίες. Πρώτον, αναφερθήκατε στα χρηματοπιστωτικά μέσα, τα οικονομικά μέσα. Ζητάμε από τις περιφέρειες να αποδείξουν ότι έχουν καλές επιδόσεις. Αντιστρέφουμε δηλαδή το βάρος της απόδειξης και της ενοχής. Αντιμετωπίζουν οι περιφέρειες της Ευρώπης κάποια προβλήματα για να πετύχουν τους στόχους, διότι συνολικά οι ευρωπαϊκές πολιτικές δεν συνδράμουν στην επίτευξη των στόχων και έχουν αρνητικό στόχο όσον αφορά τους τεθέντες στόχους, στόχους συνοχής. Πρέπει να επαγρυπνούμε. Και γι' αυτό συμφωνώ πλήρως με αυτά που είπατε. Χρειάζεται εγκάσια προσέγγιση όσον αφορά τους στόχους της ε, συνοχής στις ευρωπαϊκές πολιτικές. και η Γενική Διεύθυνση Ρίτζιο θα πρέπει να έχει μεγαλύτερο ρόλο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν μπορώ να απαντήσω στι διάφορε συγκεκριμένε ερωτήσει λόγω ελλείψεω χρόνου και μπορώ να πω σε λεπτομέρειε. Να πω δύο λόγια μόνο. Πρώτα απ' όλα το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στατικικών Επενδύσεων. Χθε την Επιτροπή την Οικονομική και την Επιτροπή Προπολογισμών ψηφίσαμε τα αποτελέσματα του τριμερού διαλόγου Το Ευρωκοινοβούλιο στηρίζει τις νέες προσπάθειες που θα επιτρέψουν να κινηθούμε προς την ισορροπία. Εκφράζουμε λύπη όμως διότι δεν έχουν ληφθεί υπόψη γεωγραφικές πτυχές και διατρέχουμε ένα κίνδυνο στον αφορά αυτό το στρατηγικό ταμείο. Θα κινητοποιηθούν στις μεγάλες μητροπόλεις, για τις μεγάλες μητροπόλεις οι πόροι και δεν ξέρω αν το Ταμείο μήπως αποσταθεροποιήσει έτσι περαιτέρω ε, τις προσπάθειες που καταβάλλονται για την επίτευξη των στόχων της συνοχής, αυξάνοντας τις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των περιφερειών, μεταξύ των λιγότερων επιγμένων περιφερειών και των μητροπολιτικών περιφερειών, που αναμφισβήτητα είναι πλέον ανεπτυγμένες. Αναφερθήκατε σε κάτι που πρέπει να μας ανησυχεί στο μέλλον. Πρέπει να προβληματιστούμε για το πλαίσιο μετά το 2020. Πράγματι, σωστά το θέσατε, πρέπει να επανακαθορίσουμε το κέντρο και την περιφέρεια. Πώς ορίζονται αυτά. Εντός Ευρώπης υπάρχουν ζώνες που είναι περιφερειακές ε, όσον αφορά την ανάπτυξη. Πρέπει να τα λάβουμε υπόψη αυτά που είπατε και σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ που υπενθυμίσατε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις διαπραγματεύσεις έκανε ό,τι μπορεί για να απορρίψει τη μακροοικονομική αιρεσιμότητα. Πρέπει να σκεφτούμε τους λόγους για τους οποίους επευλήθη η αιρεσιμότητα στην περιφερειακή πολιτική, η μακροοικονομική αιρεσιμότητα. Θα ήταν ενδιαφέρον να προσμετρήσουμε τη σοβαρότητα αυτού. Θα δράσουμε ήδη από σήμερα για να υπάρξει μεγαλύτερη ευελιξία εν τη εφαρμογή της της αυτής αρχής. Θα είχα κι άλλα να πω, αλλά δυστυχώς εξάντλησα τον χρόνο γόρευσης. Σας ευχαριστώ, κύριος Νοβάκοφ έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η μέχρι τώρα συζήτηση. Επειδή μιλάμε για παράκτης περιφερειακές περιφέρειες, θα ήθελα να σας μεταφέρω την εμπειρία που είχα ως εισηγητής Επιτροπής ΕΚΟΝ για την ειδική έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου για τις εσωτερικές πλωτές οδούς. Συγγνώμη που σας έχω γυρίσει με την πλάτη μου βέβαια, αλλά τι να κάνω. Αυτό το ζήτημα το συζητήσαμε, το ζήτημα των μεταφορών. Οι μεταφορές, υπάρχουν και άλλε παραδοσιακέ δραστηριότητε, αλλά οι μεταφορέ είναι πολύ σημαντική δραστηριότητα, ε, ναυτιλία κτλ. Και πρέπει να πω ότι το σύστημα μεταφορών είναι σπονδυλική στήλη ε, της οικονομίας για τις περιοχές αυτές. Πολλοί ε, είπαν ότι δεν γίνονται επαρκώ επενδύσεις στον τομέα των μεταφορών και ότι δεν είναι τόσο φιλόδοξο το επενδυτικό σχέδιο. Πρέπει να σας πω όμως ότι από το 2006 μέχρι το 2013 πάνω από ένα δις επενδύθηκαν ε, στις περιοχές αυτές για την βελτίωση ε, της εσωτερικής ναυσιπλοείας. Υπάρχουν όμως συμφορήσεις ακόμη, αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα της έλλειψης συντονισμού μεταξύ των περιοχών. Οι οργανώσει λοιπόν σαν τη διάσκεψη αυτή των παράκτων περιφερειακών περιοχών τη Ευρώπη είναι σημαντικέ. Αλλιώ έχουμε να αντιμετωπίσουμε την εξή πρόκληση. Επενδύουμε πολύ σε κάποια συγκεκριμένη περιφέρεια, βελτιώνουμε τις υποδομέ και λίγα χιλιόμετρα πιο πέρα, λίγε εκατοντάδε χιλιόμετρα πιο πέρα, τίποτα. Να σα δώσω λοιπόν το εξή παράδειγμα. Είναι σαν να έχει ένα αεροπλάνο και ένα αεροδρόμιο έχεις, μπορείς να απογειωθείς, αλλά δεν υπάρχει δυνατότητα να προσγειωθείς. Άρα το πρώτο αεροδρόμιο, το οποίο απογειώνεται το είναι άχρηστο τελικά, αφού δεν υπάρχει αεροδρόμιο να προσγειωθεί το αεροπλάνο. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει μια κοινή στρατηγική, μια κοινή προσέγγιση και ένα συντονισμό. Ιδίω όταν μιλάμε για τι ε, υποδομέ στον τομέα των μεταφορών και, και για τα μεταφορικά συστήματα. Φυσικά έχετε το πλεονέκτημα εσείς ότι είστε στις ε, περιφερειακές περιοχές, πρέπει να βελτιώσετε τα λιμάνια και να εστιάσετε εκεί, αν δεν έχουν εστιάσει κάποιες περιφέρειες ακόμη εκεί, γιατί δεν θα πεθάνει ποτέ αυτή η οικονομία. Όλο και περισσότερο θα αυξάνεται η ζήτηση για αυτές τις υπηρεσίες. θα βασιστούν ή βασίζονται σε εσά ή άλλες περιοχές της Ευρώπης. Αυτή είναι η βασιζονται σε εσα η αλλες περιοχες τη ευρωπης αυτη ειναι η αποψη μου. Πρέπει να συνεργαστούμε στενά με οργανωσει όπω αυτή τη διάσκεψη, αλλά απαιτείται και σημαντική προσπάθεια για να βελτιωθεί η έκφραση των πολιτικών συνοχής σε αυτές τις περιοχές. Σας ευχαριστώ πολύ. κυρία Βάν έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Και ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτήν την ε, περιεκτικότατη παρουσίαση της ε, διάσκεψης. Ε, είμαι από την Αυστρία και σίγουρα δεν είμαστε παράκτια περιοχή, είμαστε ορεινή περιοχή, γι' αυτό λοιπόν συγχωρήστε μου την παρέμβαση, αλλά είχα κάποια σχόλια που ήθελα να κάνω και κάποιες ερωτήσεις. Καταρχάς θεωρώ άξιο συγχαρητηρίων το γεγονός ότι δεν περιοριζόμαστε μόνο στις 28 χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά θέλουμε να συμπεριλάβουμε και άλλες χώρες που δεν ανήκουν σε αυτήν. Γιατί η Ευρώπη δεν είναι μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση και πολύ σημαντική λοιπόν είναι η συνεργασία ανάμεσα σε όλους για να λυθούν τα προβλήματα. Κοίταξα τον ιστότοπό σας και μπορώ να πω πως είναι πάρα πολύ ενημερωτικός και βρίσκω τις αρμοδιότητες αρκετά μεγάλες. Υπάρχει η αδερφική συνοχή και η φροντίδα για το, την επίτευξη του, του, κυρίου, ε, του κυρίου στόχου που είναι η ε, χωρίς αποκλεισμούς Ευρώπη. Ε, να σας πω ότι εντόπισα τρία πάρα, πολλά, τρία πάρα πολύ σημαντικά σημεία. Η γεωργία, η βιώσιμη ανάπτυξη και οι ε, τεχνολογικές εξελίξεις. Δεν βρήκα όμως κάποια αναφορά στα κοινωνικά ζητήματα, δηλαδή στην εκπαίδευση, στην, ε, στις θέσεις απασχόλησης, στις περιφέρειες και πιστεύω πως είναι εξίσου σημαντικά ζητήματα με τα υπόλοιπα, ιδιαίτερα έχοντας ε, κατά νου τους στόχους της Ευρώπης 2020 που είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι με τους στόχους της ε, πολιτικής συνοχής. Η απασχόληση, η εκπαίδευση, η ε, μείωση του αριθμού των ε, μαθητών που διακόπτουν το σχολείο, η εξάλληψη και η μείωση σε αρχικότερο στάδιο της φτώχεια. Είναι πάρα πολύ σημαντικά θέματα και θα με ενδιαφέρε λοιπόν να μάθω τι σκοπεύετε να κάνετε για αυτά. Σας ευχαριστώ πολύ, ο κύριος Όλμπριχτ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. δεν ε, εξεπλάγει από την ποιότητα της παρουσίασής σας. Έχετε εμπειρία πάρα πολλών ετών και είδα ότι δεν ε, ασκείτε μόνο πίεση και προσπαθείτε να ε, υπερασπιστείτε συγκεκριμένες περιοχές, αλλά κύριο μέλημά σας είναι η προώθηση όλης της ε, πολιτική συνοχής και όλων των περιφερειών. Αυτή η ομάδα προβληματισμού είναι κάτι καινούργιο το οποίο καλωσορίζω. Είναι ένα αρκετά πολιτικό, πολιτικού χαρακτήρα σώμα το οποίο έχει και πολύ ε, έντονη δυνατότητα να επηρεάσει τις ε, πολιτικές εξελίξεις. Πιστεύω πως θα έπρεπε στην Επιτροπή μας να καλέσουμε τους ε, σημαντικούς φορείς στον κλάδο αυτό που μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Γι' αυτό λοιπόν είναι και πολύ σημαντικό να κοιτάξουμε την ε, μελέτη. Υπάρχουν κάποια στοιχεία της ε, μελέτης που αφορούν την ε, εποχή πριν τον κανονισμό. Για παράδειγμα, το, το ΑΕΠ. Αυτό δεν είναι κάτι καινούριο, το γνωρίζαμε από πριν. Έχουμε την αρχή της σύνδεσης με το ΑΕΠ και ποια θα είναι λοιπόν η συνέπεια της αποσύνδεσης αυτής είναι η ερώτησή μου. Διότι το ΕΠ δεν είναι καλός δείκτης σε όλες τις περιπτώσεις. Εσείς πιστεύετε πως αν αλλάξει αυτή η σύνδεση θα, αλλάξει και, θα αλλάξουν και τα δεδομένα. Είναι όπως η μακροοικονομία, είναι τεράστιος κλάδος. Σε κάποια κρατημέλη υπάρχουν στοιχεία που μας δείχνουν ότι υπάρχει σταθερότητα και σε άλλες περιπτώσεις δεν βοηθάνε αυτοί οι δείκτες. Και πιστεύω πως όταν αναφέρουμε αυτούς τους σημαντικούς παράγοντες στο, στο έργο μας, θα πρέπει να εντοπίσουμε και το χρονικό διάστημα στο οποίο θα δραστηριοποιούνται. Και για μένα αυτό το χρονικό διάστημα είναι το τώρα, το παρόν. Διότι αυτά που συζητάμε είναι τώρα σχετικά, δεν θα είναι ίσως σε έξι μήνες. Εσείς λοιπόν θεωρείτε πως είναι σωστό αυτό, πως είναι κάτι που καλώς χρησιμοποιούμε στις μακροπεριφέρειες. Αυτή ήταν η ερώτησή μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και ελπίζω να έχουμε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ανταλλαγή απόψεων και απαντήσεις σας να είναι ε, εξίσου ενδιαφέρουσες και κυρίως επίκαιρες. Να αναφέρονται στο παρόν. Και με την άποψή σας για το ότι υπάρχει ασάφεια στην πολιτική συνοχή σε αυτή τη στιγμή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Κρέσνο. Μπρέσο. Ευχαριστώ. Ζητώ συγγνώμη που κατέφθασα μόλις τώρα στο τέλος των παρουσιάσεών σας. Όμως σας καλωσορίζω κι εγώ. Εκτιμούμε όλοι μας το σημαντικότατο έργο σας που αφορά τα θέματα που μας απασχολούν και μας στην Επιτροπή μας. Δράτω με τις ευκαιρίες της παρουσίας σας για να επισημάνω ότι δημιουργήσαμε διακομματική ομάδα με πολλά μέλη αυτής της Επιτροπής για την ύπεθρο, τις ορεινές περιοχές και τις υπερπεριφερειακές περιοχές. Οπότε η συνεισφορά σας θα μπορούσε να είναι σημαντική. Ερχόμενοι τώρα σε κάποια θέματα που με ενδιαφέρουν, επισημαίνω το, τη δουλειά που κάναμε από τη μια και από την άλλη θέλω και την άποψή σα. Πιστεύω ότι χάρη όλος ιδιαίτερος το έργο αυτής της Επιτροπής όσον αφορά το σχέδιο Juncker θα καταλήξει ελπίζουμε καλά ο τριμερής διάλογος αλλά χάρη στη δουλειά που κάναμε υπάρχει θέση του Κοινοβουλίου που υπογραμμίζει την ανάγκη να εγγυηθούμε πολιτικές συνοχής εδαφικές στις επιλογές που θα γίνουν όχι μία συγκέντρωση δηλαδή αλλά μία επαρκής εφαρμογή της αρχής της εδαφικής προσεγγίσεως και να βγάλουμε από το σύμφωνο σταθερότητας όχι μόνο που, τους πόρους που οι χώρες ενδεχομένως θα, θα διέθεταν στο αρχικό σχέδιο αλλά πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και εθνικές προσπάθειες, περιφερειακές, τοπικές προσπάθειες. Άρα θέλουμε να υπάρχει δυνατότητα οι περιφέρειες να συμμετέχουν πλήρως μέσω της χρήσης της πολιτικής συνοχής σε έργα ευρύτερα που αφορούν το σχέδιο Juncker. Και η πρόσθετη πόροι εδαφική κρατική να είναι εκτός του συμφώνου σταθερότητας. Θα δούμε που θα καταλήξει ο τριμερής διάλογος βέβαια που δεν έχει ολοκληρωθεί. Τα αποτελέσματα χάρη στη δράση της Επιτροπής μας και του Κοινοβουλίου τα αποτελέσματα που πετύχαμε είναι σημαντικά. Ποια είναι η απόψή σας όσον αφορά το συντονισμό περιφερειακών πολιτικών και σχεδίου Juncker θέλουμε να είναι η απαρχή με καλύτερης πολιτικής επενδυτικής ευρωπαϊκό επίπεδο, να είναι κάτι περαστικό. Χρειάζεται συντονισμός με την περιφερειακή πολιτική, που είναι και σημαντικότερη επενδυτική πολιτική σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και θέλουμε αυτή να γίνεται όλο και πιο αναγκαία. Και να γίνει και προπτική για την επόμενη φάση, μετά το 2020 για το μελλοντικό προγραμματισμό της περιφερειακής πολιτικής και των γενικών στρατηγικών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Ή, ζητώ συγγνώμη, ίσως ήδη να είπατε κάτι όταν πήρατε το λόγο, όμως θα με ενδιέφερε να γνωρίζω ποια είναι η θέση σας όσον αφορά αυτά τα θέματα και σας ευχαριστώ. Thank you very much, Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Καλώ ήρθατε και από μένα και ευχαριστώ πολύ για τι ε, παρουσιάσει σα. Κάνατε λόγο για το μέλλον της πολιτικής συνοχή και σίγουρα συμφωνείτε φαντάζομαι ότι η πολιτική συνοχή θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο στο μέλλον μόνο εάν ε, γίνει σωστή εφαρμογή στο παρόν και μόνο εάν επιτύχουμε τους ε, στόχους που ορίζουν τα διάφορα ε, έγγραφα στρατηγικής. Επίσης βρήκα πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό που είπατε σχετικά με την ε, εφαρμογή και πώς αντιμετωπίζετε πολλές δυσκολίες σε αυτόν τον τομέα. Συγκεκριμένα αναφέρατε τις, τα προγράμματα υποδομής μικρής κλίμακας και πώς αντιμετωπίσατε πάρα πολλές δυσκολίες σχετικά με την εφαρμογή και υλοποίηση κάποιων άλλων διαδικασιών εκεί, όπως για παράδειγμα οι δημόσιες ε, ε, συμβάσεις, ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι κανόνες για, την κρατική, για τις κρατικές ενισχύσεις κτλ. Είναι πολύ χρήσιμα όλα αυτά και για εμάς, εκτός από ενδιαφέροντα, διότι είναι πολύ σημαντικό να δούμε πώς μπορούμε να απλοποιήσουμε τη διαδικασία και να επιταχύνουμε με αυτό την ε, υλοποίηση των ε, προγραμμάτων. Επίσης μας είπατε ότι έχετε πάρα πολλές ε, προτάσεις για τη βελτίωση της αποδοτικότητας των πολιτικών. Υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα παραδείγματα τα οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Σας ευχαριστώ. Αυτές λοιπόν ήταν οι ερωτήσεις από τα μέλη της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης. Ε, κύριε Ρώση, ίσως θα θέλατε να απαντήσετε πρώτος ή να μας κάνετε κάποια σχόλια. Ε, γρήγορα παρακαλώ, σύντομα. Να σας ευχαριστήσω για την προσοχή σας πρώτα απ' όλα και πώς ελήφθησαν υπόψη οι προτάσεις μας με διαθεσιμότητα, ανοιχτό πνεύμα. Συμφωνώ πλήρως με αυτά που υπόθηκαν από πλευράς αντιπροέδρου του κ. Μαζέ που πιστεύω ότι αναφέρθηκε σε περιεχόμενο με το οποίο συμφωνώ απόλυτα. Αναφέρθηκε στην ιδέα της Ευρώπης σαν θαλάσσια δύναμη και γι' αυτό ενωθήκαμε και εμείς στα πλαίσια του φορέα μας της διάσκεψης παράκτης περιφερειακές περιοχές. Όπως είπαν και άλλοι βουλευτές, σημαντικό να υπογραμμίσουμε την ανάγκη διασύνδεσης καλύτερης. Ε, και θα πρέπει να υπάρχει διασύνδεση καλύτερη μεταξύ του Κοινοβουλίου και των Περιφερειών θα μπορούμε να προβλέψουμε νέες πολιτικές συνοχής έτσι. Και θα πρέπει έτσι με, στη συζήτησή μας να ξεφεύγουμε από τα εθνικά συμφέροντα. Και αυτό το χρειάζεται η Ευρώπη. Από αυτή την άποψη και όσον αφορά τις κατευθύνσεις για τις νέες πολιτικές συνοχής, να σημειώσω ότι είμαστε πεπισμένοι ότι χρειάζεται θεματολόγιο αστικό. Προσανατολισμοί, κατευθυντήριες γραμμές, ιδέες που μετά θα χρησιμεύσουν για τον προγραμματισμό της χρηματοδότησης των Ευρωπαϊκών Ταμείων για την πολιτική συνοχής. Πρέπει να προσέξουμε όμως μη δημιουργήσουμε καινούριο διαχωρισμό μεταξύ πολιτικών για τις αστικές περιοχές και των πολιτικών για την Ήπεθρο. Διότι εκεί κινδυνεύουμε Δηλαδή η ιδέα μιας πολιτικής συνοχής που προσπαθεί να επανασυσορροπήσει τις περιφέρειες ίσως να γίνει άλλη μια πληγή. Καλό το θεματολόγιο το αστικό για να δώσει κατευθυντήριες γραμμές για τις αστικές περιοχές αλλά θα πρέπει να συνδυαστεί με το προ θεματολόγιο την Ήπεθρο το θεματολόγιο για τα πιο ισχυρά κέντρα να ταιριάξει με ε, τα θεματολόγια για τις πιο ασθενείς περιοχές. Αυτά είναι απαραίτητα ανοιχτούν υπόψη για την ανάπτυξη. Εν αυτή τη ενία είναι θεμελιώδος και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Ετέθησαν ερωτήσεις σχετικά με τις κοινωνικές πτυχές. Χρησιμοποιούμε καλά το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και αυτό δυστυχώς έχει φορτωθεί όμως υπερβολικά. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ασχολείται με παρεμβάσεις για τη στήριξη της, κατά της φτώχειας, παρεμβάσεις για την κατάρτιση, παρεμβάσεις για την επανεκπαίδευση των ανέργων και εκείνων που προσπαθούν να βρουν εργασία. Για μία ακόμη φορά ε, έχει βαρυνθεί πολύ αυτό το ταμείο από διάφορες ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί και λόγω της κρίσης που μας υποχρεώνει να αντιμετωπίζουμε περισσότερα προβλήματα που αφορούν τους πολίτες της Ευρώπης. Οι πολιτικές, οι σχετικές με το σχέδιο Juncker, όσον αφορά τις περιφέρειες, είμαστε στη διάθεσή σας, πάντα το είπαμε αυτό, είμαστε στη διάθεσή σας για συντονισμό. Μπορούμε να θέσουμε στη διάθεσή σας να συντονίσουμε και τα προγράμματα που θα εγκριθούν από το σχέδιο Juncker. Υπάρχει ένα όριο όμως που εφήγει από το βουλευτή Νόβακ να, να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και πώς για τις υποδομές, κυρίως τις βασικές υποδομές. Το σχέδιο Juncker κατευθύνεται πάνω απ' όλα στις μεγάλες παρεμβάσεις όσον αφορά τις υποδομές. Και αυτή η μεγάλη κλίμακα αν δεν διορθωθεί θα δώσει ένα ρόλο παρέμβασης στις περιφέρειες ε, εάν δεν δοθεί δυνατότητα να παρέμβουμε θα μειωθεί η, δυνατότητα ολοκλήρωσης όσον αφορά και τη συνδυασμού του σχεδίου Juncker με, τα, με, τις, με τους πόρους. Σας ευχαριστώ για μια ακόμη φορά. Ελπίζω να έχουμε και άλλες ευκαιρίες να συζητήσουμε ε, όπως η ευκαιρία που μας δώσατε σήμερα το πρωί να συζητήσουμε τα θέματα αυτά. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή σας, λέει η Πρόεδρος. Χρειάστηκε μήνες να το διοργανώσουμε αυτό. Λυπούμε. Χαίρομαι όμως, διότι ήταν πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Και ελπίζω να συνεχίσουμε και στο μέλλον τη συνεργασία μας και να ανταλλάξουμε εκ νέου απόψεις στην Επιτροπή Ρέτζι. Χαίρομαι επίση, διότι σήμερα έχουμε ένα πάνελ που θα συζητήσει πολύ ενδιαφέροντα σχετικά θέματα, συναφή θέματα. Έχουμε τώρα την παρουσίαση μελέτης για τη στρατηγική συνοχή. Διαδικαστικό μπορώ να θίξω. Εντάξει αν συμφωνείτε. Μα τελειώνει ο χρόνος. Και ο κύριος Ρούας έχει σχέδιο εκθέσεως που πρέπει να παρουσιάσει. Ίσως μπορούμε να ανταλλάξουμε το σημείο 6 με το 7 της ημέρης διάταξης. Πρώτα την έκθεση Ρούας να συζητήσουμε για να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε αυτό, διότι περνά γρήγορα χρόνος με την έκθεση. Περιμένετε λιγουλάκι, ακούστε με. Τι είχα να προτείνω. Να γίνει η παρουσίαση της μελέτης που σχετίζεται με την έκθεση Ρούρας, να μην συζητηθεί γίνει συζήτηση μετά την παρουσίαση της μελέτης, να ακούσουμε τον κύριο Ρούρας και να γίνει κοινή συζήτηση. Έτσι θα έχουμε δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε κάποιες πληροφορίες της μελέτης και την παρουσία του κυρία Ρουάς. Αυτό προτείνω. Ο καθηγητής John Butler και ο κύριος Στίβεν Καν αν έχουν την καλοσύνη να κάνουν σύντομες ε, παρουσιάσεις. Σύντομες, περιορισμένες. Χρόνου φίδου με άλλα λόγια. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και συγκεκριμένα μέλη Καλημέρα. Εκτιμούμε τη δυνατότητα που μας δίνεται να παρουσιάσουμε τη μελέτη μας. Έχουμε πλήρη επίγνωση όμως των χρονικών περιθωρίων. Ποιο είναι το πλαίσιο της μελέτης μας. Η φιλοδοξία για πιο στρατηγική συνοχή τη εφαρμογή των πολιτικών συνοχής και των παρεμβάσεων στην περίοδο 2014-2020 τονίζεται κάτι και στην έκθεση του εισηγητού που θα παρουσιαστεί στο επόμενο σημείο. Πιο συγκεκριμένα, στόχος μας οι συμφωνίε ανάπτυξη και εταιρική σχέσης στα επιχειρησιακά προγράμματα να συντονίζονται καλύτερα, να είναι πιο συνεκτικά, πιο ολοκληρωμένα. Καλύτερε ευθυγραμμίσει απαιτούνται με του στόχου τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω και τι στρατηγικέ και διαδικασίε διακυβέρνηση. Θέλουμε εναρμόνιση όσον αφορά τι προσεγγίσει των διαφόρων πολιτικών να εκμεταλλευτούμε τις συνέργειες όσον αφορά την χρήση των χρημάτων της Ευρωπαϊκής Βασικό θέμα της μελέτης και ερώτημα. Σε ποιο βάθμο έχει συμβεί αυτό μέχρι τούδε όσον αφορά τον προγραμματισμό των παρεμβάσεων για τη νέα περίοδο. Yes, thank you, John. Um... Ευχαριστώ, John. Θα είμαι λακωνικός να εστιαστώ επί των σημαντικότερων πορισμάτων. Τι κάναμε? Μεθοδολογία. Τα θεμελιώδη στοιχεία της μελέτης. Άνωθεν η προσέγγιση. Και μετά εξετάζουμε τις συγκεντρώσεις και το πέσιο εφαρμογή. Ο Τζον μετά θα καταλήξει σε συμπεράσματα και συστάσεις. Δεν, δεν, δεν λειτουργεί. Α, εξετάσαμε 11 κράτη-μέλη. Θέλαμε αντιπροσωπευτικότητα όσον αφορά τα συστήματα διοίκησης. Κεντρική διοίκηση, αποκεντρωμένα συστήματα, ομοσπονδιακά, ε, λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, πιο ανεπτυγμένες, μεταβατικές. Τι γίνεται κατακεφαλή, ε, το κατακεφαλή εισόδημα. Ήδη προγραμμάτων, εθνικά, περιφερειακά, αυτόματα και δομές των επιχειρησιακών προγραμμάτων και αν υπήρχε δυνατότητα πολυχρηματοδότησης στα επιχειρησιακά προγράμματα ή μοναδική πηγή χρηματοδότησης. The first, first Πρώτη διάσταση. Επίπεδο Ευρωπαϊκής Ενώσεως, στρατηγικά πλαίσια από τι κρατήσει γραμμέ τη κοινότητα σε στατηγικό πλαίσιο, κοινό στατηγικό πλαίσιο. Ποιο δεσμευτικό είναι αυτό. Διότι αφορά τον κανονισμό για τι κοινέ διατάξεις. Εκτός να καλύψει τα ταμεία συνοχής διαστατικά, καλύπτονται και η ανάπτυξη υπαίθρου και η αλληλεία. Εστιαζόμεθα επί διασυνδέσεων και προτεραιοτήτων για να υπάρχουν συνέργειες. Συμπληρωματικότητα. μεταξύ πόρων και πέραν αυτών που να καλύπτονται και άλλες ευρωπαϊκές πολιτικές πέρα από τα στρατηγικά πλαίσια. Τα κράτη-μέλη καλωσόρισαν το κοινό στρατηγικό πλαίσιο. Αλλά δεν είχε πρακτικές συνέπειες όσον αφορά τον προγραμματισμό όσο θα θέλαν. Είχα, υπήρχαν τεχνικές διευθετήσεις για την πολιτική συνοχή σε συνάρτηση με άλλες πολιτικές. Όμως ήταν πιο χρήσιμο α, από ότι τα παλιά προγράμματα. At the national level... Σε εθνικό επίπεδο κινηθήκαμε προς τις ε, συμφωνίες εταιρικής σχέσης. Βγήκαμε το πλαίσιο το στρατηγικό. Υπήρχε διαφορά στον αυτά τις εμπειρίες διάφορα πλαίσια συντονισμού. Όσον αφορά τον έλεγχο μέσω συμβάσεων, άτυπος τρόπος ελέγχου μέσω δικτύων, μέσω ανταλλαγής εμπειριών κλπ. Η αρχή της εταιρικής σχέσης εφαρμόστηκε εν γέννη ευρέως. Διάφορες μορφές χρησιμοποιήθηκαν, διάφορα εργαλεία, σε διάφορα επίπεδα διακυβέρνησης από εθνικό σε τοπικό και περιφερειακό. Όπως προανέφερα, συστάσεις κατά χώρα είχα περιορισμένο ρόλο στα πλαίσια. Θεματική συγκέντρωση. Από προσημειώσεις της Λισαβόνας στους στόχους Ευρώπη 2020. Ναι, βασικές αλλαγές. Λόγω χρόνου δεν θα μπω σε λεπτομέρειες. Ξέρετε τα θέματα αυτά. Η εμπειρία των κρατών μελών ανάμεικτες εμπειρίες. Εν γέννη υπήρχε συμφωνία ότι χρειάζεται προστασία και συγκέντρωση των πόρων. Έλλειψη ευελιξίας διαπιστώθηκε όμως. Εφάρμοσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την αρχή θεματικής συγκέντρωσης αυστηρότατα. Ανησυχίες εκφράστηκαν λόγω των εγχωρίων προτεραιοτήτων που στήριξαν οι χώρες και ειδικοί κανόνες προστασίας. 5% για μέτρα αστική ανάπτυξης Φερρυπίν. Η ελάχιστο μερίδιο του EFSF σε εθνικό επίπεδο δεν θεωρήθηκαν ότι ήταν κάτι υποφελές. Υπήρξαν ανησυχίε για την κατανομή των πόρων και κατά πόσο θα απορροφηθούν. Η θεματική συγκέντρωση επετεύχθη σε επίπεδα προγραμμάτων. Πρέπει να δούμε την τελική κατάληψη τα μέτρα για χαμηλή εκπομπή ανθρακοσφαιρυπίν. Δεν ξέρουμε κατά πόσο προωθηθηκαν οι πόροι και αποτελεσματικότητα. Ο τρόπο κατανομη των πόρων είναι αποτελεσματικότερο. Τελευταίο επίπεδο, η τέταρτη διάσταση, η εφαρμογή των πολιτικών στα κράτη-μέλη και οι κανόνες που θεσπίζονται από το CPR ειδώθηκαν θετικά καλό βήμα προόδου, αλλά όχι αρκε... επαρκές. Διότι υπάρχουν κανονισμοί για κάθε πόρο, κυρίως για την άπτυξη υπαίθρου, και ο στόχος της απλούστευσης δεν έχει επιτευχθεί. Απλουστεύονται τελικά τα πράγματα ή περιπλέκονται είναι η ερώτηση. Άρα η αρχιτεκτονική των προγραμμάτων. Λόγω του διαφορετικού πλαισίου. Καλύτερο θεσμικός Συντονισμός υπάρχει. Και λόγω των συμφωνιών εταιρικών σχέσεων. Υπάρχουν επιχειρησιακά προγράμματα που χρησιμοποιούν πολλαπλούς πόρους και διευκόλυνση λόγω των κανονισμών. Η χρήση αυτών όμως ποικίλει από χώρα σε χώρα. Κάποιες χώρες χρησιμοποίησαν τις ευκαιρίες που δημιουργήθηκαν, άλλες χώρες ανησύχησαν για τις συνέπειες και χρησιμοποίησαν ολοκληρωμένη ε, δαφική ε, προσέγγιση είναι κάτι καλό για συνοχή σε τοπικό επίπεδο. Η απορρόφηση όμως και η χρήση ποικίλει από χώρα σε χώρα. Δεν χρησιμοποιήθηκαν οι προσφερθείς δυνατότητες από όλες τις χώρες. Διοικητικό δυναμικό. Καλά πηγαίνουν τα πράγματα σε εθνικό επίπεδο. Σημαντικότερες ανησυχίες είναι οι κρατικές συμβάσεις και οι κρατικές ενισχύσεις. Αφορούν τους φορείς σε χαμηλό επίπεδο, όχι όσον αφορά τους μεγάλους φορείς. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, παίζει θετικό ρόλο για θετική συνοχή, αλλά ακολουθείται το τομεακή προσέγγιση στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω διαφόρων γενικών διευθύνσεων και έτσι περιπλέκονται τα πράγματα. Υπάρχει ανησυχία για τον καλύτερο εσωτερικό συντονισμό σε επίπεδο 100 μελών. Υπήρχε έλλειψη συνοχής όσον αφορά την προσέγγιση που ακολούθησαν οι διάφορες γενικές διευθύνσεις της διαπραγματεύσεις. Τέλος, στα συμπεράσματα, συναθρίζοντας λοιπόν τα πορίσματα. Πρώτον, το νέο πλαίσιο, η νέα προσέγγιση μέσω πλαισίου καθορίζει σαφώς τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θετικό το συμπέρασμα, δημιουργείται σφαιρική στρατηγική προσέγγιση και δήλωση όσον αφορά το πώς εντάσσεται η πολιτική συνοχή σε σχέση με τους γενικούς στόχους, θεματική συγκέντρωση, Υπάρχει ανησυχία από τα κάτι μέλη όσον αφορά το πώς ανταποκρίνεται τις αναπτυξιακέ ανάγκε και προκλήσει σε κάθε χώρα και περιφέρεια. Έδωσε αποτελέσματα η προσέγγιση, θεματική. Άλλαξαν οι δαπάνε στο επίπεδο προγραμματισμού τουλάχιστον το βασικό ερώτημα είναι αν αυτό τελικά θα εφαρμοστεί και στην πράξη. Θα υπάρξουν ζητήματα απορρόφησης, μακροπρόθεσμο θέμα. Τι θα γίνει μετά το 2020 με άλλα λόγια σταδιακή μεταρρύθμιση, μεταμόρφωση της ε, πολιτικής συνοχής σε πιο θεματική πολιτική και πώς αστιάζεται επί εδαφικών διαστάσεων, τοπικών διαστάσεων. Υπάρχει μεταξύ, μεγαλύτερη στρατηγική ολοκλήρωση για τη διαχείριση των πόρων. Αυτό θα ξεπεράσει το στάδιο προγραμματισμού. Θα μπορούσαμε να πούμε όμως ότι οι δημιουργηθήσεις δομές σε κάποια κράτη-μέλη αντιπροσωπεύουν μία προσπάθεια και δέσμευση για πιο συνεκτικό και συντονισμένο προγραμματισμό και προσέγγιση. Τέλος, υπάρχουν ελάχιστα σημάδια απλούστευσης. Θα το ξέρετε αυτό ήδη. Υπάρχουν στοιχεία απλούστευσης σε επίπεδο δικαιούχων, αλλά όχι εντός της εφαρμογή και του συστήματος εφαρμογής. Τέλος, η τελευταία διαφάνεια αφορά τις συστάσεις. Καταρχάς, προσβλέπουμε στην επόμενη φάση. Χρειάζεται πιο συνεργατική προσέγγιση μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κατών και Κοινοβουλίου στην κατάρτιση του στρατηγικού πλαισίου και των εγγράφων τοποθέτησης. Θα ήταν καλό αυτό για τα κράτη-μέλη. Αρχικά σχέδια από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κρατών μελών ήταν η μεγαλύτερη συνεργασία όσον αφορά τα έγγραφα θέσει Και την ετοιμασία τη ανάρξη τη νέα προγραμματική περίοδου, αυτό θα ήταν υποφελέ για στρατηγικό σχεδιασμό. Συντονισμό βελτιώθηκε σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όμω μπορούν να γίνουν περισσότερα. Κυρίω σε επίπεδο κρατών μελών. Συντονισμό μεταξύ DG Regio και Γενική Διευθύνσεω απασχόλησης βελτιώθηκε μεν, χρειάζεται όμως περισσότερο συντονισμός, κυρίως με την Άγκρη και τη Μάρε. Τέλος, μας ζητήθηκαν κάποιες συστάσεις για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θεωρούμε ότι κατά πόσο υποχρεώσεις θα υλοποιηθούν. Αυτό είναι, πρέπει να εξεταστεί περισσότερο. Από την Επιτροπή σας συστήνουμε μεγαλύτερο συντονισμό υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και χρειάζεται και καλύτερο συντονισμό στο Κοινοβούλιο μεταξύ Επιτροπών του Κοινοβουλίου. Έτσι θα επιτυγχάνεται στατική συνοχή όσον αφορά τα διάφορα ταμεία. Ευχαριστώ. Thank you, thank you very much for this. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη σύντομη και πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση η οποία και προέκυψε μετά από αίτημα της δικής μας Επιτροπής, που εκκρεμεί από πέρυσι τον Απρίλιο. Θέλαμε λοιπόν από τότε να έχουμε μια τέτοια μελέτη όπως αυτή και το τελευταίο Νοέμβρη η Επιτροπή μας ε, θέλησε να στέξει μια έκθεση δίας ε, πρωτοβουλίας για την ε, πολιτική συνοχή και συνδυάστηκε αυτό και με την ενδιάμεση αναθεώρηση της Στρατηγικής Ευρώπης 2020. Τον Μάρτιο ο κύριος Ρούας μας παρουσίασε τα βασικά σημεία της έκθεσης του και σήμερα θα ακούσουμε την, ε, το ίδιο το σχέδιο έκθεσης. Σε προθεσμία υποβολής τροπολογιών 2 Ιουλίου, ψηφοφορία στην Επιτροπή στις 17 Σεπτεμβρίου. Κύριε Ρούας, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Θα ήθελα να αρχίσω με τις ευχαριστίες μου προς εσάς και τους συναδέλφους που ζήτησαν να επιταχύνουμε λίγο τις εργασίες μας ε, σήμερα. Δυστυχώς όλοι έχουμε πτήσεις που, μας περιμένουν, που δεν θα μας περιμένουν. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω τους καθηγητές για την αμελέτη που παρουσίασαν, διότι πραγματικά δημιούργησαν ένα πλαίσιο ε, για να παρουσιάσω την έκθεση που θα ακούσετε Μόλις τώρα. Αναθεώρηση λοιπόν της στρατηγική Ευρώπη 2020 και πολιτική συνοχή. Είναι η δεύτερη ανταλλαγή απόψεων που ε, διεξάγεται για αυτό το θέμα. Και θα ήθελα να επαναλάβω τα όσα είπα και κατά την πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Προσπαθώ να συμπεριλάβω τα αποτελέσματα της ε, συζήτησής μας στην έκθεσή, στην μου. Άκουσα με μεγάλη προσοχή όλους τους ε, σκιώδεις και όλους ε, τους ευρωβουλευτές που τοποθετήθηκαν για το θέμα. Συμπερίλαβα λοιπόν όλες τις απόψεις και πραγματικά έχουμε τώρα ένα σχέδιο έκθεσης. Ε, με μεγάλη μου χαρά θα διαβάσω τις τροπολογίες σας, οι οποίες είμαι σίγουρος θα είναι πολύ επικοδομητικές και στόχος είναι να δημιουργήσουμε μια έκθεση η οποία θα καλύπτει όσο το δυνατόν περισσότερα σημεία και περισσότερε πτυχέ τη πολιτική συνοχή και τη αναθεώρηση τη στρατηγική 2020. Είμαι σίγουρος ότι έτσι θα συνεισφέρουμε στην ενδυνάμωση ε, της ε, συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα θα ήθελα να αναφερθώ και στο περιεχόμενο. Από, ότι, από όσο ξέρετε υπάρχει και ένα όριο το μήκος της έκθεσης. Το Μάρτιο εξέφρασα τις ε, βασικές μου ιδέες και έγραψε λοιπόν το σχέδιο έκθεσης και αφού άκουσα τις ε, προτάσεις και τις ιδέες όλων των, εισηγητών, ε, των σχεδόν εισηγητών και των συναδέλφων προσπάθησα να τις συνοψίσω λοιπόν και να τις περιλάβω στο σχέδιο έκθεσης που έχετε ενώπιόν σας. Για παράδειγμα, ασχολούμαι με την σημασία της επεξεργασίας της στρατηγικής σε Ευρώπη 2020 και την ε, ανάλυση των συνεργειών ανάμεσα σε αυτήν και στην ε, πολιτική συνοχή. Επίσης, ε, την σημασία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και τα κίνητρα που χρειάζονται για μια βιώσιμη ανάπτυξη. Περαιτέρω απόψεις που ακούστηκαν την προηγούμενη φορά είναι η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, η ε, πολυεπίπεδη λοιπόν διοίκηση που όμως δεν πρέπει να οδηγήσει σε αύξηση της ε, γραφειοκρατίας και σε αύξηση του κόστους. Κατά την επεξεργασία της στρατηγικής Ευρώπη 2020 πρέπει να ληφθούν επίσης υπόψη και τα αίτια που οδήγησαν στην χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση. Η πολιτική συνοχής έχει ως στόχο την ανάπτυξη σε όλους τους τομείς. Έπειτα, πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες του κάθε κράτους μέλους στην ε, αναθεωρήσει τη στρατηγική. Χρειάζομαστε επίσης ε, σωστά στρατηγικά στοιχεία, ποιοτικά ε, στατιστικά με συγχωρείτε στοιχεία. Ιδιαίτερα για τις εξόχως ε, απόκεντρες περιοχές και τις παραμεθόριες περιοχές της Ένωσης. Η πολιτική συνοχής είναι καλά πλαισιωμένη από την στρατηγική 2020 και τους στόχους αυτής. Τώρα θα ήθελα να σας υπενθυμίσω τα κύρια σημεία της ε, ανταλλαγής απόψεων του Μαρτίου, τα οποία θα βρείτε και στο κείμενο. Καταρχάς, ο κεντρικός, ο αποφασιστικός ρόλος της πολιτικής συνοχής στην ε, επίτευξη των στόχων ε, της Ευρώπης 2020. Έπειτα, Πρέπει να τονίσουμε ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, ΕΦΣΥ, είναι ένα συμπληρωματικό μέσο της ε, πολιτικής συνοχής και των διαρθρωτικών ταμείων της Ένωσης. Τρίτον, η στρατηγική Ευρώπη 2020 θα πρέπει να επιτρέψει την πολυ... Ε, ε, πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και την δημιουργία ενισχυμένων σχέσεων και στην ε, απλούστευση της ε, διοίκησης. Επίσης, όπως είπαν και αρκετοί συνάδελφοι στην ε, τελευταία μας συνάντηση και η κυρία Κρέλα νίκη σε αυτούς, υπάρχουν Υπάρχει η ανάγκη για να έρθει η διοίκηση πιο κοντά στους πολίτες. Και χρειάζεται επομένως ενίσχυση των υφισταμένων ε, δυνατοτήτων. Επίσης, χρειάζεται εκ νέου αναθεώρηση των ε, στόχων της Στατικής Ευρώπη 2020 και αξιολόγηση της εφαρμογής τους. διότι παρατηρούνται διαφορές από περιφέρεια σε περιφέρεια. Υπάρχουν διαφορετικά δεδομένα και διαφορετικές ιδιαιτερότητες ε, ούτως ή άλλως και χρειάζεται λοιπόν αυτό να αναφερθεί ε, σαφώς στο κείμενο. Χρειάζεται επίσης να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις αεροκατοικημένες περιφέρειες. Έπειτα, πολιτική βασισμένη σε πολλά και διαφορετικά κριτήρια, οικονομικά δεδομένα, για, αν είναι μια περιοχή αστική ή όχι. Θεωρούμε σημαντικό ότι πρέπει να ενισχυθεί και η ευθύνη των τοπικών αρχών. Και αυτά για μένα θεωρούνται ε, θετικά στοιχεία στην αναθεώρηση της ε, στρατηγικής. Πιστεύω πως η ανταλλαγή απόψεων για το μέλλον των διαρθρωτικών ταμείων και της μακροπρόθεσμης στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά το 2020, μετά την περίοδο δηλαδή 2014-2020, πρέπει να γίνει εγκαίρος. Χωρίς όμως να χωρίς, ε, χωρίς όμως να δημιουργηθούν προβλήματα στην εφαρμογή του φυστάμενου πλαισίου. Επίσης, θα ήθελα να τονίσω ότι το 2019 θα έχουμε μια νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ένα νέο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και χρειάζεται λοιπόν αναθεώρηση της ε, στρατηγικής ε, μέχρι τότε καθώς επίσης και θα χρειαστεί να αρχίσει η εφαρμόγη του επόμενου πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Και του των ελευθέντων θα ήθελα να πω ότι στις 2 Ιουλίου έχουμε την προθεσμία υποβολής τροπολογιών και τον Σεπτέμβριο θέλουμε να τον Ιούλιο, μάλλον την 1η Ιουλίου το απόγευμα θα γίνει και μία ακρόαση όπου θα έχουμε εκπροσώπους ε, διάφορων ε, ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και σας καλώ όλους να παραστείτε. Και το επεξηγηματικό σημείωμα θα βρείτε μία πιο λεπτομερή περιγραφή των ε, όσων σας είπα μόλις τώρα. Με χαρά μου λοιπόν να ακούσω τα σχόλιά σας και τις ερωτήσεις σας καθώς και τις τροπολογίες σας. Σας ευχαριστούμε πολύ κυρία Κρέλ. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ και την εισηγήτρια. Πιστεύω πως το σχέδιο έκθεσης είναι αρκετά ενδιαφέρον και καλογραμμένο. Αναφέρονται πάρα πολλά ε, πράγματα τα οποία συζητήσαμε ήδη την προηγούμενη φορά Και είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η σύγκριση με το τι καταφέραμε το 2007 και το 2013 και πόσο μπορούμε να το συνδέσουμε με την Στρατηγική Ευρώπη 2020. Υπάρχουν αναλύσεις, όμως πιστεύω πως χρειάζονται βελτίωση. Και αναθεώρηση και επικαιροποίηση με την πάροδο του χρόνου. Επίσης, σχετικά με την ενδιάμεση αναθεώρηση, θα ήθελα να πω ότι δεν χρειάζεται να γίνουν μεγάλες αλλαγές, ιδιαίτερα στην πολιτική συνοχή, διότι έτσι θα δημιουργηθεί σύγχυση και θα περιπλέξουμε τα πράγματα. Αντιθέτως, θα ήθελα να διαφαίνεται με σαφέστερο τρόπο στην έκθεση ότι η πολιτική συνοχή ε, δεν έχει σκοπό να εφαρμόσει και να ελοπίσει την στρατηγική Ευρώπη 2020, αλλά για να ε, ενισχύσει, να δημιουργήσει και να ενισχύσει την ε, εδαφική συνοχή και την οικονομική ανάπτυξη και ιδιαίτερα φροντίζοντας να δοθεί έμφαση στις περιοχές, στις πιο αεροκατοικημένες περιοχές ή στις περιοχές που αντιμετωπίζουν προβλήματα. Η Στρατηγική Ευρώπη 2020 είναι ε, ένα βοηθητικό εργαλείο και ο εισηγητής ε, νομίζω το ανέφερε αυτό σε, ένα, ε, σε μια υποσημείωση, όμως πιστεύω πως πρέπει να τονιστεί αυτό, διότι Φαντάζομαι πως ε, υπάρχουν ε, πολλοί που επιθυμούν να καταργηθεί εντελώς η Ιστεργική Ευρώπη 2020. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να το αναφέρουμε. Και κάτι άλλο. Δεν ξέρω κατά πόσο βοηθά, αλλά στην παράγραφο 14 αναφέρεται ότι πρέπει να δώσουμε έμφαση σε περιφερειακούς στόχους. Αυτό που καταλαβαίνω εγώ με αυτό είναι ότι, ότι δεν θα είναι πάντα δυνατόν να γίνει δεδομένων των διαφορετικών δομών που υπάρχουν στα κράτη-μέλη. Εδώ πιστεύω πως δεν πρέπει να προσπαθήσουμε να εισαγάγουμε δομές που θα περιπλέξουν τα πράγματα και θα αυξήσουν τη γραφειοκρατία, αλλά να κάνουμε προτάσεις οι οποίες κατά την εφαρμογή τους πραγματικά θα μα δώσουν τη δυνατότητα να επικεντρωθούμε στα περιφερειακά, συγκεκριμένα περιφερειακά ζητήματα και θα διευκολύνουν τη συνεργασία μεταξύ κρατών μελών. Θα βοηθήσουν δηλαδή στην υλοποίηση των ε, βασικών μας στόχων. Τέλος, Φυσικά, καλωσορίζω το γεγονός ότι αφιερώθηκε μία ξεχωριστή παράγραφος μόνο για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές, όμως ε, θεωρώ πως αυτό ε, γίνεται εις βάρος άλλων περιφερειών, οι οποίες αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες δυσκολίες. Νησιά, για παράδειγμα, ή αραιοκατοικημένες περιοχές και περιφέρειες, πρέπει να συμπεριληφθούν και αυτές ε, οι περιφέρειες στην έκθεση, διότι πραγματικά κατά την ενδιάμεση αναθεώρηση θα πρέπει να γίνει ιδιαίτερη μνήα στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν αυτές οι περιοχές και πώς μπορούμε να τα λύσουμε χρησιμοποιώντας και τη στρατηγική 2020. Επίσης φυσικά αναφέρεται κύριε Ισηγητά ότι πρέπει να επικεντρωθούμε σε συγκεκριμένες προτεραιότητες. Αυτό με βρίσκει απόλυτα σύμφωνη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να δώσουμε το μήνυμα ότι τα λίγα χρήματα που έχουμε στη διάθεσή μας θα τα χρησιμοποιήσουμε με όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερο τρόπο έτσι ώστε να υλοποιηθούν οι στόχοι της ε, ευρωπαϊκής πολιτικής. Γι' αυτό λοιπόν θα υποβάλω σχετικές τροπολογίες και ε, πραγματικά με χαρά μου αναμένω την ακρόση της ε, Ιουλίου. Σας ευχαριστώ πολύ. Ξεκινήσαμε λοιπόν με τους σκιώδεις ηγητές. Πρώτη ήταν η κυρία Κρέλ και τώρα θα συνεχίσουμε με τον κύριο Παπαδημούλη. Α, η κυρία Τόμασίτς. Εσείς πρώτα κυρία Τόμασιτς. Θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Ρούας για την εξαιρετική του έκθεση και τις συγκεκριμένες προτάσεις. Αυτές τις προτάσεις θα πρέπει να τις λάβει υπόψη η Κομισιόν όταν θα εκπονήσει προτάσεις για την ενδιάμεση αξιολόγηση της Αττικής του 2020 που θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη του 2015. Μια βελτιωμένη, αναθεωρημένη στρατηγική για την Ευρώπη του 2020 θα ενδυναμώσει την ανταγωνιστικότητα. Θα παίξει σημαντικό ρόλο για την εφαρμογή και της νέας οικονομικής διακυβέρνησης για μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα και ανάπτυξη. Η γενική η βασική στόχη της στρατηγικής Ευρώπη 2020 και σε ευρωπαϊκό και σε εθνικό επίπεδο δεν προσαρμόζονταν πάντοτε στις ε, πραγματικότητες ε, ή στο δυναμικό των πόλεων και των περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενίοτε διαφορετικά μέτρα, δείκτες ή ποσοτική ε, θα ήταν πιο ενδεδειγμένη προσέγγιση για να εφαρμοστεί αποτελεσματικά αυτή η στρατηγική. Καλό θα ήταν να υπάρχει επίσης μία μονοαπευθυντική θηρίδα, ένα one-stop shop για εξορθολογισμό των διαδικασιών και των δράσεων. Η προσέγγιση αυτή θα βοηθήσει να αποθεθούν επικαλύψεις και θα δημιουργήσει συνέργειες. Θα ήθελα να υπογραμμίσω επίσης τη μεγάλη σημασία της ε, προσέγγισης που θα λαμβάνει υπόψη τα τοπικά και τα περιφερειακά χαρακτηριστικά και όχι μόνο εθνικούς ε, ε, στόχους. θα πρέπει να είναι ένας γνώμονας η στρατηγική αυτή και για την ανταλλαγή καλών πρακτικών. Ο διάλογος μεταξύ εθνικών, περιφερειακών, τοπικών αρχών θα φέρει πιο κοντά τους πολίτες στις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα τους δώσει την αίσθηση της ε, ιδιοποίησης, της κυριότητας ε, της στρατηγικής αυτής. Ευχαριστώ. Sorry, Mr. Van Miltenburg. Συγγνώμη, πρόκειται ο κύριος Βαν Μίλτεμπρουκ. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Πρόεδρε, θέλω να συγχαρώ τον εισηγητή. Και δεν το λέω απλά για να το πω. Πραγματικά είναι εξαιρετικό το έγγραφο, το στηρίζω. Βέβαια, πιστεύω ότι ε, θα βοηθήσουν και τροπολογίες αρκεί να μην αλλοιώσουν ε, τη γενική κατεύθυνση της έκθεσης. Εξαιρετική και η έκθεση. Και... Ε, συστάσεις των δύο μιλητών. Να μιλήσω καταρχάς για δύο πράγματα. Πρώτο, το Ταμείο Σαρδικών Επενδύσεων. Και δεύτερον, Στρατηγική Ευρώπη 2020. Πώς συνδέονται αυτά τα δύο. Και χρονοδιάγραμμα. Αναθεώρηση δηλαδή. Επανεξέταση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Ευρώπη 2020. Σε σχέση και με το πολιτές νοσομικό πλαίσιο. Έχουμε διάφορα ταμεία. με επενδύσεων, διαφορετικό ταμεία και το περιβόητο ταμείο Juncker ε, το Ευρωπαϊκό των Στατικών Επενδύσεων. Στο πλαίσιο της Αρδικής 2020. Πώς συνδέονται, αν συνδέονται μεταξύ του αυτά τα ταμεία. Εγώ πιστεύω ότι η συνοχή είναι το πλέον σημαντικό οριζόντιο στοιχείο και πολύ σωστά το ανέφερε και ο εισηγητή. Στόχος είναι να επιτευχθούν οι στόχοι της 2020 και να βάλει η πολιτική συνοχή. Υπάρχουν στρατηγικοί στόχοι ξεκάθαροι και θα πρέπει να εγγυηθούμε ότι η πολιτική συνοχή θα έχει σχέση με τη στρατηγική 2020. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων που ανακοινώθηκε με Πανοκρουσίες Λέγεται και στην παράγραφο 16 ότι δεν έχει άμεση σχέση, ξεκάθαρη σχέση με την Ευρώπη 2020. Ίσως καταθέσω σχετική τροπολογία γιατί νομίζω ότι η διατύπωση αυτή είναι αρκετά μετριοπαθής. Έχουμε κάποιους συγκεκριμένου στόχου στρατηγική ε, Ευρώπη δηλαδή 23% του ΑΕΠ ε, πρέπει να επενδυθεί στην έρευνα και την ανάπτυξη, για παράδειγμα. Αλλά αυτοί οι στόχοι θα μπορούσαν να μην επιτευχθούν εάν πηχαίρει σε αυτά τα κονδύλια της ε, στρατηγικής αυτής για άλλου λόγους. Και ίσως να μην προωθηθεί καινοτομία ή να μην δημιουργηθούν οι θέσει εργασία και ανάπτυξη που είναι και οι επιδιωκόμενοι στόχοι. Είναι απαραίτητο, το τονίζει και ο εισηγητή, οι στόχοι να προσαρμοστούν αναπεριφέρεια. Δηλαδή να έχουμε μια εδαφική προσέγγιση. Άλλες περιφέρειες μπορούν να εστιάσουν περισσότερο στην έρευνα και την ανάπτυξη. Άλλες περιφέρειες πρέπει να δώσουν περισσότερη προσοχή στο θέμα της ανεργίας, για παράδειγμα. Πιστεύω λοιπόν ότι πρώτη προτεραιότητα πρέπει να είναι η επίτευξη των γενικών στόχων που δεν θα πρέπει να ε, μας διαφεύγουν. Άρα θα ήθελα ο κ. Συγητής να μου πει Πώς μπορούμε να το πετύχουμε αυτό και έρχομαι στο χρονοδιάγραμμα γιατί είναι και αυτό ένα ζήτημα πολιτική συνοχής, ενδιάμεση αξιολόγηση. Μα λέει στην παράγραφο 12 ο συγητή ότι η διάμεση αξιολόγηση στρατηγική Ευρώπη 2020 θα πρέπει να είναι κάπως περιορισμένη. Είτε μιλάμε για αυτή την στρατηγική 2020 είτε για μετά το 2020 θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να λαμβάνεται υπόψη πολιτική συνοχή και το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο, γιατί όλα αυτά συνδέονται μεταξύ του. Καταλήγω Πρέπει να υπάρχει καλύτερο συντονισμό. Οι στρατηγικοί στόχοι πρέπει να επιτευχθούν. Και η ανάπτυξη, απασχόληση, καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος. Ευχαριστώ πολύ για μια κομφάρα τον εισηγητή. Και περιμένω να μπορέσουμε να συνεργαστούμε περισσότερο πάνω στο κείμενο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Νομίζω ότι όσοι υποστηρίζουμε τον ορθό λόγο θα πρέπει να δούμε τα στοιχεία, τους αριθμούς, τα γεγονότα. Και οι αριθμοί δυστυχώς λένε ότι τα τελευταία χρόνια, κύριε Ρούας, η πολιτική συνοχής έχει αποδυναμωθεί μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει αυξηθεί η φτώχεια, έχει αυξηθεί η ανεργία, έχουν αυξηθεί και οι κοινωνικές ανισότητες και οι περιφερειακές ανισότητες. Αυτό είναι αποτέλεσμα μιας πολιτικής και καταγράφεται και στην πέμπτη έκθεση της συνοχής που μας παρουσίασε η Κομισιόν. Σωστά ισχυρίζονται οι τεχνοκράτες ότι αν δεν υπήρχε η πολιτική συνοχής οι ανισότητες θα ήταν μεγαλύτερες και η φτώχεια και η ανεργία και οι κοινωνικές ανισότητες και οι περιφερειακές ανισότητες. Αλλά αυτό τι σημαίνει ότι όταν μιλούμε για αναθεώρηση πρέπει να εξηγήσουμε τι θέλουμε να αλλάξει. Εμείς πιστεύουμε και εγώ προσωπικά και η πολιτική μου ομάδα ότι πρέπει να ενισχυθεί η πολιτική συνοχής. Και επειδή ο συνάδελφος από τους φιλελευθέρους σωστά επεσήμανε τη σύνδεση με το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, πρέπει να ενισχυθούν οι πόροι που διατίθενται από τον προϋπολογισμό τον κοινοτικό για να ενισχύσουμε την πολιτική συνοχής. Κύριε Ρούας, από ό,τι ξέρω είστε από την Πορτογαλία. Τι είναι η Ευρώπη 2020, η αναθεώρηση των στόχων της Λισαβόνας. Έχουμε μια ιστορία 15 ετών όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση θέτει στόχους η πολιτική που ακολουθείτε και τα μέσα που διατίθενται δεν επιτρέπουν την επίτευξη των στόχων για την απασχόληση, τη συνοχή, την άνοδο της έρευνας, το να μην εγκαταλείπουν τα παιδιά των φτωχών οικογενειών το σχολείο νωρίς, και αντί να αλλάξουμε την πολιτική και να ενισχύσουμε τα μέσα για την επίτευξη των στόχων, αλλάζουμε τους στόχους. Εγκαταλείπουμε τους φιλόδοξους στόχους, έτσι έγινε και με τη Λισαβόνα. Και τώρα, πού είναι οι μελέτες επιπτώσεων από την Κομισιόν, θα πετύχουμε τους στόχους του Ευρώπη 2020 σε ό,τι αφορά την απασχόληση. Αυτό το 75% θα επιτευχθεί, ναι ή όχι. Και η αναθεώρηση θα οδηγήσει στην ενίσχυση των προσπαθειών για να επιτύχουμε αυτούς τους στόχους. Ή απλώς θα μεταθέσουμε για τρίτη φορά κάποιους στόχους μέσω της αναθεώρησης για την τρίτη δεκαετία. Δέκα χρόνια με τη Λισαβόνα, 10 χρόνια με το Ευρώπη 2020, άντε άλλο ένα ραντεβού για την επόμενη δεκαετία από το 2020 μέχρι το 2030. Αυτά πρέπει να συζητήσουμε και να δούμε εάν η ισχύουσα πολιτική των νεοφιλελεύθερων Ταλιμπάν που έχουν μια θρησκευτική πίστη στην άποψή τους ακόμη και αν τη διαψεύδει η πραγματικότητα, θα αλλάξει. Θέλουμε ανάπτυξη. Θέλουμε κοινωνική συνοχή. Γιατί δυσχωρείτε κυρία Πρόεδρε. Μιλώ λίγο, δεν μιλώ πολύ. Και ο Πρόεδρος ή η Πρόεδρος οφείλει να ακούει όλους τους ομιλητές με την ίδια προσοχή. Έτσι. Και χωρίς σχόλια και μορφασμούς. Ευχαριστώ πολύ. Λέω λοιπόν ότι ο κύριος Ρούας κάνει μια φιλότιμη προσπάθεια να θέσει κάποιους στόχους, αλλά νομίζω ότι πρέπει να βάλουμε το δάκτυλο στην πληγή και να συνεννοηθούμε. Υπάρχουν κάποιοι που θέλουν να καταργήσουν και αυτή την ισχυρή πολιτική συνοχής και λένε ότι και αυτά τα λεφτά πρέπει να λιγοστέψουν και να πάνε για επενδύσεις, να πάνε στους πιο πλούσιους, στους πιο ισχυρούς, στις επιχειρήσεις. Υπάρχουν και κάποιοι άλλοι που λένε ότι πρέπει να ενισχυθεί η πολιτική συνοχής για να καταπολεμήσουμε τις ανισότητες και τις κοινωνικές και τις περιφερειακές. Εμείς θα καταθέσουμε τροπολογίες ζητώντας να ενισχυθεί αυτή η διάσταση, η κοινωνική αναπτυξιακή. Πιστεύουμε ότι πρέπει και αυτοί οι στόχοι να μπουν με την ίδια δεσμευτικότητα για να μιλάμε όχι απλώς για ένα σύμφωνο σταθερότητας, αλλά για ένα σύμφωνο βιώσιμης ανάπτυξης της Ευρώπης και της ευρωπαϊκής οικονομίας και θα εξαρτήσουμε την στάση μας στην ε, τελική, τελικά απέναντι στην έκθεση Ρούας ανάλογα με το πόσο ο θα αντιμετωπίσει τις τροπολογίες που θα καταθέσουμε στη διάρκεια των ημερών που έχουμε μπροστά μας. Ευχαριστώ. Thank you, Madame Vanna. Ευχαριστώ πολύ. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω για την παρουσίαση της μελέτης Πιστεύω πως πραγματικά μας δίνει μια καλή γενική εικόνα για τα νέα στοιχεία που έχουν ε, εισαχθεί και θα μας βοηθήσει στο έργο μας σε αυτήν εδώ την Επιτροπή. Και επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο ακόμα, ε, θα περιοριστώ σε μία συγκεκριμένη ερώτηση. Έχει να κάνει με την ε, εφαρμογή της αρχής της εταιρικής σχέσης. Πιστεύω πως αυτή η αρχή είναι ένα από τα σημαντικότερα καινούρια στοιχεία για την νέα περίοδο και είμαι πεπισμένη ότι θα μας βοηθήσει στον προγραμματικό σχεδιασμό και στις ε, συζητήσεις και διαβουλεύσεις με τους ε, ενδιαφερόμενους ε, φορείς. Αυτή η αρχή είναι κάτι που θεωρώ πως είναι κάτι πάρα πολύ θετικό και θα ήθελα να ρωτήσω αυτή η θετική αξιολόγηση της αρχής της εταιρικής σχέσης θα συμπεριλάβει τους κοινωνικούς εταίρους, θα συμπεριλάβει όλους τους ενδιαφερόμενους ε, φορείς σε όλα τα στάδια της ε, διαδικασίας. Σύμφωνα με αυτά που προβλέπει ο κανονισμός, κατά το προπαρασκευαστικό στάδιο του σχεδιασμού, όταν γίνεται, ε, γίνεται λόγος για την συμπερίληψη στον ε, σχεδιασμό και στην παρακολούθηση. Και αναφέρεται επίσης ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα έπρεπε να παίξει έναν τέτοιο εποπτικό ρόλο. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να ρωτήσω περισσότερα γι' αυτό. Τώρα σχετικά με την έκθεση του κυρίου Ρούας. Ήδη κατά την πρώτη ανταλλαγή απόψεων στην Επιτροπή εξέφρασε την άποψη ότι η έκθεση είναι πολύ εξισορροπημένη και πως με βρίσκει σύμφωνη σε πάρα πολλά σημεία. Υπάρχουν βέβαια και ορισμένα σημεία τα οποία βλέπω με αρκετή επιφύλαξη, ήδη τα ανέφεραν και οι προλελήσαντες, πρέπει να προσέξουμε το τοπικό και το περιφερειακό επίπεδο ε, στο οποίο θα ε, χρειαστούν επενδύσεις, επενδύσεις σε μεγάλη κλίμακα και αυτές οι επενδύσεις από πού θα προέλθουν, από τα διαρθρωτικά ταμεία. Η σημασία των επενδύσεων ε, πρέπει να τονιστεί, δεν πρέπει να υποτιμήσουμε την αξία ε, των επενδύσεων. Η στρατηγική Ευρώπη 2020 έχει δημιουργήσει ε, τις σωστές προϋποθέσεις και εμείς πρέπει να φροντίσουμε για την πολιτική εφαρμογή της στρατηγικής αυτής, ιδιαίτερα ε, για τις ε, περιφέρειες οι οποίες ε, δεν έχουν τα οικονομικά μέσα για να επιτύχουν τους στόχους της στρατηγικής. Πρέπει λοιπόν να τονιστούν οι στόχοι, ιδιαίτερα για αυτές τις πιο αδύναμες περιφέρειες. Τώρα, η διατύπωση βέβαια ορισμένων περιφερειακών στόχων δεν με βρίσκει απόλυτα σύμφωνη. Δεν αναφέρονται για παράδειγμα προτεραιότητες. Πιστεύω πως πρέπει να αναφερθεί η έλλειψη πολιτικής θέλησης, η έλλειψη συγκεκριμένων στόχων και η έλλειψη της ε, διαπραγματευτικής δυνατότητας. Πιστεύω πως πρέπει να ενισχυθεί ο τοπικός παράγοντας για να μπορέσει να συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της Ευρώπης 2020. Και ε, σχετικά με την τεχνική προσαρμογή έχω μία σύντομη παρατήρηση. Την τελευταία φορά που συζητήσαμε αναφέραμε τον κανονισμό για τις ε, κοινέ ε, διατάξεις. Πιστεύω πως θα χρειαστούν κάποιες τροπολογίες που θα αφορούν την βιώσιμη ανάπτυξη και τις ποιοτικέ θέσεις εργασίας ε, και στοιχεία που θα ε, ενισχύσουν την συμμετοχική διαδικασία. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Τέσσερα μέλη έχουν ζητήσει το λόγο ακόμα. Θα σας ζητήσω να είστε πολύ σύντομοι, διότι έχουμε ξεφύγει εντελώς από το πρόγραμμά μας. Και αυτό μου θυμίζει ότι ίσως ε, θα χρειαστεί να περιορίσουμε το χρόνο αγόρευσης των μελών. Γιατί διαφορετικά δεν θα καταφέρουμε να τελειώσουμε την εμερήσια διάταξη. Δεν γίνεται όταν ο καθένας μιλάει για πάρα πολύ ε, καιρό. Κυρία Μόρκοβα, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Συμφωνώ μαζί σας, κυρία Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη. Θέλω να εκτιμήσω τη μελέτη που παρουσιάστηκε εδώ. Είναι μεγάλη η μελέτη, πολύ καλή. Και με, μου να ε, θέσω κάποιες ερωτήσεις που θα τις διατυπώσω ίσως και το απόγευμα μιλώντας στην Επίτροπο. Πιστεύω ότι η Επίτροπος θα πρέπει να απαντήσει. Θα περιοριστώ σε δύο σύντομες ερωτήσεις και θα εκτιμούσα απάντηση. Ανησυχώ, διότι στα συμπεράσματα στο σημείο 7 η έκθεση λέγει ότι δεν υπάρχουν μεγάλα σημάδια απλούστευσης. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε να εξασφαλίσουμε ότι όσον αφορά τα διθετικά ταμεία και την πολιτική συνοχής ότι θα πετύχουμε τη μεγαλύτερη δυνατή απλούστευση των διαδικασιών. Γι' αυτό διερωτώ Μήπως τη μελέτη σας το αναφέρετε. Δεν είχα το χρόνο να εξετάσω το κείμενο λεπτομερώς και διαρωτώ με κατά πόσο το πρόβλημα της έλλειψης απλούστευσης οφείλεται στην πολύ μεγάλη γραφειοκρατία, στο διοικητικό άχθος. Τι κρύβεται πίσω από αυτό το ότι η απλούστευση δεν έχει επιτευχθεί. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για τους τελικούς ε, δικαιούχους. Και ένα άλλο ερώτημα. Συνεργαστήκατε με 11 κράτη-μέλη. Είναι ένα σχετικό δείγμα. Ποιος σας έδινε πληροφορίες, τα Υπουργεία, οι Περιφέρειες, πληροφορίες ερχόταν και από τα δύο επίπεδα. Τα συμπεράσματά σας τροφοδοτήθηκαν σε εκείνους που σας έδωσαν τις πληροφορίες. Είμαι από τη Σλοβακία και του χρόνου η Σλοβακία θα αναλάβει την Προεδρία της Ένωσης και πιστεύω ότι κατά τη διάρκεια της Προεδρίας θα χρειαστεί να επιφέρουμε νέες βελτιώσεις στην πολιτική συνοχής. Δώσατε πληροφορίες σε εκείνους που σας έδωσαν τις πληροφορίες αρχικά στα κράτη-μέλη με τα οποία συνεργαστήκατε. Και κάτι άλλο. Ενθαρρύνεται την Ευρωπαϊκή Ένωση να παρακολουθεί την εφαρμογή Τη αρχής τη εταιρική σχέση στην υλοποίηση των προγραμμάτων. Είναι σημαντικότατο, διότι η αρχή τη εταιρική σχέσης είναι σημαντικότατη για τον προγραμματισμό. Εξαλείφει τη δυνατότητα επικάλυψης και διαφθοράς. Αυξάνει τη διαφάνεια. Και ίσως κάποιος στην Επιτροπή μας ίσως να ετοιμάσει έκθεση ιδίας πρωτοβουλία για να εξετάσει το θέμα στο μέλλον. Αυτά είχα να ρωτήσω. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ λέει Πρόεδρος. Ο κ. Μαζί είναι επόμενο να πάρει το λόγο. Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ. Οι συζητήσεις που έγιναν σήμερα το πρωί ήταν άκρο ενδιαφέρουσες και οι συζητήσεις για την έκθεση του συναδέλφου Ρουάς δεν απομακρύνεται πολύ από τη συζήτηση που διεξήχθη το πρωί με την διάσκεψη για τις παράξει περιφερειακές περιοχέ Συνοψίζοντα, εν πρώτης, πρέπει να επαναλάβουμε και στην έκθεση έκθεση συνοχής να επανέλθουμε σε αυτό στην έκθεση έκθεση που λέει ότι οι στόχοι της συνοχής έχουν υποχωρήσει σοβαρά από το 2008 και μετά και αυτό υπόθηκε από τον συνάδελφό μου, τον κύριο Δημήτρη Παπαδημούλη. Δεν θα μακρηγορήσω, αλλά θα ήθελα να παραθέσω την έκθεση, την έκτη έκθεση συνοχής, η οποία αναφέρει ότι μετά την κρίση του 2008 το εισόδημα πάρα πολλών πολιτών της Ευρωπαϊκής μειώθηκε το επίπεδο απασχόλησης υποχωρεί στις περισσότερες χώρες μέλη. Η ανεργία ποτέ δεν ήταν τόσο υψηλή α, εδώ και τουλάχιστον 20 χρόνια. Ότι το φαινόμενο του κοινωνικού αποκλεισμού επιδεινούται και η φτώχεια επιδεινούται εξίσου παντού. Και σαν συνέπεια αυτών οι διαφορές οι περιφερειακές όσον αφορά την απασχόληση και την ανεργία έχουν επιδεινωθεί. Έχουν αυξηθεί μάλλον διαφορές. Μετά η άλλη ανησυχία Έχουμε το συνέστημα ότι η περιφερειακή πολιτική σήμερα έχει αποδυναμωθεί, έχει χάσει τη φύση της και έχει συναρτηθεί με νέους στόχους, νέους στόχους που δεν θα διορθώσουν τελικά τις διαφορές της αναπτυξιακές και δεν θα διευκολύνουν την σύγκληση που απαιτούν οι συνθήκες. Και τρίτον, ανησυχίες όσον αφορά το μέλλον, τι θα γίνει μετά το 2020. Τώρα, όσον αφορά τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ενώσεως για το 2020, είχαμε πει για την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020 για τις περιφέρειες. Τους είπαμε ότι ο δικός σας χάρτης για το 2014-2020 είναι η στρατηγική της Ευρωπαϊκής ε, ε, Ενώσης 2020. Καθορίστε στόχους και θα πετύχετε. Έχετε συμφέρον να πετύχετε στόχους. Όμως δεν λάβαμε καθόλου υπόψη στοιχεία μακροοικονομικά και στοιχεία που άπτονται των εφαρμοζομένων πολιτικών σε επίπεδο κατών μελών. Είναι το εθνικό πλαίσιο, το ευρωπαϊκό πλαίσιο και το διεθνές. Και υπάρχουν όλοι αυτοί οι περιορισμοί που εμποδίζουν τις περιφέρειες από το να κινηθούν προς τους στόχους αυτούς. Πιστεύω λοιπόν ότι εμεί δεχτήκαμε να συναντήσουμε την περιφερειακή πολιτική με τους στόχους της στρατηγικής Ευρώπης το 2020. Σας το λέω, λέω ότι σκέφτομαι για να μην αφήσουμε να περάσει η στρατηγική 2020 όπως εξέπνευσε και η στρατηγική της Λισαβόνας και να βάγει η στρατηγική της Λισαβόνας δεν θέλουμε να βαγίσει και αυτή αυτή είναι η πραγματικότητα που θέλουμε να τονίσουμε και το τελευταίο σε αυτή τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2020. Πιστεύω ότι δεν λαμβάνουμε υπόψη επαρκώς την οικονομία την τόπια, την τοπική. Δηλαδή σε πολλές περιφέρειες, σε πολλές περιοχές δεν είναι οι μεγάλες βιομηχανίες οι επενδύσεις που δίνουν τη μεγάλη προστιθέμενη αξία ακόμα και είναι αναγκαίε. δεν έχουν αυτά το μεγαλύτερο αντίκτυπο όσον αφορά την απασχόληση. Σε πολλές περιοχές και περιφέρειες ο πρώτο εργοδότης είναι τα νοσοκομεία, η τοπική αυτοδιοίκηση και τρίτον, πολύ συχνά, τα εμπορικά κέντρα. Είναι οι εργοδότες, αυτή είναι η πραγματικότητα για πολλές περιοχές στην Ευρώπη που έχουν μείνει πίσω αναπτυξιακά και πιστεύω ότι η έκθεση θα έπρεπε αυτό να το λαμβάνει υπόψη. Ευχαριστώ. Πολτσακ. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ. Θα προσπαθήσω να μείνω στα δύο λεπτά. όπω ζητήσατε, θέλω να συγχαρώ τον κύριο Ρούας. Εξαιρετική έκθεσή του. Σε ό,τι δεν αφορά τη συζήτηση για το σημείο 14, εγώ έχω αντίθετη άποψη. Νομίζω δηλαδή ότι πολύ σωστά τα λέει ο κύριος ε, Ρούα. Έχει επιλέξει σωστή διατύπωση. Νομίζω ότι πρέπει να έχουμε υπόψη ε, τους περιφερειακούς στόχους ακριβώς σε σχέση με τη στρατηγική για την Ευρώπη του 2020. Άρα διαφορούν τους προλέλησαν τους συναδέλφους που είχαν αντίθετη άποψη. Επίσης θεωρώ ότι θα πρέπει να έχουμε στοιχεία από την Κομισιόν για να δούμε τι ρόλο διαδραματίζουν οι τοπικές αρχές. Έτσι θα μπορέσουμε όταν έρθει η στιγμή της ενδιάμεσης αξιολόγησης να βασιστούμε ε, στα στοιχεία αυτά των αρχών, των τοπικών αρχών και στην κατάστασή τους και εκεί να βασίσουμε αυτή την αξιολόγηση. Το πιο σημαντικό στοιχείο το έδωσε ο κύριος Ρώας στο τέλος της εισαγωγής του όταν ρώτησε τι κάνουμε μετά το 2020. Πιστεύω ότι η έκθεση αυτή θα μπορούσε να συμπληρωθεί ακριβώς με αυτό που είπε στο τέλος της τελογικής του έκθεσης, συγκεκριμένα το σημείο 19 και το σημείο 20. Αυτά τα σημεία νομίζω ότι ε, θα πρέπει να συμπληρωθούν από όσα λέει στο τέλος στην ετολική του έκθεση. Νομίζω ότι σίγουρα αυτή η συζήτηση έχει σχέση με την προηγούμενη, τη μελέτη των δύο κυρίων, Μπάρτλερ και Κα, όπου λέγεται σε αυτή τη μελέτη θα πρέπει να υπάρχει περισσότερο συντονισμός. Είναι κάτι που δεν το έχουμε πετύχει. Τα κράτη-μέλη λένε ότι φταίει η Κομισιόν, η Κομισιόν λέει ότι φταίνουν τα κρατη Δεν θέλω να είμαι ο κριτής, αλλά πιστεύω ότι θα πρέπει να εκφράσουμε την άποψή μας για την ανάγκη καλύτερου συντονισμού. Και πρέπει να ακούσουμε και την άποψη των περιφερειών. Η εμπειρία των περιφερειών είναι σημαντική γιατί αυτή είναι ο κινητήριος μοχλός, η περιφέρεια είναι ο κινητήριος μοχλός. Αυτή είναι η πρώτη μου παρατήρηση, δεύτερη παρατήρηση. Για τη μελέτη πάντα. στην περίληψη λέει ότι η αρχή της εταιρικής σχέσης έγινε σεβαστή κατά μεγάλο βαθμό. Το διάβασα συγκεκριμένα έτσι στο έγγραφο. Τι θα πει αυτό. Διαπιστώθηκαν παρά τα αυτά ελλείψεις και ανεπάρκειες σε ό,τι αφορά την εφαρμογή της αρχής εταιρικής σχέσης. Ο κύριος Φανίστελ Ρόι, ευχαριστώ πολύ. Δεν έχουμε πολύ χρόνο, άρα δεν θα ασχοληθώ με την ε, μελέτη, αλλά θα θέσω το ερώτημα. Πώ θα συνεχίσουμε. Έχουμε αυτή την έκθεση δύο πρωτοβουλία. Πέρχεται σε πολύ σωστή χρονική στιγμή, γιατί θέλουμε να δούμε τι κάνουμε με αυτή τη στρατηγική 2020. Το ίδιο κάνει όμω και η Επιτροπή Απασχόληση, αλλά δεν ανταλλάξαμε γνωμοδοτήσει. Είναι κάπω τρελό ότι σύντομα εμεί ολοκληρώνουμε το έργο μα, πηγαίνουμε στην Ολομέλεια με δύο εκθέσει ασυντόνιστα μεταξύ των δύο επιτροπών. Η κάθε μία στη δική της βέβαια, στο δικό της πεδίο αρμοδιτών, αλλά χωρίς να έχουμε συντονιστεί μεταξύ μας. Πώς θα πετύχουμε τη μεγαλύτερη συνεκτικότητα στο Κοινοβούλιο. Υπάρχει μάλιστα αυτή την εβδομάδα μια μεγάλη ακρόαση της Επιτροπής Απασχόλησης για το μέλλον της Αθήκης για την Ευρώπη 2020. Βέβαια όλοι μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε εδώ μέσα, αλλά τέλος πάντων. Τι να πω. Η πρόεδρος ή κάποιος άλλος δεν μπορεί να το λύσει αυτό το πρόβλημα. Να υπάρχει δηλαδή μια συντονισμένη συζήτηση στην Ολομέλεια για την Ευρώπη 2020. Εμείς ετοιμάσαμε τη στρατηγική και δώσαμε και τα λεφτά. Μιλάω για το δεύτερο ταμείο βέβαια και το κοινωνικό ταμείο. Δεν θα έπρεπε να έχουμε μια συντονισμένη δράση και να προετοιμαστούμε. Όχι απλά να κάνουμε μια συζήτηση να μην μείνει αυτή η έκθεση σε απλά κάποια παρουσίαση του εισηγητού, δύο-τρία λόγια από τους υπόλοιπους και μετά τίποτε. Όχι, αξίζει πολύ περισσότερα. Δεν ξέρω, ίσως πρέπει και κάποιες άλλες επιτροπές ε, να ασχοληθούν, αλλά λίγο με ανησυχεί αυτός ο τρόπος εργασίας, δεν μου φαίνεται πολύ καλός. Πρώτος και εγώ ανησυχώ. Γιατί πράγματι δαπανάμε χρόνο να επαναλαμβάνουμε ουσιαστικά τα ίδια και τα ίδια αντί να εστιάζουμε στη βασική συζήτηση. Όμως, ένα από τα συμπεράσματα, ένα από τα πορίσματα της μελέτης, είναι καλύτερο συντονισμό μεταξύ των επιτροπών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και ακριβώς αυτό είπατε κι εσείς. Σίγουρα δεν μπορούμε να σταματήσουμε μια άλλη επιτροπή από το να κάνει τη δουλειά της, αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε όμως είναι να προσπαθήσουμε να έχουμε ένα είδος συντονισμού. Για να δώσουμε ένα συμπληρωματικό όραμα. Σας ευχαριστώ και τώρα θα δώσω το λόγο. Α, ξέχασα. Με συγχωρείτε κύριε Μοσκού, σας ξέχασα. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, Τρεις παρατηρήσεις αν με επιτρέπετε. Πρώτον, είμαστε εδώ σε ένα θεσμικό όργανο. Όλοι, νομίζω τουλάχιστον, εκλεγήκαμε, έχουμε τα ίδια δικαιώματα, τις ίδιες υποχρεώσεις. Και δεν μου αρέσει που κάποιοι συνάδελφοι ε, μιλάνε πάρα πολύ γρήγορα και άλλοι όχι. Πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία. Εγώ έρχομαι έχοντα διανύσει μια απόσταση 8.000 χιλιόμετρων και έρχομαι εδώ, έχω μείνει ένα μήνα εδώ και θέλω να συζητήσουμε για αυτή την πολύ σημαντική έκθεση. Υπάρχουν κάποιε παρατηρήσει που πρέπει να συζητήσουμε. Σήμερα το πρωί είχαμε δύο πολύ σημαντικέ εκθέσει, δύο σημαντικέ ακροάσεις μετά το πέρα των οποίων υποτίθεται πρέπει να γίνει συζήτηση και δεν μπορούμε να φτάσουμε μέχρι το τέλο. Είναι λυπηρό. Ή θα πρέπει να εφαρμοστεί μια πειθαρχία, να υπάρξει πειθαρχία από όλου στον χρόνο αγόρευση, γιατί νομίζω ότι αυτό είναι και ο καλύτερο τρόπο να διαχειριστούμε την κατάσταση. Αλλιώ δεν γίνεται. Είχα κάποιε παρατηρήσει για την έκθεση. Θα συγχαρώ τον εισηγητή φυσικά όπω και οι υπόλοιποι. Ελπίζω να μπορέσω να καταθέσω και εγώ τι τροπολογίε μου. Και με ικανοποίηση διαπιστώνω ότι αφιερώσατε έστω και μια παράγραφο στις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες και στα υπερπόντια ε, διαμερίσματα και εδάφη. Έχουμε το άτομο 349 που είναι πολύ σημαντικό γιατί κατά κάποιο τρόπο ε, αναφέρει τις ιδιαιτερότητές μας και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε ως υπερπόντια εδάφη. Πολύ καλό αυτό. Θα καταθέσω σχετικά κάποιες τροπολίες. Όμως, κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να οργανωθούμε καλύτερα. Δεν ξέρω αν χρειάζεται να κάνουμε πιο πολλές συνεδριάσεις ή ας κρατήσουν δύο μέρες. Αλλά έχουμε 17 σημεία, πολλές εκθέσεις, συζητήσεις. Είναι και κουραστικό και τρέχουμε και δεν φτάνουμε. Άλλοι μιλάνε γρήγορα, άλλοι μιλάνε αργά. Έχω εργαστεί και αλλού, ήμουν 10 χρόνια στην Συνέλευση. Ε, έχω εμπειρία από άλλα θεσμικά όργανα. Πρέπει να βελτιώσουμε τη μέθοδο εργασία μας. Thank you. Σας ευχαριστώ πολύ. Πράγματι είναι ένα θέμα. Ε, όλοι πρέπει να προσπαθήσουμε να βρούμε ένα τρόπο. Πράγματι ένας τρόπος είναι να περιορίζουμε το χρόνο αγόρευσης για τη συμμετοχή στις συζητήσεις, γιατί μόνο έτσι μπορούμε κάπως να προγραμματίσουμε το χρόνο μας και έτσι όλα τα σημαντικά θέματα που είχαμε στην ημερήσια διάταξη για σήμερα, για παράδειγμα, μπορούμε να τα συζητήσουμε. Γιατί είχαμε όλα αυτά τα θέματα που ήταν και αλληλοσυνδεδεμένα μεταξύ τους και η ιδέα μας ήταν να γίνει μια κοινή συζήτηση για όλα αυτά τα θέματα. Πριν διακόψουν διερμηνείς θα δώσω, γιατί έχουμε άλλα πέντε λεπτά, θα ήθελα να δώσω το λόγο στην κυρία Γιάρα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επίσης, ό,τι αφορά τους ε, δύο κυρίους που μας ε, παρουσίασαν τη μελέτη Θέλω να σας ρωτήσω, μπορείτε να δώσετε γραπτές απαντήσεις βουλευτέ. Και θα βρούμε εμεί έναν τρόπο να συζητήσουμε μια ακόμη φορά ίσως. Δυστυχώ είμαστε εκτός ε, χρόνου. Δεν μπορούμε να σα δώσουμε ξανά το λόγο. Κυρία Γιάρα το έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Εκ τη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σημειώνουμε τα σημεία του σχεδίου έκθεση για την περιφερειακή πολιτική σε σχέση και με την ε, αναθεώρηση της, την ε, άμεση αναθεώρηση της στρατηγικής για την Ευρώπη 2020 θα έχει, πρέπει να έχει ολοκληρωθεί αυτή η αναθεώρηση στα τέλη αυτής της χρονιάς ή τις αρχές επόμενης. Και θα λάβουμε υπόψη μας, επεξεργαζόμενη την αναθεώρηση, τα σχόλια του εισηγητή σας για την πολιτική συνοχή και την αναθεώρηση αυτής της στρατηγικής. Ευχαριστώ πολύ. Κύριος Μπέρκοβιτς από την Κομισιόν. Πρέπει ή δεν πρέπει να πάρει το λόγο. Ωραία, δεν πρέπει, οπότε τον ευχαριστώ γιατί δεν έχουμε χρόνο τους ή άλλους. Κύριε Ρούας, εσείς θέλετε λίγο το λόγο. Κάνα δυο λεπτάκια. Ναι, ναι, ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Ούτε καν δύο λεπτά. Θέλω να πω απλά. Υπήρξαν πράγματα που δεν ελήφθησαν υπόψη, γιατί όπως είπα, υπήρχε όριο λέξεων για την έκθεση. Επίσης, «24 χρόνια ήμουν δήμαρχος στην Πορτογαλία. Έχω εμπειρία, αρκετά μεγάλη εμπειρία για όλα αυτά τα θέματα» και ξέρω ότι πρέπει να ε, σεβόμαστε κάποια όρια και κάποιους περιορισμούς. Όλα τα σχόλια τα άκουσα, τα σημείωσα και θα προσπαθήσω να τα συμπεριλάβω στην έκθεσή μου. Συμφωνώ επίσης με την πρόταση του κ. Φανίστελ Ρόι για τον καλύτερο συντονισμό των γνωμοδοτήσεων των διαφόρων επιτροπών. Κυρία Πρόεδρε, ολοκληρώνοντας, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω γιατί δεν θέλω να έχουμε ακόμα καλύτερη καθυστέρηση και να μην χάσω και το δικό μου αεροπλάνο. Thank you very much uh, for this discussion. Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συζήτηση. Εγώ ε, αναλαμβάνω την ευθύνη να έρθω σε επαφή με τις άλλες επιτροπές που θα επεξεργαστούν το ίδιο θέμα για να δω πώς μπορούμε να βελτιώσουμε το κοινό μας έργο στο μέλλον. Σας ευχαριστώ πολύ λοιπόν. Σε αυτό το σημείο ε, θα ολοκληρώσουμε τις εργασίες μας. Διακόπτουμε την πρωινή συνεδρία σε αυτό το σημείο και θα συνεχίσουμε με τη συνεδρίαση των συντονιστών ε, που θα γίνει και κλεισμένα των θυρών. Άρα και χωρίς διερμηνία. Μα έχουμε κάποια ραντεβού με τον κύριο Van Είχατε πει 12.30 θα ολοκληρώσουμε. Εγώ δεν μπορώ να μείνω παραπάνω. Πρέπει να αναβληθεί σας παρακαλώ για το απόγευμα. Τι ώρα. Τι ώρα το απόγευμα. Βλέπω τη μέση διάταξη οπότε προτείνω να ξεκινήσουμε τις συνεδρίες των συντονιστών στις 5.30 αλλά να περιορίσουμε τη συζήτηση μετά τις ψηφοφορίες. Μόνο από το σημείο της μέσης διάταξης. Νομίζω ότι μπορούμε να το πετύχουμε αυτό. Τώρα δεν μπορώ να μείνω. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Πρέπει να φύγω. Yes, Mrs. D'Amato. Siamo perfettamente d'accordo. Συμφωνούμε απόλυτα. Ας ακούσουμε την Επίτροπο και μετά κάνουμε τη συνεδρίαση μας. Okay. Is, is it acceptable, Uh, I'm sure it is acceptable, although I won't be able to attend, whereas I can attend now. But what I will do is uh, write in... Κοιτάξτε, θα γράψω ένα email στους συντονιστές μου και σε εσά και στον κύριο Σόλτε και θα πω ποιες είναι απόψεις μου για τα θέματα που αντιμετωπίζουμε και ότι κάνουμε προσπάθεια να παρίσταμε η συνεδρία των συντονιστών να ληφθεί υπόψη. Εγώ της αλλαγής όμως δεν μπορώ να παραστώ.